Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Εγώ θα προεδρεύσω σήμερα το απόγευμα στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και συνεχίζουμε τα επόμενα σημεία. Μια ενημέρωση από τους διερμηνείς. Βρισκόμαστε στην 36η μέρα των διαμαρτυριών μας ε, μετά την μονομερή επιβολή από τη Διοίκηση Εργασιακών Συνδικών και τους διερμηνείς. Ε, με τα λύπη σας ε, ενημερώνουμε ότι η συνεδρίαση, ε, η διερμηνία θα διακοπεί κατά την προβλεπόμενη ώρα λήξη της συνεδρίασης. Ευχαριστούμε για την κατανόηση. We thank you again, interpreters. Ευχαριστούμε και πάλι τους διερμηνείς, λέει ο και σας ευχόμαστε καλή τύχη στις διεκδικήσεις σας. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Και εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη συνεδρίαση α, όπως προβλέπετε σε 3,5 ώρες και να ολοκληρώσουμε κατά την προβλεπόμενη ώρα λήξης. Περνάμε λοιπόν στη ημερήσια διάταξη. Έχουμε καταρχήν την εφαρμοστική απόφαση για την ε, υπαγωγή ε, στο κατάλογο και νέων ψυχοτρόπων ε, ουσιών. Δεν πρόκειται να σας αναφέρω με λεπτομέρειες όλες τις ψυχοτρόπες ουσίες που περιλαμβάνονται στο οικείο τμήμα της ημερήσιας διάταξης. Η ουσία όμως είναι η η διαβούλευση σε ό,τι αφορά το σχέδιο εφαρμοστικής απόφασης για τη συμπερίληψη νέων ψυχοτρόπων ουσιών. Η συγκητής για το σημείο αυτό είναι ο συνάδελφός μας, ο κύριος Σκρίπεκ. Θα μας κάνει εκείνο την παρουσίαση και μετά θα υπάρξει χρόνος και για τους και οδησηγητές αν θέλουν να υποβάλουν σχόλια. Κύριε Συγκητά, έχετε το λόγο. Κύριε Σκρίπεκ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σίγουρα. η ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών και η προστασία τους είναι βασική μέρημνα των κοινοτικών θεσμικών οργάνων και των κοινοτικών οργανισμών. Θέλουμε να προστατεύσουμε τους πολίτες μας από εσωτερικές και εξωτερικές απειλές. Βέβαια, είναι συγκλονιστικό να χάνουν τη ζωή τους συμπολίτε μας από ε, κάποια ναρκωτικά που μπορούν να τα παραγγείλουν και να τα παραλάβουν ε, στο στο, στη ταχυδρομική του θηρία. Ε, και μάλιστα μπορούν ακόμη και παιδιά να παραγγείλουν τέτοιε ναρκωτικέ ουσίε, ερήμην των γονιών του. Και μάλιστα οι εγκληματικέ συμμορίε ε, και οι παρασκευαστέ τέτοιων ουσιών στέλνουν τέτοια ναρκωτικά στα ε, σπίτια των Ευρωπαίων πολιτών. Ε, βέβαια, η Ευρωπαϊκή ε, νομοθεσία προβλέπει κάποια συνεργασία σε ό,τι αφορά τον εντοπισμό αυτών των ψυχοτρόπων ουσιών που είναι ουσιαστικά νόμιμες ε, ε, παρεστησιογόνες ουσίες και το 2018 είχαμε ένα κατάλογο που εμπλουτίζεται συνεχώς μετά από στοιχεία των κρατών μελών που μεταδίδονται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεχώς έχουμε την προσθήκη νέων ψυχοτρόπων ουσιών και ναρκωτικών. Το πρόγραμμα της φεντανίλης είναι γνωστό και έχει ε, προκαλέσει το θάνατο πολλών Ευρωπαίων πολιτών και αυτά τα δύο ψυχοτρόπα φάρμακα έχουν σκοτώσει πάνω από 65 Ευρωπαίους πολίτες από τον Ιούνιο του 2017 μόνο, μόνο την τελευταία διατηρία και κυρίως στη Σουηδία. Εκεί είχαμε ε, εκτενή χρήση αυτού του ναρκωτικού και μάλιστα έχουν ελκυστικά ονόματα όπως η θετική ηρωίνη, η MPF, η μεθοξύλ. Είναι πολύ πιασάρικα ονόματα και πολύ συχνά οι χρήστες δεν γνωρίζουν τη δραστικότητα αυτών των ναρκωτικών και μερικά τέτοια ναρκωτικά είναι, έχουν 50 φορές ισχυρότερη δράση από τα οπιούχα και ε, οδηγούν σε αναπνευστικά προβλήματα και μπορεί ο χρήστης σε δύο λεπτά ε, η σχεδόν ακαρία να πάθει ασφυξία και να πεθάνει. Και με το καταπληκτικό έργο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας μπορούμε να κρατούμε μείωτη την προσοχή μας και την εγρήγορσή μας ε, κατά των ναρκωτικών θανατηφόρων αυτών ναρκωτικών που φτάνουν ε, στα γραμματοκιβώτια μας και μερικά έχουν ε, ε, την ιατρική χρήση, αλλά χρησιμοποιούνται και από τους ανθρώπους και είναι εθιστικά. Ευχαριστώ που συμβάλαμε στην ποινικοποίηση της χρήσης και αυτών των δύο ουσιών για να αποτρέψουμε άλλους θανάτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω αυτό το μήνα να εγκριθεί στην Επιτροπή μας και να περάσει στην Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου και προσβλέπω σε ένα αίσιο πέρας όλης αυτής της διαδικασίας. Χωρίς μικρόφωνο δυστυχώς ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε κύριε Σιγητά για την παρουσίαση που μας κάνατε. Έχουμε λίγο χρόνο τώρα για τους και ηγητές που μπορούν να λάβουν το λόγο και να υποβάλουν τα σχόλιά τους, αν το επιθυμούν φυσικά. Πρώτα, ο σκιώδης ηγητής του ΕΛΚ, που είναι ο κύριος Μπρίς Οχτεφέ, ο οποίος όμως απουσιάζει τον αναπληρώνει κανένας. Όχι. Η κυρία Άννα Χέντ όμως, η σκιώδης ηγετήρα των Σοσιαλιστών, είναι παρούσα και έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ απόλυτα ε, με τον εισηγητή. Όπως μας είπε, αυτά τα δύο ναρκωτικά είναι πολύ επικίνδυνα. Οι δύο αυτές ψυχοτρόπες ουσίες είναι εξαιρετικά τοξικές. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω αυτά που μας είπε πολύ σωστά ο εισηγητής. Επαναλαμβάνω ότι αυτές οι δύο ψυχοτρόπες ουσίες είναι υπεύθυνε για μια σειρά θανάτων Ευρωπαίων πολιτών. ιδίως η πρώτη ουσία, φεντινόλη, που έχει συνδεθεί με 77 θανάτους, το σάκλο προπανό φεντινόλ. Και μάλιστα χρησιμοποιείται μερικές φορές σπρέι που εισπνέουν οι χρήστες. Ιδιαίτερα σε τέτοια περίπτωση στη χρήση σπρέι ο κίνδυνος ε, υπερβολικής δόσης είναι πολύ μεγάλος και μάλιστα είχαμε την περίπτωση ενό παιδιού που χρησιμοποίησε το σπρέι του γονιού του και δυστυχώ πέθανε από ασφυξία. Και η δεύτερη ουσία είναι υπεύθυνη για 13 θανάτους. Όπως είπε ο εισηγητής, ελπίζω το Σεπτέμβριο να εγκριθεί αυτή η έκθεση και στην Ολομέλεια για να ξεκινήσουμε επιτέλους να καταπολεμούμε αυτά τα επικίνδυνα ναρκωτικά. Μάλιστα. Άλλος κανεί παρακαλώ θέλει το λόγο. Δεν βλέπω ούτε την κυρία Παγασάουρ Τουντούα από τους Φιλελεύθερους, ούτε την κυρία Άντερσον από την ΚΟΕ. Άλλος κανείς? Όχι, οπότε ολοκληρώνουμε. Μην ξεχνάτε την διορία για την υποβολή τροπολογιών που λήγει στις 16 Ιουλίου 4 το απόγευμα. Εντάξει. Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλει το λόγο για σχολιασμό. Οκ, εντάξει. Περνάμε στο επόμενο σημείο, το υπαριθμό 19 και μάλιστα εγκαίρω. Ε, αποστολή της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών στην Κύπρο, 3 με 5 Απριλίου, τρέχοντος έτους. Παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης της αποστολής επειδή εγώ ήμουν επικεφαλής αντιπροσωπείας, εγώ θα σε ενημερώσω για αυτή την αποστολή. Και μάλιστα έχω προβλεφθεί ένα τέταρτο για τη σχετική συζήτηση. Απλώς ήθελα να σας παρουσιάσω κάποιες απόψεις για τις εξελίξεις αυτής της επίσκεψής μας στην Κύπρο στις αρχές Απρίλιο. Θα θυμάστε ότι στόχος της αποστολής ήταν η συγκέντρωση πληροφοριών για τη, τελευταία ε, γεγονότα και τα έργα της Επιτροπής Αγνωμένων στην Κύπρο με βάση το ενεργητικό φορέα που συστήθηκε υπό την αιγύδα των Ηνωμένων Εθνών για να ε, διαλευκανθούν οι περιπτώσεις αγνωμένων κατά την περίπτωση ε, ε, της ε, Διαρευνητικής Επιτροπής για τους Αγνωμένους που έγινε κατά τη στιγμή της διχοτόμησης του νησιού. Και μάλιστα η αντιπροσωπή αυτή ήθελε να ε, κάνει μια αξιολόγηση των, ε, των εργασιών σε ό,τι αφορά τον, ε, την ταυτοποίηση και να προβλέψει το μέλλον και το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για την ανάκτηση όλων τουλάχιστον της πλειοψηφίας των αγνοωμένων καθώς και το βαθμό συνεργασίας μεταξύ των ενεχομένων αρχών. Και τη χρηματοδότηση του σχεδίου αυτής της Διερευνητικής Επιτροπής που επιβαίνει κυρίως σε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια είναι τώρα αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά του σχέδιου έκθεσης ε, των πεπραγμένων της Απόστολης. Σας έχω μοιράσει το σχέδιο. Καταρχήν το υπόβαθρο. Είχαμε ένα ψήφισμα τον Ιούνιο, 18 Ιουνίου του 2008 σχετικά πρόσφατα. Εκεί η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών ζήτησε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσει μια συνέχεια στο θέμα των αγνοωμένων στην Κύπρο και να κάνει τα απαραίτητα διαβήματα για να πείσει τις εμπλεκόμενες πλευρές να συμβάλλουν ε, ενεργά και δραστήρια στην, ε, προκειμένου, να, στις προσπάθειες για τη διερεύνηση της τύχης κάθε αγνοωμένου στη δήλωση τη 9 η Ιουλίου 2011 σχετικά με, την εργασία, με τις εργασίες της αποστολής για τους αγνωμένους και το ψήφισμά μας στις 12 Φεβρουαρίου του 2015, στην τρέχουσα θητεία δηλαδή, ε, σχετικά με τους ομαδικούς τάφους αγνοωμένων της Άσιας στο χωριό Ορνήθη, στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνισε την ανάγκη να προχωρήσουν γρήγορα οι εργασίες για την ενέβραση και την ταυτοποίηση των αγνοωμένων. Μάλιστα το 2016 ο υποφαινόμενος ορίστηκε μόνιμος εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το ζήτημα των αγνοωμένων στην Κύπρο. Γι' αυτό και συστήσαμε αυτή την αποστολή προκειμένου να συλλέξουμε πληροφορίες για τις τελευταίες εξελίξεις στο έργο της Διερευνητικής Επιτροπής και το επίπεδο συνεργασίας των ε, αρμοδίων αρχών. Εμείς ε, θεωρούμε ότι υλοποιήσαμε πλήρως και το πρόγραμμα εργασιών μας και το στόχο της ε, αποστολής. Από τις 3 μέχρι τις 4 Απριλίου 9 με 8 9 με 10 το βράδυ μερικές φορές, δηλαδή εξαντλήσαμε πραγματικά το ημερήσιο πρόγραμμα. Δουλεύαμε συνεχώς. Ξεκινήσαμε με κάποιες συνεδριάσεις, συναντήσεις με ε, την εκπρόσωπο, την ειδική αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και αρχηγό της Ενευτικής Δύναμης του ΟΗΕ στην Κύπρο, την κυρία Ελίζα Σπέχαρ. Επίσης, συναντηθήκαμε με τον κύριο Πολ Αγρή Αρνή, που συνόδευε την κυρία Σπέχαρ και είναι μέλος Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους στην Κύπρο, έχει οριστεί από τον ΟΗΕ. Και η κυρία Σπέχαρ και ο κύριος Αρνή μα έκανε μια συνοπτική παρουσίαση για την εντολή και τα τρέχοντα καθήκοντα αυτή τη ειρηνευτική δύναμη των ΗΕ στην Κύπρο για να αποφευθούν περαιτέρω συγκρούσεις μεταξύ τη ελληνοκυπριακής και τη τουρκοκυπριακή κοινότητα στο νησί. Μα ενημέρωσαν για τις ε, ε, αρχές της ε, διένεξης, τα, τις εχθροπραξίες του 1974, τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και την de facto κατάπαυση του πυρός του 1974 και επίσης μας παρουσίασαν διεξοδικά την εντολή που μας ενδιαφέρει και επίσης μας έδωσαν κάποια στοιχεία για τον προϋπολογισμό αυτής της Διερευνητική Επιτροπής που είναι αυτή τη στιγμή 3 εκατομμύρια ευρώ από τα οποία 2,6 εκατομμύρια προέρχονται απευθείας από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Επίσης απάντησαν στις ερωτήσεις των μελών σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στις ε, στρατητικές ζώνες, τις περιορισμένες ζώνες και μας εξήγησαν ότι αυτό δεν είναι πια πρόβλημα. Σε 51 περιπτώσεις έχει ε, εγκριθεί η πρόσβαση στα αρχεία και η σχετική βέβαια ε, στις συγκεκριμένες ζώνες. Ό,τι αφορά την πρόσβαση στα αρχεία όμως, η Διερευνητική Επιτροπή περιμένει περισσότερες άδειε από τις αρμόδιες τουρκικές αρχές. Επίσης, συναντήσαμε κάποια μέλη της ε, Διερευνητικής Επιτροπής για, τις, για τους αγνοωμένους. Η κυρία Κιουτσούκ, που είναι το τουρκοκύπριο μέλο, συναντηθήκαμε τον κύριο Νέστορα, Νέστορα που είναι ο Ελληνοκύπριο μέλος τη ε, ε, Επιτροπής και ήταν παρόν και ο κύριο Ανρί Αρνή που είναι το μέλος του ΟΗΕ στην Επιτροπή αυτή. Ε, συζητήσαμε τις ε, εργασίε εκταφιασμού, ταυτοποίηση και επιστροφής των σωρών των νεκρών Και επίσης κάποια κοινοτικά σχέδια γίνονται και στις δύο πλευρές, και στην τουρκοκυπριακή και στην ελληνοκυπριακή πλευρά και έχουν εκδηλώσει και οι δύο κοινότητε την εμπιστοσύνη του για τι ανθρωπιστικέ πτυχέ του έργου τη Διερευνητική Αποστολή. Τη Διερευνητική Επιτροπή, κυρία Κουτσούκα ενημέρωσε του βουλευτέ ότι έω τι 31 Μαρτίου 2018 είχαν πραγματοποιηθεί 1218 εκταφέ και ταυτοποιηθεί τα λείψανα 868 ατόμων. Ο κύριος Νέστορας επισήμανε τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζει το έργο της ΔΕΑ και τόνισε ότι ο χρόνος είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Όπως ξέρουμε, οι οικογένειες ακόμη θρυνούν. και μας υπενθυμίζουν ότι ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. Επίσης, ο κύριος Αρνή υπενθύμισε τη σημασία που έχει η αποκατάσταση εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο κοινότητων και ανέφερε τη σημασία που έχει η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επίπεδο προϋπολογισμού. Η κυρία Κιουτσούκ διευκρίνησε ότι δεν υπάρχει χρονικό όριο για το έργο. Τα τρία μέλη υπογράμμισαν ότι η ιδέα δεσμεύεται από την εντολή της, μεταξύ άλλων από τον κατάλογο των αγνοωμένων που καθορίστηκε σε πολιτικό επίπεδο. Και το γεγονός επίσης ότι η ιδέα δεν είναι αρμόδια να εξακριβώσει την αιτία θανάτου των αγνοωμένων. Μάλιστα, ε, επισκεφθήκαμε και ένα ιατροδικαστικό εργαστήριο ή ανθρωπολογικό εργαστήριο της ΔΕΑ. Συζητήσαμε με εμπειρογνώμονες και επιστήμονες και επίσης ε, πήγαμε και στην ε, Βουλή των Αντιπροσώπων και συναντήσαμε τον πρόεδρο τον κύριο Σιλούρη ε, και την πρόεδρο της κυρία Κούτρα Κούκουμα ε, που είναι η πρόεδρο τη Μόνιμη Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων Εγκλωβισμένων Αγνοωμένων Παθόντων και μέλη τη Επιτροπή και συζητήσαμε για την πολιτική διάσταση τη ε, επιχείρηση και τις προσδοκίες που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλουμε να υλοποιηθούν. Επίσης, συναντηθήκαμε με τον κύριο Φώτη Φωτίου, που είναι ο ειδικό Επίτροπος για τα ανθρωπιστικά θέματα. Και συζητήσαμε για το έργο της Επιτροπής αυτής και μάλιστα κρίνουμε αυτό το θέμα στο πιο τραγικό στην κυπριακή ιστορία. Και έχουν πέρασει 44 χρόνια και ακόμη πολλές οικογένειες περιμένουν την ολοκλήρωση ε, των εργασιών. Ο κύριος Φωτίου επισήμανε την ανάγκη να αποκτηθεί πρόσβαση στα αρχεία του τουρκικού στρατού προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά τον εντοπισμό των λιψάνων και κάλεσε τους βουλευτές να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους να μεταφέρουν τα μηνύματα στις τουρκικές αρχές. Επίση, ο Επίτροπο Προεδρία αναφέρθηκε στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου τη 10η Μαου 2001 και στη μη συμμόρφωση τη Τουρκία, καθώ και στην κατάσταση των εγκλωβισμένων στη Χερσόνησο τη Καρπασία. Επίσης, συναντηθήκαμε με συγγενεί αγνοωμένων. και οι δύο πλευρέ και η τουρκοκυπριακή και η ελληνοκυπριακή κοινότητα ήταν πολύ συγκινημένε ε, Αποτίσαμε φόρο τιμή ε, και εκφράσαμε το σεβασμό μας προς τους ισχυρισμού τις ευαισθησίε τους, ε, τις προσδοκίε τους και την ανάγκη να κρατήσουμε αυτό το θέμα στο ανθρωπιστικό επίπεδο και να αποφύγουμε μια πολιτικοποίηση του ζητήματος. Όλοι υπογράμμισαν την οδύνη των οικογενειών, άσχετα από την κοινότητα στην οποία ανήκουν. Και επίσης βίωσαν πολλές εμπειρίες ό,τι αφορά την παρακολούθηση του έργου του εκταφιασμού και της ταυτοποίησης των λειψάνων και εξέφρασαν την προσδοκία να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία. Επίσης, ε, συναντηθήκαμε με την Δικοινοτική Ένωση Συγγενών με τον τίτλο «Μαζί μπορούμε» που εκπροσωπήθηκε από τον κύριο Χρήστο Ευθυμίου, την κυρία Σευγγύλ Ουλουντάχ και την κυρία Χριστίνα Παύλου Σολομή Πατσιά. Εκατακλείδη, η αντιπροσωπεία αναγνωρίζει ότι το ζήτημα των αγνοουμένων σε μετασυγκρουσιακές καταστάσεις αποτελεί πολύ σημαντικό στοιχείο της διαδικασίας πολιτικής, νομικής και κοινωνικής μετάβασης από την οποία πολλές ευρωπαϊκές χώρες ε, έπρεπε να διέλθουν και εξακολουθούν να διέρχονται. Οι συγγενείς των αγνοωμένων έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται σχετικά με την τύχη των οικείων τους. Οι οικογένειε των αγνοωμένων και των θυμάτων βίων εξαφανίσεων και οι ανάγκες αυτών των οικογενειών πρέπει να τεθούν στο επίκεντρο όλων των δράσεων που αφορούν τα θέματα αυτά. προκειμένου έτσι να προαχθεί η συμφιλίωση εντός των κοινωνιών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρακολουθεί ενεργά την κατάσταση στην Κύπρο και μετά το πέρας των συναντήσεων θα θέλαμε να πούμε ότι στηρίζουμε το έργο της ΔΕΑ αναγνωρίζουμε τον ρόλο μετά τη σύγκρουση, μετά τη σύραξη και που διαδραματίζει για την πρόθεση της αλήθειας, της μνήμης και της συμφιλίωσης στην Κύπρο, καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει να διαθέτει επαρκής και το τονίζω, επαρκής πόρους στην ΔΕΑ, στην Διερευνητική Επιτροπή Αγνωμένων, ώστε να είναι σε θέση να διεκπαιρεώσει τη σημαντική αποστολή τη. Και καλούμε τις κυβερνήσεις της Τουρκίας και της Κύπρου να συνεχίσουν να στηρίζουν το έργο της ΔΕΑ, να διπλασιάσουν τι προσπάθειες του για την ανέβρεση των ατόμων που εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στους καταλόγους ευνοωμένων και να διασφαλίσουν την ελεύθερη διάθεση στη ιδέα όλων των πληροφοριών που θα μπορούσαν να διευκολύνουν την αποστολή της. Καλούμε την τουρκική και την ελληνική κυβέρνηση, αλλά και τα Ηνωμένα Έθνη να παράσχουν πρόσβαση στη ΔΕΑ σε πληροφορίε καταχωρισμένε στα αρχεία του. Η αντιπροσωπή επίση υπογραμμίζει επίση το δικαίωμα ενημέρωση σχετικά με την τύχη αγνωμένων συγγενών αυτό αποτελεί θεμελιώδη δικαίωμα των ε, ενδιαφερομένων οικογενειών και πρέπει να διασφαλιστεί. Επαναλαμβάνουμε επίσης και διατρανώνουμε το ανθρωπιστικό ζήτημα των αγνοωμένων στην Κύπρο, που είναι ένα αυτοτελέ ζήτημα και δεν θα πρέπει να επηρεαστεί από οποιαδήποτε άλλη πολιτική σκοπιμότητα, ούτε να συνδέεται με τη προσδοκία επανάληψη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Ε, σίγουρα το, προέχω, το ζήτημα προέχει είναι η επανασυφιλίωση και η επανένωση της νήσου, της Μεγαλονήσου. Και αυτή είναι και η δική μας ευχή, να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος. Αυτά, ε, συντομία, τα βασικά στοιχεία της έκθεσής μας και αν θέλει κανείς το λόγο, πολύ ευχαρίστως να τον ακούσουμε. Ο κύριος Μαυρίδης. Μάλιστα ο κύριος Μαυρίδη συμμετείχε σε αυτή την αντιπροσωπεία. Και ο κύριος Δεχόφσκι επίσης, που δεν μπορώ να προφέρω και το όνομά του. Ο κύριος Μαυρίδης όμως πρώτος σήκωσε το χέρι και προηγείται να μιλήσει. Thank you, Um, I my mother tongue. Η επίσκεψη αυτής της αποστολής ε, ε, και οι επαφές της είναι ένα πολύ σοβαρό βήμα σε ένα απόλυτα ανθρωπιστικό θέμα. Ευχαριστίες ιδιαίτερες σε όλη την αποστολή που επισκέφθηκε την Κύπρο, αλλά ιδιαίτερες ευχαριστίες στο συνάδελφό μας, τον κύριο Αγγιλάρ, ο οποίος είναι ο ειδικό εισηγητής για αυτό το θέμα. Παρεμπιπτόντως, κατανοώ πλήρως την προσπάθεια ισορροπίας αφαιρώντας όσο γίνεται τις πολιτικές σκοπιμότητες, οι οποίες όμως αναπόφευκτα υπάρχουν ενώ όσο συνεχίζεται η κατοχή της Κύπρου. Γι' αυτό θα περιοριστώ σε τρία γενικά σχόλια, χωρίς να μπω στην πολιτική κατάσταση, παρόλο που έχω συγκεκριμένη άποψη για το ποιο είναι ο θήτης και ποιο είναι το θύμα. Το πρώτο μου σχόλιο είναι ότι δίνουμε μια μάχη ενάντια στον χρόνο. Γι' αυτό και ο ρόλος μας εδώ ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πέραν από την χρηματοδότηση, είναι πολιτικός. Να πιέσουμε τις διαδικασίες, γιατί δυστυχώς κάθε μέρα που περνά φεύγουν άνθρωποι που έχουν πληροφορίες και χάνουμε πάρα πολύ κρίσιμη ενημέρωση και πληροφόρηση για να εντοπίσουμε ένα ακόμα αγνοούμενο της τραγωδίας της Κύπρου. Το δεύτερο σχόλιο μου είναι ότι συμμερίζομαι πλήρως ότι η απονομή της δικαιοσύνης και η ανέβρεση της αλήθειας οδηγεί στη συμφιλίωση και στη λύτρωση. Όμως εδώ θα πρέπει να τονίσω δύο πράγματα. Ότι υπάρχουν παραδεχτά γεγονότα και από τις δύο πλευρές υπάρχει για το κράτος δικαίου. Τα παραδεχτά γεγονότα είναι ότι η Τουρκία έχει σκόπιμα μετακινήσει ωστά και το δεύτερο είναι ότι όντως υπάρχει απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου το οποίο καλεί την Τουρκία επιτέλους να συνεργαστεί πλήρως. Τελειώνω, κύριε Σέρμαν, ε, ε, με μία τελευταία φράση. Θεωρώ ότι αυτό που κάνουμε εδώ είναι πλήρως ανθρωπιστικό και γι' αυτό να αφήσουμε έξω οποιασδήποτε πολιτικές σκοπιμότητες. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ κύριε Μαυρίδη. Με συγχωρείτε που σας είπα ότι πρέπει να τελειώσετε, αλλά μόλις κατάλαβα ότι έχουμε άλλο ένα θέμα που πρέπει να σας απασχολήσει πριν αρχίσει η ακρόαση στις 3.30. Γι' αυτό θα παρακαλούσα τους υπόλοιπους συναδέλφου που σήκωσαν το χέρι να είναι σύντομοι. 1,5 λεπτό παρακαλώ, 2 λεπτά το πολύ, για να μην καθυστερήσουμε. για να διατηρήσουμε τα δικαιώματα των διερμηνέων που όμως μας ε, ανήγγυλαν θα σταματήσουν στις 6.30 ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ για τη θαυμάσια προφορά του ονόματός μου. Θα ήθελα να πω τα εξή. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ για την τόσο ισορροπημένη παρουσίαση που μας κάνατε. Καλύψατε όλα τα θέματα που μας απασχόλησαν. Αυτή η αποστολή ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και ελπίζω ότι με την αποστολή μας ε, θα συμβάλλουμε στην ειρήνη μεταξύ του βορείου και του νοτίου τμήματος της Κύπρου. Προτιμώ να μην, να μην χρησιμοποιήσω τις λέξεις ε, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι. Πρέπει οπωσδήποτε ε, να αποφευχθεί η απάλληψη από μεριά της Τουρκίας των ε, συνεπειών αυτής της, ε, αυτού του μακελιού. Πρέπει οπωσδήποτε να φτάσουμε σε μια συμφωνία που να γίνει αποδεκτή και από τις δύο πλευρές. Αυτό είναι κλειδί για να επιληθεί το πρόβλημα και ελπίζω κάποια μέρα να μπορέσουμε να επισκεφτούμε την Κύπρο και τα τείχη μεταξύ του βόρειου και του νότιου τμήματος να έχουν καταρριφθεί και να γιορτάσουμε την ενοποίηση της Κύπρου. Ο, ο κύριος Άνταμοφ, που επίσης ήταν μέλος της αντιπροσωπείας μας, παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ. Και εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Νομίζω ότι επιτύχαμε το στόχο της επίσκεψης αυτής 100% και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους αδέλφους που συμμετείχαν και να ευχαριστήσω και εσάς κύριε Πρόεδρε γιατί ως επικεφαλής παίξατε πολύ σωστά το ρόλο σας. Ε, Ήταν μια δύσκολη αποστολή με έντονη συναισθηματική φόρτιση γιατί εντοπίσαμε μια ανθρώπινη τραγωδία που ε, κρατάει εδώ και 44 χρόνια. Αυτή η τραγωδία, αυτή η δυστυχία δεν πρέπει να πολιτικοποιηθεί. Πρέπει να εξετάσουμε αυτά που σβαίνουν εκεί ως άνθρωποι, απλώς ως άνθρωποι. Σας ευχαριστώ που η έκθεσή σας ήταν ε, αντικειμενική. Και ο κύριος Χριστοφόρου ήταν εκεί θα ήθελα από καρδιά να σα ευχαριστήσω τόσο εγώ όσο και ο Κυπριακό λαό για την πραγματικά σημαντική και υπεύθυνη αποστολή που πραγματοποιήσατε εσεί ω πρόεδρο αλλά και τα μέλη τη αποστολή. Γι' αυτόν κύριε Αγγιλάρ, πραγματικά σα ευχαριστούμε και θεωρούμε ότι ήταν μια σημαντική θετική συμβολή σε αυτόν το καθαρά ανθρωπιστικό θέμα. Το θέμα των αγνωμένων δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ήταν το αποκορύφωμα μια τραγωδία που συνετελέστηκε στην Κύπρο εξαιτία τη τουρκική εισβολή και τη κατοχή του 1974. Είναι απότοκο αυτών των εγκλημάτων που διαπράχθησαν μέσα από την παράνομη εισβολή και κατοχή, η οποία κρατάει εδώ και 44 χρόνια. Και ενώ είναι καθαρά ανθρωπιστικό αυτό το ζήτημα, είναι το δικαίωμα των οικογενειών να μάθουν για την τύχη των αγνωμένων του, η Τουρκία, συνεχίζοντα αυτήν την απαράδεκτη στάση και συμπεριφορά, κρατεί τα αρχεία του τουρκικού στρατού κλειστά και δεν τα ανοίγει για να πληροφορηθούμε για την τύχη των αγνωμένων, κρατά κλειστέ στρατιωτικέ περιοχέ και δεν επιτρέπει την πρόσβαση για να μπορέσουν να βρεθούν πληροφορίε για του αγνωμένου και μετακινεί ακόμα και ω τάγνωμένο. Πιστεύω ότι αυτή η στάση και συμπεριφορά πρέπει να στυλιτευτεί και να σταλεί το ισχυρό μήνυμα στην Τουρκία ότι τουλάχιστον για αυτό το καθαρά ανθρωπιστικό ζήτημα οφείλει να επιδείξει επιτέλου ευαισθησία μετά από 44 χρόνια. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να επιταχυνθούν οι ρυθμοί για του αγνοούμενου, για την ανέβρεση των αγνοούμενων μα. Και να καταστεί δυνατόν χρειάζεται περαιτέρω οικονομική ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι και η μόνη η οποία συνεισφέρει σε τόσο ψηλά ποσά. Η δική σα συμβολή και προ αυτήν την κατεύθυνση είναι ιδιαίτερα σημαντική για να υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση αυτού του ζητήματο και θα ήταν μια σημαντική ανθρωπιστική επιτυχία και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για όλου εσά, εάν πραγματικά κατορθώσουμε να αλλάξουμε αυτά τα δεδομένα και το θέμα των αγνωμένων τη Κύπρου να μπει στην πρώτη γραμμή και να υπάρξει πραγματικά αποτέλεσμα όσον αφορά την ανέβρεση των αγνωμένων μα και την πληροφόρηση, το δικαίωμα στην πληροφόρηση των οικογενειών, είτε είναι Τουρκοκύπροι είτε είναι Ελληνοκύπροι. Για μα αυτό το θέμα δεν διαχωρίζει του ανθρώπου. Εμεί το θεωρούμε ένα θέμα ανθρωπιστικό. Εμεί ω ελληνοκυπριακή πλευρά κάναμε τα πάντα προ αυτή την κατεύθυνση. Ο πρόεδρο Κυπριακή Δημοκρατία αγωνίζεται με όλε τι δυνάμει Απλώ αναμένουμε και τη συμβολή του υπέτειου για ό,τι συμβαίνει εδώ και 44 χρόνια στην Κύπρο μα τη Τουρκία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι. Και εσεί θέλετε παρακαλώ. Παρακαλώ. Πώ λέγεστε. Ο κύριο Χρυσόγονο. Ο κύριο Χρυσόγονο. Παρακαλώ. Η τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, υπήρξε ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, το οποίο δυστυχώς συνεχίζεται έως σήμερα. Συνεχίζεται έως σήμερα όχι μόνο με την κατοχή και τον επικισμό του βόρειου τμήματος του νησιού, αλλά ακόμη και με ενέργειες ή παραλήψεις, οι οποίες αντιβαίνουν σε στοιχειώδεις κανόνες όχι μόνο του δικαίου, αλλά θα έλεγα και κάθε έννοια ανθρωπισμού, όπως είναι η άρνηση της Τουρκίας να συμβάλλει ώστε να εξευρεθούν έστω τα ίχνη των αγνοουμένων, οι οποίοι στην πραγματικότητα όλοι ξέρουμε ότι εκτελέστηκαν με τον πιο βάρβαρο και απάνθρωπο τρόπο από τα τουρκικά στρατεύματα ή τους τουρκοκύπριους παραστρατιωτικούς. Ε, συνεπώς, θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να στυλιτεύσει με τον πιο έντονο τρόπο τη συμπεριφορά αυτή της Τουρκίας, διότι η συμφιλίωση μεταξύ των λαών δεν μπορεί να στηρίζεται στη λύθη, αλλά πρέπει να στηρίζεται στην ιστορική αλήθεια. Και μόνο αυτή αποτελεί το ισχυρό βάθρο στο οποίο μπορούμε πραγματικά να συμφιλειωθούμε. Okay, points taken. Ωραία, τα σημειώνουμε. Και εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω αγαπητοί συνάδελφοι ως μόνιμος συζητητής σας και πρόεδρος της αντιπροσωπείας για τη συμμετοχή σας, τη συμβολή σας, την καλή σας θέληση, ε, τον τονισμό της ε, ανθρωπιστικής διάστασης αυτής της προσπάθειας, τη συμπαράσταση της οικογένειας και τον, τονισμό του δικαιώματός τους να λάβουν τα οστά των ε, αγνωμένων και ε, καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει την χρηματοδότηση ούτως ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια. Επίσης, Σωστό είναι και αυτό που αναφέρθηκε. ότι η Επιτροπή αυτή ζητάει εδώ και πολύ καιρό να μπορέσει να μπει στις ε, στρατιωτικές ζώνες περιορισμένης πρόσβασης. Στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Υπόθηκε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος και ότι αρκετά, ε, αρκετά οστά έχουν εκταφεί και έχουν ταυτοποιηθεί και είμαστε σε φάση ε, ταυτοποίησης και άλλων. Άρα όλο και περισσότερες οικογένειες θα ενημερωθούν. Και αυτό είναι ενθαρρυντικό. Τέλος. Ελπίζω ή μάλλον θα ήλπιζα να έχει ακολουθηθεί ένα παρόμοιο παράδειγμα σε άλλες περιπτώσεις ε, σειράξεων στο εσωτερικό της Ένωσης όπου έχουν υπάρξει θύματα και αγνοούμενοι θα επιθυμούσα αυτό λοιπόν το παράδειγμα να δημιουργήσει θετικό κλίμα για να βρούμε τα ωστά πολλών θυμάτων ε, συγκριούσεων ακόμη και στην ειδική μου χώρα, την Ισπανία. Το είπα επανειλημμένα όταν ήμασταν στην Κύπρο. Είχαμε ένα τρομερά αιματηρό εμφύλιο πόλεμο στη δεκαετία του 30 του παρελθόντος αιώνος. Και οι αγνώμενοι δεν είναι 3.000, είναι εκατοντάδες χιλιάδες. Εκατοντάδες χιλιάδες. Αλλά δεν υπήρχε καμία παρόμοια στάση. Όπως αυτή που διαπιστώσαμε στην Κύπρο, όπου οι κοινότητες ανταποκρίθηκαν στα αιτήματα των οικογενειών για να επιληθεί το θέμα και για να αντιμετωπιστούν δίκαια οι οικογένειες από τις αρχές με την πλήρη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ε, χρηματοδότηση της Ένωσης που εξυπηρετεί αυτό το σκοπό που επιμένω είναι ανθρωπιστικός βεβαίως υπάρχει πολιτική διάσταση πάντα υπάρχει και ελπίζουμε να επαναληφθούν οι συνομιλίες μετά τις καλοκαιρινές διακοπές Αυτή είναι μια άλλη πλευρά για να προωθηθεί η επίλυση του θέματος. Αλλά εμείς απλώς συνοδεύουμε την εργασία της ΔΕΑ και νομίζω ότι παίξαμε αυτό το ρόλο και το παίξαμε όσο καλύτερα μπορούσαμε. Οπότε να περάσουμε στο επόμενο θέμα της μέρης της διάταξης. που είναι προϋπολογισμός, να συζητήσουμε δηλαδή την έκθεση για το Γενικό Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, όλα τα τμήματα. που θα μας την κάνει ο ε, εισηγητής ο κύριο Χρυσόγονο και μετά θα ακούσουμε τις κοιόδες εισηγητής. Έχετε το λόγο κύριε Χρυσόγονο. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο σε σχέση με την εξέλιξη του ευρωπαϊκού εγχειρήματο. Ε, οι αυξανόμενε μεταναστευτικέ πιέσει στη Μεσόγειο, σε συνδυασμό με την μείωση τη προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, είναι σημαντικέ προκλήσει για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τα κράτη-μέλη. Οι προκλήσει αυτέ ε, πρέπει να έχουν ω αποτέλεσμα λύσει από συνεργασία για να μπορέσουμε να προασπιστούμε τι βασικέ βασικέ αξίε και αρχέ Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και να υπάρχει αλληλεγγύη και υποστήριξη για την δικαιοσύνη, την συνέχεια και τη συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια ομαλά λειτουργούσα Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαιοσύνη και Ελευθερία είναι απαραίτητη προπόθεση για την καταπολέμηση τη εγκληματικότητα και τη διαφθορά και για την εξασφάλιση τη ε, σωστή εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων εντό Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς, ε, το επίπεδο των οικονομικών πόρων που παρέχεται από τον ενωσιακό προϋπολογισμό για το ε, άμεσο μέλλον θα ε, χρηματοδοτηθεί πλήρως. Θα υπάρξει μία, ένας μόνιμος βιώσιμος μηχανισμός για τη χρηματοδότηση των δράσεων για την ασφάλεια και για τη μετανάστευση. Η αύξηση περίπου 7% ε, των πιστώσεων υποχρεώσεων για τον ε, τίτλο 3 ασφάλεια και ηθαγένεια για το 2019 είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση δηλαδή από 3,5 δις ευρώ το 2018 σε 3,73 δις ευρώ το 2019. Το ίδιο ισχύει και για την αύξηση των πιστώσεων υποχρεώσεων ε, από 11,2 δις σε 11,5 δις το 2019, όπως επίσης και πιστώσεις, ε, στην αύξηση των πιστώσεων πληρωμών ε, για το... Ε, τομέα 3. Ε, υπάρχει ένα περιθώριο επίσης υπό τον τίτλο 4 και υπάρχει και διάθεση πάνω από ενός δις ε, ευρώ ε, για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την ανθρωπιστική μας βοήθεια και το, μέσο ευρωπαϊκής, το Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας ε, που επίσης βεβαίως είναι θετικό. Η σημαντική αύξηση ε, του, των, ε, ταμείων για, την, για το άσυλο και τη μετανάστευση και των σχετικών πιστώσεων ε, πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ για να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί ο νέος κανονισμός Δουβλίνου και το 1,75 δις ευρώ που ζητάει η Ελλάδα για την, το, τον κατεπήγοντα μηχανισμό από τον Ιανουάριο του 2019 επίσης πρέπει να θεωρηθεί μια θετική εξέλιξη. Να σημειώσω επίσης ότι 1,44 δι ευρώ θα χρηματοδοτηθούν από τον Ενωσιακό Προϋπολογισμό για τη χρηματοδότηση τη της διευκόλυνσης ε, για τους πρόσφυγες στην Τουρκία και 5,6 ε, δι ευρώ για την 560 ε, εκατομμύρια ευρώ για την κρίση στη Συρία. Όσον αφορά τώρα την, το μέσο για την ε, δικαστική, την εξαρτησία του δικαστικού τομέα στην Τουρκία. Ε, θα υπάρξει η έγκριση των χρηματοδοτικών ροών ε, κατόπιν παρακολούθησης της εξέλιξης. Όσον αφορά τώρα το μέσο το προενταξιακό, αύξηση, μείωση 253, 253 εκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με το αρχικό έγγραφο στρατηγικής, κάτι το οποίο επίσης ε, είναι ευπρόσδεκτο. Το γενικό επίπεδο υποστήριξης ε, για το ΕΑΖΟ ε, σε σχέση με τα αρχικά ποσά που είχε εξαγγείλει η Κομισιόν είναι επίσης ευπρόσδεκτο. Αύξηση 16% των διοικητικών δαπανών για να καλύψουμε τις νέες ευθύνες της γραμματείας για την προστασία των συνόρων όπως επίσης και για τους κανόνε κανόνες προστασίας δεδομένων και για την παρακολούθηση και τη συμμόρφωση με τους κανόνες προστασίας δεδομένων των ε, ε, υπηρεσιών που παλιά ήταν στον τρίτο πυλώνα. Επίσης, Πρέπει να πούμε ε, ότι δεν ισχύει το ίδιο για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την ε, διαχείριση των μεγάλης κλίμακας ε, πληροφορικών συστημάτων για τον τομέα της ασφάλειας, της ελευθερίας και της δικαιοσύνης, το eu δηλαδή. Ε, το 2019 θα είναι πάρα πολύ δύσκολο έτος για το Ιουλίσα, ε, δεδομένη σημαντικής αύξησης των καθηκόντων του και του προϋπολογισμού. Αναμένεται λοιπόν ότι το 2019 θα χρειαστεί ενίσχυση των πόρων του, το Λίσα για να μπορέσει να επιφέρει τα αποτελέσματα που χρειάζεται βάσει της τρέχουσας εντολής του. Ένας προϋπολογισμός 4,9 εκατομμυρίων ευρώ ε, για το την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ε, είναι επίσης ένα θετικό ε, ένα θετικό μέτρο. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε διασυνοριακά να αναλαμβάνει καθήκοντα χωρί να υπάρχουν προηγούμενε διαδικασίε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα παράνομα έσοδα ε, που, κάνουν, που έχουν οι κλιματικές δραστηριότητες, οι κλιματικές ε, οργανώσεις κάθε χρόνο με παράκαμψη των ευρωπαϊκών κανόνων. Θα υπάρξει πιο αποτελεσματική δίωξη και καλύτερη ανάκτηση των ποσών που αποτελούν αντικείμενο απάτη. Κρίμα είναι λοιπόν που η Eurojust είναι ο μόνος οργανισμός ε, ε, δικαιοσύνης ε, που αντιμετωπίζει περικοπές για το 2019 με αντιπαραγωγική μείωση των πιστώσεων υποχρεώσεων για το πρόγραμμα δικαιοσύνης κατά 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ε, Επίση, υπάρχουν και ανησυχίε γιατί τρέχουσα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χρηματοδότηση τη Eurojust ε, από το 2021 έως το 2027, στο νέο δηλαδή ΠΔΠ, ε, δεν θα είναι επαρκή γιατί θα υπάρξει περικοπή κατά 15% περίπου σε ετήσια βάση σε σχέση με το 2018. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν ε, πρέπει να τονιστεί ότι τέτοιου είδους μείωση δεν είναι βιώσιμη λόγω της επιχειρησιακής ανάπτυξης και των πολιτικών προτεραιοτήτων για την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ότι οι απειλές στην ασφάλεια έχουν διαφοροποιηθεί στην Ευρώπη και έχουν ενταθεί κατά τα τελευταία χρόνια. Ε, έχουν, φτάσει, έχουν εμφανιστεί με νέου είδους τρομοκρατικές επιθέσεις και οργανωμένη εγκληματικότητα όπως και ε, ε, με έγκλημα στον κυφέρνο χώρο. Ε, ο Γιώργος, συγγνώμη κυρία Χρυσόγωνε, πρέπει να σας υπενθυμίσω, λέει ο Πρόεδρος, ότι ε, έχουμε και ένα χρονοδιάγραμμα γιατί έχουμε και μία ακρόαση στις 3.30 και υπάρχουν και δύο ευρωβουλευτές που θέλουν να πάρουν το λόγο. Μήπως μπορείτε λοιπόν να ολοκληρώσετε. Να πω λοιπόν ε, απευθεία στα συμπεράσματά μου. Πρέπει λοιπόν να έχουμε στο μυαλό μα ότι η σωστή εφαρμογή του προπολογισμού, ειδικότερα ε, στον κρίσιμο, τομέα των πολιτικών ελευθεριών, τη δικαιοσύνη ε, και των εσωτερικών υποθέσεων, πρέπει να διατηρηθεί για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τις βασικές αρχές Ευρωπαϊκή Ένωση όπω προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η αλληλεγγύη, η συνεργασία και η δημοκρατία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε, κυρία Χρυσόγωνα. Δύο συνάδελφοι ζήτησαν το λόγο. Ο κύριος Δεχόφσκι, ε, σκιώδης ηγητής. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας για την πρόταση του και να πω ότι κρίμα γιατί πρώτη φορά από τότε που έγινε Ευρωβουλευτής δεν έγιναν επαρκείς διαβουλεύσεις με τους σκιώδεις ηγητές. Εδώ βλέπουμε για πρώτη φορά μερικέ προτάσει του προπολογισμού. Αυτό είναι έλλειψη σεβασμού προ του σκιώδη ηγητέ. Ελπίζω να μην επαναληφθεί με τέτοια κατάσταση. Στον τομέα 3. Για να δούμε τι αυξήσει ε, του προπολογισμού, γιατί είναι θεμελιώδου σημασία. Πολύ φοβούμαι πάντω ότι η, η αύξηση που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2019 δεν είναι αρκετή. Ελπίζω στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο αυτή η εξασφάλιση κονδυλίων για την ασφάλεια και τη μετανάστευση θα σταματήσει. Και να δούμε πώς θα εξασφαλίσουμε τα κονδύλια για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που ανέφερε ο εισηγητής. Πριν όμως συμβούν όλα αυτά, θα πρέπει ήδη για το 2019 ε, εγγυηθούμε κάποια πράγματα, δηλαδή να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στα καθήκοντά μας στα θέματα μετανάστευσης και οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν επαρκή χρηματοδότηση για να ανταπεξέλθουν στην αποστολή τους. Εμείς όχι μόνο είμαστε υπέρ αυτού του στόχου, αλλά και υπέρ ε, του, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης του Ασύλου, του Eurojust και της Europol. Χαίρομαι που ο προπολογισμό για το επόμενο έτος ε, ε, προβλέπει κάποια κονδύλια για το άσυλο, τη μετανάστευση και την ένταξη, ώστε να γίνει μια καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων. Και μαζί με το Ταμείο Συντερική ασφάλεια θέλουμε να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά την παράτυπη μετανάστευση, την τρομοκρατία και τα διασυνοριακά εγκλήματα. Επίσης, ε, η διασυνδέσεις και η σωστή ισορροπία είναι σημαντικό θέμα για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Yes. Yeah, Thank you, Chair, dear colleagues. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Ως σκιώδης ε, για την γνωμοδότηση της ΛΥΜΠΕ τάχθηκα υπέρ των μηχανισμών ευελιξία που θα μας επιτρέψουν να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις και τη μετανάστευση. Χαίρομαι που αυτή η ιδέα έχει συμπεριληφθεί και στο σχέδιο γνωμοδότηση του κ. Χρυσόγωνου. Θα πρέπει να τονίσω ότι η στήριξη Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας, η υποστήριξη για το άσυλο είναι πολύ σημαντική. Θέλουμε μάλιστα να γίνει μια κανονική υπηρεσία αυτό το γραφείο στήριξη άσυλο. Κρίμα που ο προπολογισμό της Europol δεν είναι επαρκή, γιατί είναι το δεξί μας χέρι στην προσπάθεια αντιμετώπιση της λαθροδιακίνησης και της πάταξης τη εμπορία ανθρώπων. Πολλά σχέδια της Europol δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη, γιατί δεν υπάρχουν πόροι για την εκπαιδεύσή τους. Είναι παράλογο να έχουμε περιορισμό του προϋπολογισμού κατά 8 εκατομμύρια ευρώ του προϋπολογισμού της Europol για το 2019 σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2018. Θέλουμε να επαναχωρήσουμε σε σχέση με τη δέσμευσή μας να καταπολεμήσουμε το διασυνοριακό έγκλημα. Επίσης, και η Eurojust θα υποστεί περικοπές στο, στη χρηματοδότηση και με, τη χρηματοδο... με την περικοπή της χρηματοδότησης Europol και Eurojust θα υποσκάψουμε την υλοποίηση των προτεραιοτήτων μας. Θα πρέπει να ρίξουμε νερό στο κρασί μας και σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τους πόρους επίσης των βασικών ε, επιχειρησιακών μας οργανισμών. Ευχαριστούμε κύριε Μαμίκινς. Σας ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις σας. Αυτά ως προς το θέμα αυτό δεν έχουμε άλλο χρόνο για τη συζήτηση. Ε, είναι όντως φλέγοντο ζήτημα του προϋπολογισμού και καθόλου εύκολο για το δημοσιονομικό έτος 2019. Το μόνο που μας απομένει είναι να σας αναγγείλω τη διορία για την υποβολή τροπολογιών που είναι για την γνωμοδότηση και το σχέδιο προπολογισμού για το 2019 και τις ε, σχετικές δημοσιονομικές τροπολογίες είναι η 19η Ιουλίου τρέχοντας έτους, 5 το απόγευμα, 19 Ιουλίου. Αυτή είναι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Και αυτά συνάδελφοι, σας ευχαριστώ και πάνω στην ώρα μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι και πάλι ε, δικός μου προβληματισμός και προσωπική και πολιτική μου ανησυχία ή θεωρήσεις και μάλιστα είμαι ο συγγητής της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών για τον κώδικα περί θεωρήσεων και τις ανθρωπιστικές θεωρήσεις. Το έχουμε συζητήσει επανειλημμένως, αλλά έχουμε συμφωνήσει στην ανάγκη να αναπτύξουμε περαιτέρω αυτό το σημείο με μια πολιτική που θα είναι βασικό στοιχείο του χώρου Σέγγεν. Ε, εξετάζουμε εδώ δύο θέματα. Τον ίδιο τον κώδικα για τις θεωρήσεις που είναι πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που ξεκίνησε μάλιστα πριν από τέσσερα χρόνια κατά την έναρξη της τρέχουσας κοινοβουλευτικής θητείας. Μάλιστα δυστυχώς έφτασαν σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις, διακόπησαν και έλαβαν ε, νέα μορφή με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον κώδικα περί θεωρήσεων. Έχουμε όμως και μια έκθεση πρωτοβουλίας, ένα άλλο θέμα που παράλληλα εξετάζουμε, ε, που μου ανέθεσε η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ με θέμα τις ανθρωπιστικές θεωρήσεις, που είναι πολύ ευαίσθητο θέμα και πάγιο αίτημα ε, της πλειοψηφίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να ανταποκριθούμε στο αίτημα να δημιουργήσουμε νόμες διάβλους ε, άφηξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μειώσουμε τη τραγική απώλεια ανθρώπινων ζωών στη Μεσόγειο και να λύσουμε αυτή τη μεταναστευτική κρίση. Δεν υπάρχουν έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα και μετά την ε, πρόταση για τον κώδικα για τις θεωρίες το 2008 που θα διέπει ε, τις προϋποθέσεις για την εισαγωγή στο χώρο Σέγγεν. Το θέμα αυτό του λεγόμενου κώδικα για τις θεωρήσεις ε, έχει σταματήσει και δεν έχει αναθεωρηθεί. Η πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή του 2014, για την οποία είμαι εγώ εισηγητή, απεσύρθη, όπω είπα, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω αδιεξόδου με το Συμβούλιο. Η δική μα Επιτροπή, πάντω, ε, ε, εργάστηκε ακαταπώνητα και πολύ επικοδομητικά και με αμύωτο ενδιαφέρον για την πρόταση. Εκφράσαμε την απογοήτευσή μας για το γεγονός ότι δεν έγινε καμία προσπάθεια από το Συμβούλιο να βρεθεί μια διέξοδος και να ε, ληφθούν υπόψη τα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σήμερα εξετάζουμε τη νέα πρόταση για τον κώδικα θεωρήσεων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ταυτόχρονα θα συζητήσουμε την έκθεση πρωτοβουλία για τι ανθρωπιστικέ θεωρήσει που εκπώνουμε αυτή τη στιγμή. Απέναντι στην απροθυμία του Συμβουλίου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, συμβιβαστούν για το θέμα αυτό. Και με την πρωτοβουλία αυτή ε, διαρευνούμε εναλλακτικές λύσεις για να αποτρέψουμε τη συνέχιση τραγικών και απαράδεκτων θανάτων στη Μεσόγειο. Γιατί πολλοί συνανθρωποί μας παίζουν τη ζωή τους κορώνα γράμματα, είναι διατεθειμένοι να περάσουν πάση θυσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να, περάσουν τα, να φτάσουν στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, για να δούμε ε, τι γίνεται με το με τον κώδικα θεωρήσεων. Καταρχήν θα σας κάνω μια σύντομη εισαγωγή για το θέμα του κώδικα για τις θεωρήσεις και κατόπιν θα ακούσουμε τις παρεμβάσεις των κοινοτικών θεσμικών οργάνων. Ε, πρώτα τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου και μετά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από το Συμβούλιο θα ακούσουμε τον κύριο Καρλ Άγγουστ Λούξ, που είναι πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για τις Θεωρήσεις της Αυστριακής Προεδρίας Καλώς ήρθατε κύριε Λούξ. Θα μας παρουσιάσει εκπρόσωπος της Αυστριακής Προεδρίας ε, τη συζητήσει την κατάσταση των διαπραγματεύσεων στο Συμβούλιο. Μετά θα ακούσουμε την κυρία Γιολάντα Γαγιέκο Κασίλτα Γκράο, που είναι ε, επικεφαλής του τμήματος ε, πολιτικής θεωρήσεων και ασφάλειας εγγράφων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και μετά θα ακούσουμε τους ε, βασικούς ενδιαφερομένους. Θα σας κάνω μια σύντομη εισαγωγή πρώτα απ' όλα, γιατί σίγουρα έχουμε πολλά έγγραφα που περιγράφουν το έργο μας την τελευταία τετραετία. Ανακεφαλαιώνοντας, θα ήθελα να πω ότι έχουμε πρώτα την ρητή απογοήτευσή μας ότι παρά την τεράστια προσπάθεια που κάναμε, αποτέλεσμα δεν έχουμε δει ακόμη. Και νομίζω ότι είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή να δηλώσουμε αυτή την ε, απογοήτευσή μας και την λύπη μας. και την βαθύτατη δυσαρέσκειά μας και ανησυχία ταυτόχρονα για τις τόσο χρονοβόρες προσπάθειες που όμως α, ε, ε, απέβησαν άκαρπες. Η ιδέα εδώ είναι ότι ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε μια πρωτοβουλία για να διευκολύνει την έκδοση θεωρήσεων και να ε, απλουστεύσει, να συντομεύσει τη διαδικασία, να την καταστήσει πιο προσιτή, σε περίπτωση που υπάρχει θεμητός λόγος εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρά την πρόθεση αυτή Τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δυστυχώ δεν κατέστη δυνατό να εγκριθεί η πρόταση και όλε οι προτάσει για τη διευκόλυνση της έκδοση θεωρήσεων παραγωνίστηκαν με μία μονοκοντιλιά στο βωμό της ε, ιδέας της ασφάλειας. Και έτσι επισκιάστηκε όλη η προσπάθεια διευκόλυνση των θεωρήσεων για θεμητούς λόγους, για ε, οικονομικούς, επαγγελματικούς, ε, εκπαιδευτικούς, γιατί πολλοί άνθρωποι έχουν εύλογο ε, συμφέρον και νόμιμο θεμητό συμφέρον να, να, να περάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά τίποτα. Το μόνο επιχείρημα που κυριάρχησε ήταν η ασφάλεια και επισκέσει όλα τα υπόλοιπα επιχειρήματα. Και αυτό είναι αξιολύπητο, είναι εξοργιστικό, αποθαρρυντικό, αποκαρδιωτικό το γεγονός ότι ακόμη περιμένουμε ένα αποτέλεσμα και υλοποίηση του αρχικού στόχου, δηλαδή της διευκόλυνσης της έκδοσης θεωρήσεων για, για νομ, νόμιμους λόγους. Θα πρέπει να βρεθούν τρόποι να πλουστευτούν τα στοιχεία της υποβολής αίτησης. Τα κράτη-μέλη είναι αρμόδια για την εξέταση των γράφων της ιατρικής ε, ασφάλειας και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τα θέματα που είναι πολύ σημαντικά ε, καθορίζουν τη δυνατότητα εκατομμυρίων ανθρώπων να εισέλθουν στο, στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια για νόμιμους λόγους. Και η διαδικασία που προβλέπει ο κώδικας των θεωρήσεων ε, έχουν κρίσιμο ρόλο για πολλούς οικονομικούς παράγοντες, για, για τον τουρισμό, για τις κρουαζιέρες, για τον κλάδο για πολλά επαγγέλματα αλλά και για πολλές περιφέρειες της Ευρώπης όπως ε, για τη δική μου πατρίδα που εξαρτάται από τον τουρισμό σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τις κρουαζιέρες στις Κανάριες νήσους οπότε η ιδέα της διευκόλυνσης δυστυχώς ε, παραγωνίστηκε ε, υπό το πρόσχημα της παρεμπόδισης της μετανάστευσης με πρόσχημα την ασφάλεια. Αναφέρθηκαν πολλά θέματα για την ασφάλεια, την εσωτερική ασφάλεια, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τη διαλειτουργικότητα. Και όλα αυτά κυριάρχησαν και θόλωσαν το τοπίο. Δημιούργησαν μία σύγχυση μεταξύ το θέμα της διαχείρισης της μετανάστευσης και της καταπολέμησης τρομοκρατίας. Δεν ε, είναι ε, ίδιο πράγμα. Άλλο η διαχείριση της μετανάστευσης και άλλο η, αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Αλλά έγινε μια σύγχυση των δύο θεμάτων. Και παρακολούθηκε η όλη διαδικασία για τη διευκόλυνση των θεωρήσεων. Το θέμα είναι να δώσουμε ένα νέο ρόλο στην πολιτική θεωρήσεων και φυσικά υπάρχει σύνδεση μεταξύ κάποιων οικονομικών κριτηρίων και οικονομικών παραγόντων με το θέμα της μετανάστευσης και υπάρχουν και ανησυχίε των κρατών μελών. Ως εκ τούτου, ε, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και το θέμα της πολιτικής επανεισδοχής και της διασυνδέση με το θέμα αυτό. Βέβαια, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η διευκόλυνση ε, των θεωρήσεων ως ε, λόγος ε, για να διαφωνηθούν κάποιες συμφωνίες επανεισδοχής. Αλλά θα πρέπει να δούμε το όλο θέμα στο ισχύον μεταναστευτικό πλαίσιο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν τεκμήρια, δεν υπάρχουν αδιάστητες αποδείξεις για το κατά πόσο η πολιτική θεωρήσεων μπορεί να επηρεάσει ε, ή να βελτιώσει τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες για θέματα επανεισδοχής. Το θέμα αυτό είναι ακόμη προσυζήτηση. Επίση, υπάρχει το θέμα των τρίτων χωρών που δεν έχουν τι ιδιαιτερότητε που απαιτείται από τον κανονισμό για την καλύτερη νομοθεσία και τις κατευθυντήριες γραμμές και την νομοθετική πρόταση για τις νέες διαδικασίες που θα ισχύσουν στο μέλλον. Οπότε, εξακολουθούμε να διατρανώνουμε την προσήλωσή μας στην ανάγκη πρόθεσης ε, και διεκπαιρέωσης αυτής της νομοθετικής διαδικασίας πριν το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής θητείας. Και νομίζω ότι δεν είναι τοπικό ή κάτι τέτοιο, είναι εφικτό. Και θα ακούσουμε τώρα την Αυστριακή Προεδρία, γιατί όπως είπα και χθε στον Αυστριακό Υπουργό, στον Υπουργό Δικαιοσύνης της Αυστρίας, το θέμα αυτό και η Αυστριακή Προεδρία θα είναι η τελευταία εκπεριτροπής Προεδρία που θα είναι λειτουργική για την τρέχουσα νομοθετική διαδικασία. Γιατί η επόμενη Προεδρία του πρώτου εξαμήνου του 2019 θα είναι κυρίως επικεντρωμένη στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το επόμενο, και επίσης ε, δεν θα έχει πολύ έντονες νομοπαρασκευαστικές ε, διαδικασίες, γιατί τα τέλη Μαΐου του 2019 θα έχουμε τις ευρωεκλογέ. Οπότε ουσιαστικά όλοι οι ευρωβουλευτές θα είναι απασχολημένοι με την προεκλογική εκστρατεία στις περιφέρειές τους. Και θα είναι συγκεντρωμένοι στην πολιτική και εκλογική διάσταση του κοινοβουλευτικού του έργου και όχι στην νομοθετική. Οπότε τώρα είναι η ώρα να ανταπεξέλθουμε στο νομοθετικό μας έργο, γιατί γι' αυτό έχουμε εκλεγεί και ειδικά με τη συνθήκη της Λισαβόνας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι νομοθετικό σώμα. Οπότε η Ευστριακή Προεδρία έχει ακόμη μια τελευταία ευκαιρία να συμβάλλει στο να ευοδοθεί αυτή η προσπάθεια και μετά το τούνελ που μας έχει εγκλωβίσει, στο οποίο έχουμε εγκλωβιστεί την τελευταία τετραετία, να δούμε επιτέλους το φως στην άκρη του τούνελ και να εγκρίνουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Περνάμε λοιπόν στην ακρόαση των, των εκπροσώπων των θεσμικών οργάνων και πρώτα στον εκπρόσωπο της Αυστριακής Προεδρίας, τον κύριο Καρλ Όγκουστ Λούξ, που είναι πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για τις Θεωρήσεις. Έχετε το λόγο κύριε Λούξ. Κύριε Ισίτα, κυρίε και κύριοι, όπω είπε ήδη ο εισηγητή, αναλάβαμε το θέμα αυτό που εδώ και αρκετό χρόνο εκκρεμεί, έχει να κάνει με τη φύση του θέματος. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η Προεδρία μας έχει το στόχο να ολοκληρωθεί κατά τη ε, διάρκεια της Προεδρίας μας η εξέταση αυτού του θέματος. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ίσως λοιπόν να χρειαστεί να ολοκληρωθεί λίγο μετά την Προεδρία μας. Στις 14 ε, Μαΐου υπέβαλε νέα πρόταση Κομισιόν και τη συζητήσαμε στο Συμβούλιο. καταλήξαμε σε μια κοινή θέση. Οπότε έχω και την εντολή να ξεκινήσω τις συζητήσεις μαζί σας με βάση αυτή την κοινή θέση. Αυτή η εντολή είναι πολύ κοντά στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που τη θεωρούμε ισορροπημένη. Στόχος μας είναι από τη μία ε, να είναι ανοιχτή η πυρό μας, η, η πυρός μας για τους ε, πολίτες τρίτων χωρών και να απλουστευτούν ε, οι διαδικασίες για τα ταξίδια όσο γίνεται. Όταν λέτε κύριε Σιγητά ότι πρώτα απ' όλα έχει να κάνει με τον τουρισμό, συμφωνώ και η δική μου χώρα εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό και όπως και πολλά άλλα κράτη-μέλη μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα αυτό. Θέλουμε να ευνοηθεί περαιτέρω ο τουρισμός, αλλά και οι άλλες ταξιδιωτικές ε, ε, υποχρεώσεις που έχουν οι πολίτες. Φυσικά θέλουμε οι προϋποθέσεις για την ασφάλεια των πολιτών μας να διατηρηθούν. Τι προβλέπει λοιπόν αυτή η πρόταση. Στο μέτρο, στο μέλλον συγγνώμη, θα είναι πιο εύκολο να πάρει κανείς ε, μια θεώρηση για πολλαπλές εισόδους. Θέλουμε να δώσουν την ευκαιρία στους ε, ταξιδιώτες αν ήδη ε, έχουν λάβει μια βίζα στο παρελθόν να μπορούν κατόπιν να λάβουν μια βίζα που να ισχύει και για μια πενταετία στην πιο συνηθισμένη περίπτωση. Είναι πολύ σημαντικός τρόπος αυτός για να βοηθήσουμε και τις οικονομικές σχέσεις μεταξύ των χωρών αλλά και τον τουρισμό. Μία περαιτέρω διευκόλυνση. Είναι υποβολή ηλεκτρονικά αιτήσεων. Βεβαίω, θέλουμε να κάνουμε αυτό που λέμε μια επίθεση ψηφιοποίηση. Πρέπει να το κάνουν αυτά τα κράτη-μέλη και θέλουν να το κάνουν. Θα δίδεται η δυνατότητα λοιπόν στο μέλλον ακόμη πιο εύκολα στους ε, πολίτε να υποβάλουν επιγραμμικά τι αιτήσει του, χωρί να χρειάζεται να πάνε κάπου χωρίς να χρειάζεται να υποβάλουν χαρτιά. Έτσι μπορεί κάποιος ο οποίος μένει μακριά από τα προξενία να κάνει ε, εύκολα την ε, αίτησή του για βίζα. Κάτι άλλο. Αύξηση της τιμής των θεωρήσεων που έχει μείνει ήδη από το 2006. Γι' αυτό υπάρχει πρόταση να περάσει από 60 στα 80 ευρώ. Αυτή η αύξηση ούτως ή άλλως έχει καλυφθεί από τον πληθωρισμό από το 2006. Δηλαδή στην ουσία είμαστε περίπου στην κατάσταση του 2006. Είναι σημαντικό τα έσοδα να διαμορφωθούν έτσι, ούτως ώστε να μπορούμε να προσλαμβάνουμε επαρκές προσωπικό, να έχουμε επαρκή εξοπλισμό, για να βοηθάμε τους ετούντες. Ούτως ώστε η διαδικασία να είναι όσο πιο απλή και πιο ευχάριστη γίνεται. Αυτό είναι προφανές ότι πρέπει να γίνει σε μια Ευρώπη όπου όλες οι κυβερνήσεις πρέπει να κάνουν περικοπές. Η πολιτική των προσφυγικών θεωρήσεων είναι πολύ σημαντικό στοιχείο στις σχέσεις με τις τρίτες χώρες και μπορεί ε, να παίξει ρόλο μόχλευσης και για άλλους τομείς, για παράδειγμα για την καταπολέμηση της διαφθοράς ή για την καλή διακυβέρνηση. Δεν είναι κάτι καινούριο. Εδώ και χρόνια έχουμε συμφωνίες ε, διευκόλυνσης θεωρήσεων με τρίτες χώρες που πολλές φορές συνδυάζονται με συμφωνίες επιστροφών και με την, ε, ε, το βαθμό της θέλησης των τρίτων αυτών κρατών να δεχθούν τους υπηκόους τους που επανέρχονται από τις δικές μας χώρες. Αυτές είναι οι διαπραγματεύσεις που όπως τις λέμε back to back, δηλαδή συνδέουμε σε πολλές συμφωνίες με τις τρίτες χώρες αυτά τα δύο στοιχεία. Και απόδειξε ότι λειτουργεί αυτή η προσέγγιση ήταν η περίπτωση του Μπαγκλαντές. Είχαμε τρομερά προβλήματα για την επιστροφή υπηκόων του Μπαγκλαντές αλλά με βάση το, την εργαλειοθήκη του Κορεπέρ όπως την αποκαλούμε τα κράτη-μέλη αξιοποίησαν τις διαπραγματεύσεις για τις βίζες ούτως ώστε με σταδιακό τρόπο να καταφέρουμε κάτι. Υπάρχει μία κλιμάκωση. Κυρίως θέλουμε να ε, εντοπίσουμε εκείνους οι οποίοι ε, θα μπορούσαν να κάνουν κατάχρηση αυτών των θεωρήσεων είτε με διπλωματικά διαβατήρια. Αλλά εν πάση περιπτώσει οι διευκολύνσεις που θα παρέχει αυτός ο νέος κώδικας για τις βίζες θα βοηθήσει και τα κράτη-μέλη και η μακροχρόνια βίζα επίσης θα βοηθήσει. Αλλά βεβαίως αυτά δεν θα πρέπει να οδηγήσουν σε τρομερές δαπάνες για τα κράτη-μέλη. Είναι ένα μέσο που το αξιοποιούμε επιτυχημένα εδώ και πολλά χρόνια. Και η περίπτωση του Μπαγκλαδές όπως είπα δείχνει ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις συζητήσεις για τις βίζες για άλλα θέματα. Τώρα κάτι άλλο είναι το outsourcing, δηλαδή εξωτερική, ε, εξωτερικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με την ε, διαμεσολάβηση για τις ε, βίζες. Θέλουμε βεβαίως να ελέγχονται Θέλουμε να ε, υπάγονται σε σαφείς διατάξεις για να μην υπάρχουν καταχρήσεις. Γιατί θα έφυγαν πρώτα απ' όλα τους ετούντες και θέλουμε στο μέλλον να βοηθήσουμε να αποφευχθούν ε, οποιασδήποτε καταχρήσεις. Κάτι άλλο σημαντικό για μας. Είναι η εκπροσώπηση του χώρου Σέγγεν, που νομίζουμε ότι είναι ε, μια πολύ επιτυχημένη ιστορία. Για παράδειγμα, κάποια χώρα ε, εξυπηρετεί κάποια άλλη χώρα του χώρου Σέγγεν. Για παράδειγμα, εδώ και πολλά χρόνια, μέσω του outsourcing και μέσω της εκπροσώπησης από άλλη χώρα δεν χρειαζόμαστε 300, 300 ε, σημεία για να ε, λαμβάνουν ε, βίζες ή υπήκοοι των διαφόρων χωρών. Θέλουμε στο μέλλον να δημιουργήσουμε περαιτέρω ένα ευρύτερο δίκτυο. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε όλα τα κράτη-μέλη να αξιοποιήσουν ε, και να εμπλουτίσουν περαιτέρω αυτό το δίκτυο. Βεβαίως θα ήταν προβληματικό αυτό που προβλέπει η αρχική πρόταση όπως βλέπουμε στην περίπτωση του Φίτζι όπου ένα κράτος ε, χρειάστηκε να αναλάβει την εκπροσώπηση όλων των άλλων και τελικά δεν μπόρεσε να τα βγάλει πέρα και έκλεισε αυτό το προξενείο. Και η κατάσταση έγινε ακόμη χειρότερη για αυτό το τρίτο κράτος από την προηγούμενη. Τα μικρότερα κράτη-μέλη, αλλά ακόμη και μεγαλύτερα πρέπει να υπολογίζουν τι αριθμό αιτήσεων θα τους υποβληθεί για να στείλουν επαρκές προσωπικό, επαρκή εξοπλισμό. Και φοβάμαι ότι, όπως δείχνει το παράδειγμα Φίτζο, αλλά και πολλά άλλα, ότι ορισμένες φορές αν αναλάβει κανείς πολλά, μετά δεν τα βγάζει πέρα. Όπως σα είπα, σε γενικές γραμμές είναι πολύ ισορροπημένη η πρόταση τη Επιτροπής. Σε γενικές γραμμές το Συμβούλιο συμμερίζεται την άποψη τη Επιτροπής. Ε, βέβαια, υπάρχουν ε, μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών διαφορετικές απόψει, Αλλά έχουμε κάθε καλή θέληση να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ε, διαφορές απόψεων, ούτως ώστε εφόσον όλες οι πλευρές δείξουν την σωστή διάθεση να καταλήξουμε και θέλουμε οπωσδήποτε να ξεκινήσουμε όπως σας είπα τις οργανικές διαπραγματεύσεις και ή δυνατόν να τις ολοκληρώσουμε πριν τη λήξη της Προεδρίας. Αν θα το καταφέρουμε εξαρτάται από όλους. Και από την Επιτροπή και από εσά, αλλά και από εμά. Αλλά ούτως ή άλλως προσβλέπουμε ήδη στην καλή και επικοδομητική συνεργασία με εσά. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Και χαίρομαι που θα κάνουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων και για την εργασία που έχουμε ενώπιόν μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμεί θέλουμε περιμένουμε εναγωνίως αυτές τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ε, ευρωπαϊκών θεσμών για να υπάρξει μια όθηση και να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε να ολοκληρωθεί αυτό το θέμα. Να ακούσουμε τώρα την άποψη της κυρίας Γιολάντα Καγιέγκο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που προσκαλέσατε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ακρόαση αυτή. Ε, ήδη αναφέρθηκε η, ε, η αναθεώρηση της πρότασης ώστε να βελτιωθούν ε, οι πτυχές εφαρμογής. Εξακολουθούμε να διατηρούμε κάποιες από τις προτάσεις που παρουσιάσαμε το 2014 που σκοπό είχε να βελτιώσει τον κώδικα για τις θεωρήσεις, να είναι κάπως πιο ευέλικτη η διαδικασία και πιο απλή για τους ετούντες. Και υπάρχουν και κάποια παραδείγματα της διευκόλυνσης αυτής ε, είχαν ως αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει ε, να δίνει τη δυνατότητα έξι μήνες πριν το πολύ, σε ε, αντίθεση με, εννέα, ε, με, συγγνώμη, με τρεις μήνες ε, με, στην πιο παλιά πρόταση και εννέα μήνες για τους ναυτικούς είναι η περίοδος που πρέπει να κάνουν την αίτησή τους για τη χορήγηση της θεώρησης. Επίσης προτείνουμε και κάποιες αλλαγές σε θεωρήσεις βραχυπρόθεσμες, βραχίας διαμονής, 10 ημέρες και επίσης κατά περίπτωση αξιολογήσεις όταν χρειάζεται να εξετάσουμε περισσότερο την αίτηση θεώρησης. Υπάρχουν και, μια, και νέα ε, στοιχεία. Ε, το πρώτο είναι η αύξηση των εξόδων για τη χορήγηση θεώρησης, ε, κάτι που δίνει τη δυνατότητα στα προξενία των κρατών μελών να έχουν τα οικονομικά μέσα να μπορέσουν να επεξεργαστούν αυτές τις θεωρήσεις, εναρμονισμένοι κανόνες για τις θεωρήσεις πολλαπλής εισόδου και το τρίτο στοιχείο είναι η χρήση ε, της σημασίας που μπορεί να έχει η ε, θεώρηση ε, στην εξωτερική πολιτική. Αυτό είναι κάτι το οποίο το κάναμε στις διαπραγματεύσεις που αφορούσαν τη σύνδεση της πολιτικής θεωρήσεων και των ζητημάτων επανεισδοχής. Όσον αφορά τώρα τους οικονομικούς πόρους, προτείνουμε την αύξηση των εξόδων. Είχαν παραμείνει ίδια από το 2006, μια μικρή αύξηση, 80 ευρώ και είναι είναι μικρότερη από, αυτά, από αυτήν που άλλοι τουριστικοί προορισμοί ε, χρεώνουν. Έτσι τα κράτη-μέλη θα μπορέσουν να διατηρήσουν ένα επαρκές επίπεδο προσωπικού, αλλά να παρέχουν και καλές υπηρεσίες στους ετούντες. Ε, πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψη ότι για τους περισσότερου ταξιδιώτες ε, το έξοδο, είναι ένα, το έξοδο της θεώρησης είναι ένα μικρό κόστο, ένα κλάσμα των εξόδων του συνολικού ταξιδιού και δεν θα έπρεπε να είναι αποτροπή για, την, ε, για το ταξίδι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση πρέπει να μπορούν οι τακτικοί ε, ταξιδιώτες να έχουν μια θεώρηση πολλαπλής εισόδου μέχρι πέντε έτη. Υπάρχει λοιπόν ένα αλυσιδωτό σύστημα, δηλαδή μια σταδιακή αύξησης ε, σύμφωνα με την ε, σωστή χρήση των προηγούμενων θεωρήσεων. Αυτό σημαίνει εξοικονόμηση κόστου και για τα προξενία και για του ετούντε, και μετά βέβαια θα υπάρχει και μια ε, αντιστάθμιση, πούμε, γιατί θα υπάρχει μια μια θεώρηση που θα διακεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Υπάρχει βέβαια και η αυθόρμητη, ε, το αυθόρμητο ταξίδι, ε, κάτι το οποίο επίση πρέπει να καλύπτεται από το νέο ε, κώδικα θεωρήσεων. επίση. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη πει ότι η πολιτική μα για το θέμα αυτό σκοπό έχει να ενισχύσει την πολιτική των τρίτων χωρών όσον αφορά την επανεισδοχή των παράτυπων μεταναστών. Υπήρξαν εκκλήσει ακόμη και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πολιτική θεωρήση ε, πιο αποτελεσματικά στη συνεργασία με τις τρίτες χώρες και ειδικότερα στον τομέα τη διαχείριση των συνόρων. Το να χρησιμοποιηθεί λοιπόν η πολιτική των θεωρήσεων θα είναι ένα από του μοχλού βελτίωση αυτή τη συνεργασία με τι τρίτε χώρε. γιατί τη Frontex επίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρότεινε ε, πιο συγκεκριμένου όρου. Αν, μια αν ένα κράτο μέλο δεν ε, σέβεται τι υποχρεώσει τη, ε, να μπορεί να χρησιμοποιείται δηλαδή μια θεώρηση σε συγκεκριμένε περιπτώσει και με συγκεκριμένα αντικειμενικά κριτήρια. Αυτή η νέα προσέγγιση δεν θα έχει αντίκτυπο στου ταξιδιώτε, ε, δηλαδή στο δικαίωμά τους να ε, αιτηθούν ε, θεώρηση. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν καθιστά τη διαδικασία πιο, αποτελεσ... πιο απλή, πιο ασφαλή και όσον αφορά τώρα τη διευκόλυνση των ε, φοιτητών και των σπουδών ε, υπάρχει δυνατότητα στα εξωτερικά σύνορα να χορηγείται η θεώρηση υπό συγκεκριμένε προποθέσει βέβαια. Με τι αλλαγέ αυτέ η πρόσβαση για μία ε, νόμιμη πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση διευκολύνεται. Επίση είναι πάρα πολύ σημαντικό να θεωρείται η Ευρωπαϊκή Ένωση ασφαλή προορισμό για του ταξιδιώτε. Με πολύ χαρά λοιπόν θα συνεχίσουμε τι συζητήσει με το Κοινοβούλιο, με το Συμβούλιο για να υπάρξει μια ταχεία έγκριση τη πρόταση. Ελπίζουμε κι εμεί εντό τη Τρέχουσα κοινοβουλευτική Θητεία να ολοκληρωθεί ε, το ε, θέμα αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την πρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα οι εμπλεκόμενοι ενδιαφερόμενοι φορείς ε, με τη σειρά ε, που κάθονται. Ε, βλέπω εδώ την κυρία Ματσάδο, που είναι υπεύθυνη για τις δημόσιες σχέσεις της ΟΤΡΕΚ ξενοδοχείων εστιατορίων καφετεριών στην Ευρώπη, οργανώσει που ανήκουν στην ΕΤ, τον Ευρωπαϊκό Ιδιωτικό Τομέα στον Τουρισμό. Κύριε Ματσάντο, έχετε το λόγο. Σα ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σα, αγαπητά μέλη τη Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, αγαπητοί συνάδελφοι. Σα ευχαριστώ που καλέσατε την ΕΤ, τον Ευρωπαϊκό Ιδιωτικό Τομέα στον Τουρισμό, στην ακρόασή σα. Είμαι μία, είμαστε μία από τις ενώσεις της Ευρωπαϊκές, το ΝΕΤ, που συγκεντρώνει οκτώ διαφορετικές ενώσεις που εκπροσωπούν τον κλάδο του τουρισμού. Τι προσφέρει ο τουρισμός στην Ευρώπη. Προσφέρει περίπου 27 εκατομμύρια θέσεις απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι η μεγαλύτερη σοσιοοικονομική δραστηριότητα, κοινωνικο-οικονομική δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως είναι γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χάνει μερίδιο αγορά και φαίνεται ότι συνεχίζεται αυτή η ευθύνος απορία. Από το 2015 μέχρι το 2016 η διεθνεί αφήξει τουρισμών επηρεάστηκαν από τι τρομοκρατικέ επιθέσεις. Πέρυσι όμως ευτυχώ ε, είχαμε κάποιες ενδείξεις ανάκαμψης με αύξηση 8% της, ε, των αφήξεων, των τουριστικών αφήξεων στην Ευρώπη. Φυσικά χρειάζεται αναθεώρηση τη πολιτική θεωρήσεων για να συνεχίσουμε να προσελκύουμε τον τους τουρίστες και να στηρίζουμε την οικονομική ανάπτυξη. Η πρόταση του 2014 ε, βρίσκεται σε ένα διαφορετικό πλαίσιο σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί σήμερα. Και θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η μελέτη αντικτύπου του 2014 έδειξαν ότι τα κέρδη από την, ε, μια τέτοια διαδικασία μπορούν να δημιουργήσουν 1,3 εκατομμύρια νέες θέσεις απασχόλησης. Το θέμα είναι να κρατήσουμε τα αναμενόμενα κέρδη και να τα αυξήσουμε. Τα αποτελέσματα των δημοσίων διαβουλεύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους κανόνες ε, Σέγγεν έδειξαν ότι ένα των, ένα τρίτο μάλλον των, των ερωτηθέντων είπαν ότι οι τρέχουσες διαδικασίες θεωρήσεων αποτρέπουν τους τουρίστες από το να ταξιδέψουν στην Ένωση. Θέλουμε λοιπόν εύκολες, ε, απλές, προσιτές ε, και οικονομικά επίσης ε, προς τις διαδικασίες για τη χορήγηση θεωρήσεων, που θα πληρούν φυσικά τις υψηλές προδιαγραφές της ασφάλειας. Είμαστε υπέρ της μείωσης του γραφειοκρατικού άχθους, είμαστε υπέρ της απόφασης, ακούσατε τα παραδείγματα και φυσικά μέσα σε 10 μέρε να διεκπεραιώνεται η διαδικασία και όχι 15, να μπορούν 6 μήνε και όχι 3 μήνε να προγραμματίζουν τα ταξίδια του. Αυτό είναι πολύ σημαντικά. Επίση, το μνημόνιο προβλέπει ότι οι σύγχρονες, ε, ε, σύγχρονοι τρόποι επικοινωνία είναι πολύ πιο εύκολοι. Δεν χρειάζεται αυτό προσώπος να πηγαίνει στο προξενείο. Επίση, το άρθρο 28 περιλαμβάνει την ίδια ιδέα. Και όπω ακούσαμε, χαιρόμαστε για τη δυνατότητα ε, ε, υποβολή αίτηση στα εξωτερικά σύνορα. Αυτό προωθεί τον τουρισμό, αλλά θα πρέπει φυσικά να γίνεται αφού έχουν προηγηθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας. Ε, έχουμε και εμείς όμως κάποιες ανησυχίες. Καταρχήν σε ό,τι αφορά τι θεωρήσει πολλαπλών εισόδων. Είμαστε υπέρ τη εκτεταμένη χρήση, αλλά το σύστημα τη αλληλουχία που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Cascade System έχει κάποιε αδυναμίε. Καταρχήν, είναι δυσανάγνωστο, δυσνόητο για του ταξιδιώτε. Επίση, ένα μικρό αριθμό των τουριστών θα εκπλήρει το πρώτο κριτήριο. Θέλουμε λοιπόν αυτές οι βίζες πολλαπλών εισόδων να χρησιμοποιείται ε, από τους ε, ταξιδιώτες που έχουν ε, χρησιμοποιήσει δύο θεωρήσεις την τελευταία διετία. Σε ό,τι αφορά τα ταξιδιωτικά έγγραφα, θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποια εναρμόνιση των γράφων, των δικαιολογητικών. Τώρα, σε ό,τι αφορά την απόδειξη στέγασης, υπάρχουν, όταν υπάρχουν περιπτώσεις ότι έχουν ε, ακυρωθεί κρατήσεις ή δεν εμφανίζονται οι πελάτες ή χρησιμοποιούν πλαστά έγγραφα για τα ταξιδιωτικά πρακτορία αυτό είναι πραγματικά πρόβλημα, είναι πρόβλημα γιατί δεν μπορούν να κάνουν κράτηση αν δεν γνωρίζουν τον αριθμό το, του γκρουπ αλλά αυτό εξαρτάται από το επιτυχή αριθμό των ε, αιτήσεων αλλά χωρίς προηγούμενη κράτηση δεν δίνεται η ακρόαση Γι' αυτό προτείνουμε κάποια ελαστικότητα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ε, ναι, ισχύει είτε η απόδειξη στέγασης ή η απόδειξη επαρκών μέσων για τη διαμονή ή η απόδειξη του πράκτορα ότι έχουν ε, ληφθεί ρυθμίσεις για την κράτηση με βάση το άρθρο 14.1β και το παράρτημα 3α. Επίσης, ε, Έχουμε και κάποιες ανησυχίες για το κόστος, ιδιαίτερα για τους ανηλίκους. Σε περίπτωση που έχουμε ε, ολόκληρη οικογένεια που έρχεται, το κόστος αυξάνεται. Γνωρίζουμε τη θέση των κρατών μελών, την άκουσαμε επανειλημμένως. Θεωρούν ότι ε, θα πρέπει να καλυφθεί το γραφειοκρατικό κόστος. Βέβαια, το τέλος θεώρησης ε, είχε παραμείνει σταθερό για πολλά χρόνια. Αλλά νομίζω ότι είναι κάπως κοντόφθαλμη αυτή η προσέγγιση, γιατί η οικονομική δραστηριότητα των υποκοντρήτων χωρών ε, ανταποκρίνεται, αντιπροσωπεύει το 2% του ΑΕΠ. Οπότε οι κυβερνήσεις θα πρέπει να αντιμετωπίσουν ως επένδυση. Ε, αυτό που μας προβληματίζει είναι όλα, όλα τα συναφή κόστη. Η ταξιδιωτική και η ιατρική ασφάλεια, το κόστος των δικαιολογητικών εγγράφων, ε, το κόστος ε, μετάβασης προς το αρμόδιο γραφείο για την παροχή των βιομετρικών στοιχείων. Αυτό είναι που επιβαρύνει περισσότερο τον τουρίστα. Επίσης, ε, μερικές φορές θα πρέπει κάποιος να ζητήσει άδεια για να διεκπαιρεώσει όλες αυτές τις διατυπώσεις. Οπότε, είτε να μην υπάρξει αύξηση του τέλους θεώρησης, είτε οποιαδήποτε αναθεώρηση του τέλους θεώρησης να αντισταθμιστεί από μείωση των συναφών τελών τη δυνατότητα, για παράδειγμα, να υποβληθεί το αίτημα θεώρηση σε προξενείο άλλη χώρα μέλου. Είμαστε υπέρ τη προξενική συνεργασία και ξέρω ότι οι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών δραστηριοποιούνται, αλλά θα θέλαμε ακόμη ε, μεγαλύτερη δραστηριοποίησή του σε περίπτωση που το επιθυμούν οι ταξιδιώτες, οι τουρίστες. Η πλήρης ψηφιοποίηση ε, του συστήματος ε, αίτησης θεωρήσεων επίγει και ε, δεν θα πρέπει να στηριζόμαστε αποκλειστικά στο σύστημα με υπόθεμα χαρτί. Χρειαζόμαστε διαλειτουργικότητα του συστήματος. Ξέρω ότι ε, θα πρέπει να συνδυάσουμε το αίτιας με το σύστημα πληροφοριών και τις θεωρήσεις και φυσικά ε, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ε, για τους ταξιδιώτες να παρέχουν τέτοια στοιχεία αλλά δεν είναι επαρκή λόγο να μην εκπροσωπούνται τα κράτη-μέλη σε τρίτε χώρε. Αλλιώ θα αποθαρρύνονται οι τουρίστε από το να ταξιδέψουν στο χώρο Σέγγεν. Ευχαριστώ. Ακούσαμε λοιπόν από τον τουριστικό κλάδο οι οποίοι φυσικά έχουν ε, προσδοκίες απλούστευσης των ε, πολυπλόκων διαδικασιών που ισχύουν αυτή τη στιγμή για να εισέλθει κανείς για οποιοδήποτε λόγο απόλυτα νόμιμο στην, ε, στο χώρο Σέγγεν. Τώρα όμως ε, θα ακούσουμε και τους εξωτερικούς ε, παρόχους υπηρεσιών. Έχουμε τον κύριο Chris Dix, ο οποίος είναι επικεφαλής του Business Development VSF, VFS Global, ο οποίος θα μας παρουσιάσει την άποψή του για το θέμα αυτό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που μας ζήτησε να συμμετάσχουμε σε αυτήν την ακρόαση για να παρουσιάσουμε την άποψη των παρόχων υπηρεσιών για το outsourcing των θεωρήσεων. Είμαστε τμήμα της εταιρείας Κουόνι που την, είναι ιδιοκτησία της, ε, ε, του ιδιωτικού κεφαλαίου του. E ο κύριος ε, Καρκάριαν, ο επικεφαλής μας, εφήβρε αυτή την, το outsourcing για τις θεωρήσεις το 2001. Ξέρετε πώς έχει αλλάξει η κατάσταση από τότε. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία μας εξυπηρετεί 59 κυβερνήσεις σε 139 χώρες και έχει 2.630 κέντρα για υποβολή αιτήσεων. Και έχουμε βοηθήσει πάνω με 173 ετούντες βίζα. Ε, είμαστε ένα μεγάλο τμήμα της αγοράς, αλλά δεν είμαστε μονοπόλιο. Είναι πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον. Υπάρχουν πολλές εταιρείε που είναι ιδιαίτερα ενεργές. Άρα πρέπει να βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας και προς τους ετούντες και προς τις κυβερνήσεις. Και το καλωσορίζουμε ιδιαίτερα αυτό. Αλλά τι σημαίνει αυτή η ιδιωτικοποίηση, το outsourcing. Καμιά φορά υπάρχουν παρανοήσεις. Να σας εξηγήσω περί πρόκειται. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Κατόπιν θα ασχοληθώ με τις ε, βελτιώσεις που η εξωτερική εξωτερήκευση έχει δώσει και για τις κυβερνήσεις και για τους ταξιδιώτες και θα ολοκληρώσουμε με κάποιες συστάσεις για το πώς ε, το νομικό πλαίσιο για τις εταιρείε μας θα μπορούσε να βελτιωθεί περαιτέρω για να βελτιώσουμε και εμείς την υπηρεσία που προσφέρουμε στους ετούντες. Αυτό θα είναι το τρίτο σημείο. Πρώτον λοιπόν, υπενθυμίζω, τι κάνουμε εμείς για να ε, μην υπάρχουν παρανοήσεις. Το outsourcing δεν σημαίνει ότι τις αποφάσεις για το ποιο θα πάρει βίζα τη δίνει μια ιδιωτική εταιρεία. Η αρμοδιότητα είναι θέμα των προξενικών αρχών πάντα για την έγκριση της βίζας. Εμείς, ε, οι εξωτερικοί συνεργάτες, οι εξωτερικές υπηρεσίες που βοηθάνε, ε, δεν επηρεάζουν την ε, προξενική απόφαση. Εμείς συλλέγουμε τις αιτήσει, οργανώνουμε το περιεχόμενο, στέλνουμε πακέτα στο προξενείο και όταν ληφθούν οι αποφάσεις από το προξενείο οργανώνουμε την ε, επιστροφή των, των διαβατηρίων με τις βίζες στους ετούντες. Τα κέντρα μας αυτά παρακολουθούνται στενά από τις επιχειρήσεις και χαιρετίζουμε νέες προτάσεις που θα εντείνουν αυτή την επίβλεψη. Η επιχείρησή μας βασίζεται στην αξιοπιστία. Είμαστε υπέρ του δίκαιου ανταγωνισμού, αλλά δεν θέλουμε χαμηλού επίπεδου εταιρείε να καταστρέψουν την εμπιστοσύνη που έχουμε δημιουργήσει με τις κυβερνήσεις εδώ και χρόνια. Γι' αυτό θα θέλαμε η Ένωση να θέσει ακόμη πιο απαιτητικά απαιτητικέ ελάχιστες προδιαγραφέ. Δεύτερο σημείο. Η, εξωτερική, η εξωτερήκευση είναι ο καλύτερο τρόπο οι κυβερνήσει να βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών. Ποιε είναι οι προκλήσει που αντιμετωπίζουν οι κυβερνήσει. Τι ξέρετε, όσο και εγώ. Υπάρχουν πολλέ αιτήσει, χρειάζεται πιο, περισσότερο προσωπικό, χώρο, υπάρχουν θέματα ασφάλεια που ήδη αναφέρθηκαν. Και όλοι αυτοί οι περιορισμοί σημαίνουν κόστος. Αλλά παράλληλα πολλές κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν ε, περιορισμό των ε, προπολογισμών τους. Οπότε εμείς, μια εξωτερική υπηρεσία, μπορούμε να προσαρμόσουμε καλύτερα τις υπηρεσίες μας με βάση και την αμοιβή που λαμβάνουμε. Και αν ε, υπάρχουν περισσότερες αιτήσει, μπορούμε να επενδύσουμε και περισσότερες υπηρεσίες που, που παρέχουμε. Εμείς μπορούμε να μεγαλώσουμε τα κέντρα μας, να προσλάβουμε περισσότερο προσωπικό, εάν προβλέπουμε περισσότερες αιτήσει. Μπορούμε να προσαρμοστούμε καλύτερα στις εναλλαγές της ε, ζήτησης. Ενώ η πείρα έδειξε ε, ότι πολλά προξενία δεν είναι σε θέση να κάνουν τέτοιες προσαρμογές με την αναγκαία ευελιξία που μπορούμε εμείς. Αυτή η προσαρμοστικότητα σημαίνει ότι δεν ε, υπάρχουν πια αυτές οι ουρές που βλέπαμε μπροστά από τα προξενία που ξεκίναγαν ε, μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα και όπου υπήρχε έφορο έδαφος για οποιοδήποτε προσπαθούσε να γδάρει τους ετούντες. Πολλές φορές, για παράδειγμα, πουλούσαν τη θέση στην ουρά κάποιοι που πήγαν νωρί. Ακόμη και η πρόσβαση στα γκισέ των προξενείων δεν ήταν στην ουσία δωρεάν. Για να φτάσει κανείς σε αυτό το γκισέ έπρεπε να πληρώσει στον δρόμο απ' έξω κάποιον που δεν μπορούσε φυσικά να φτάσει το προξενείο. Και η εξωτερήκευση σημαίνει ότι μπορούν να κάνουν την αίτησή τους μετά από ραντεβού για παράδειγμα γιατί αποφεύγουν αυτές τις ουρές. Και τα προξενία δεν ε, χρειάζεται να δεχτούν τους ετούντες και δεν ε, χρειάζεται να κάνουν τις ε, διοικητικές διαδικασίες ρουτίνας. Άρα μπορούν να επικεντρώσουν περισσότερο στην εξέταση των αιτήσεων επί της ουσίας και έτσι μειώνονται οι καθυστερήσεις ιδιαίτερα στις περιόδους μεγάλης ζήτησης με το σύστημά μας, ο ετών μπορεί να φτάσει τη στιγμή που έχει το ραντεβού του και σε μια ώρα να ξαναφύγει. Όταν ήμουν υπεύθυνο στην Ινδία για τι ε, Βρετανικέ βίζε στην αρχή τη δεκαετία του 2000, κάναμε ό,τι μπορούσαμε, ούτω ώστε όλοι οι ετούντε να λαμβάνουν ε, σε μια μέρα την ε, απάντηση στο αίτημά του, στην αίτησή του. Αλλά δεν καταλαβαίναμε τι κόστο και τι προσπάθεια έπρεπε να κάνουν αυτοί που κάνουν αιτήσει. Έπρεπε να ταξιδέψουν στη νύχτα, έπρεπε να κάνουν χιλιάδες, ε, σε πολλέ ώρε χιλιάδε άτομα, ουρέ ε, στη βροχή, στον ήλιο, με μικρά παιδιά. Όλοι οι ετούντε θεωρούν ότι είναι βελτίωση. Τώρα δίνουμε στου ετούντε και τουριστικέ υπηρεσίε, προωθούμε διάφορου προορισμού και του ε, προετοιμάζουμε για την επίσκεψή του. Οι βίζε μα είναι τώρα πολύ πιο προσβάσιμε στους ε, ε, επισκέπτες, στους ετούντες με πιο, πολύ πιο εύκολο ε, τρόπο. Και διαπιστώνουμε ότι όταν γίνει η εξωτερική, εξωτερήκευση των θεωρήσεων αυξάνεται ο αριθμός των αιτήσεων. Τέλος, για να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε και να επεκτείνουμε τις υπηρεσίες μας προς όφελος των ταξιδιωτών, οι εξωτερικοί πάροχοι θέλουν ένα ευέλικτο νομικό πλαίσιο και παράλληλα αυστηρές προδιαγραφές για να διατηρηθεί και να βελτιωθεί το επίπεδο των υπηρεσιών. Το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο θα μας βοηθήσει όλους. Προστατεύει και τους ταξιδιώτες και τις κυβερνήσεις και τους παρόχους ε, υπηρεσιών γιατί τους δίνει νομική ασφάλεια για την δραστηριότητά τους. Αυτοί οι κανονισμοί όμως πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτοι για να προσαρμόζονται στις νέες ανάγκες και σε νέες τεχνολογικές εξελίξεις. Τα κράτη-μέλη του Σέγγεν πρέπει να υποφεληθούν από αυτές τις ε, αλλαγές για να προωθήσουν τον τουρισμό, την ε, οικονομία τους και για να αξιοποιήσουν πλήρως την εξωτερήκευση. Ο κώδικας για τις βίζες εγκρίθηκε όταν ξεκινούσε η διαδικασία εξωτερήκευσης από τις κυβερνήσεις των χωρών Σέγγεν. Έκτοτε οι κυβερνήσεις και οι εξωτερικοί πάροχοι συνεργάζονται, έχουν γίνει εταίροι ούτω ώστε να βρεθούν λύσεις στις προκλήσεις διαχείρισης ε, των ε, θεωρήσεων. Το VFS Global Χαίρεται για αυτές τις τροποποιήσεις που εισάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι χρειάζονται επιπλέον βελτιώσεις στο κείμενο, ούτως ώστε οι εξωτερικοί πάροχοι να βελτιώσουν ακόμη περαιτέρω την υπηρεσία τους. Για παράδειγμα, ε, υπάρχει μια τροπολογία που λέει ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν ε, δορυφορικά κέντρα υποβολής αιτήσεων όπου δεν εκπροσωπείται κανένα κράτος Σέγγεν. Αυτά τα δορυφορικά κέντρα θα ήταν πραγματική βελτίωση στις υπηρεσίες που προσφέρονται. Αλλά η διαδικασία αυτό σημαίνει και ψηλό κόστο. Και αν είναι πολύ χαμηλός ο αριθμός των, ετούντων, όλα αυτά που χρειάζονται, τα γραφεία, το προσωπικό, βιομετρικό εξοπλισμός, ε, ασφάλεια και κόστος μεταφορέ. Άρα προτείνουμε να το επεκτείνουμε και σε πόλεις όπου δεν υπάρχουν προξενία, όχι μόνο σε χώρες αυτό θα βελτίωνε την κατάσταση. Πρώτα απ' όλα οι ταξιδιώτες θα είχαν πολύ πιο κοντά το κέντρο υποβολής αιτήσεων. Αλλά αυτό θέτει το ευρύτερο θέμα του ότι ε, η αμοιβή για τους παρόχους είναι το 50% του κόστους ε, της ε, θεώρησης αλλά δεν διευκρινίζεται εάν περιλαμβάνει και φόρους πωλήσεων. Εμείς θέλουμε να διευκρινιστεί ότι πρέπει να μην περιλαμβάνει το φόρο πωλήσεων, να προστίθεται ο φόρος πωλήσεων που μπορεί να επιβάλλει κάποιο κράτος. Επίσης ε, θέλω να πω ότι οι ταξιδιώτες είναι ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες μας και το κόστος της αμοιβή μας ποτέ δεν ήταν θέμα. Οι ετούντες με χαρά πληρώνουν αν έχουν καλές υπηρεσίες. Οι Visa Schengen επιτρέπουν πρόσβαση σε 26 χώρες και το κόστος, είναι, το κόστος τους είναι σχετικά χαμηλό σε σχέση με άλλες χώρες όπου πηγαίνουν πολλοί τουρίστες. Επαναλαμβάνω, αυτό που είναι πολύ σημαντικό για τις κυβερνήσεις και τους ταξιδιώτες είναι η ποιότητα των υπηρεσιών που τους παρέχουν οι εξωτερικοί πάροχοι. Ναι, θέλουμε στενότερη επιτήρηση από τα κράτη-μέλη Σέγγεν. Οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο παράρτημα 10 του κώδικα και θα θέλαμε ακόμη πιο αυστηρέ προδιαγραφέ για τι για τις ε, εταιρείε μα, ούτω ώστε οι ταξιδιώτε πάντα να λαμβάνουν τι καλύτερε υπηρεσίε χωρί κρυμμένο κόστο. Η εταιρεία μου με χαρά θα συνεργαστεί με το Κοινοβούλιο για να ε, εκπονήσουμε αυτέ τι ε, προποθέσει. Σα διαβεβαιώ ότι η εταιρεία μου γνωρίζει πλήρω ότι η περαιτέρω αύξηση τη εξωτερήκευση ασχολείται από την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε και προ τι κυβερνήσει και προ του ταξιδιώτε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιώσουμε περαιτέρω το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχουμε μέσω συνεχών επενδύσεων στην καινοτομία, ούτω ώστε να διασφαλίσουμε ότι σήμερα θα είμαστε στο επίπεδο που θα απαιτήσουν οι κυβερνήσει και οι ταξιδιώτε από εμά αύριο. Ιδιαίτερα προωθούμε τι ψηφιακέ λύσει και σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Τηρήσατε ακριβώ το χρόνο σα. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στον επόμενο προσκεκλημένο μα, που είναι ο κύριο Tim, Tim που εκπροσωπεί την Ένωση Πλειοκτητών τη Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ισηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να είμαι εδώ ε, σήμερα σε αυτήν την ακρόαση. Είμαι πρόεδρος της Ένωσης ε, Πλειοκτητών ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ε, Επιτροπής Κοινωνικών Ζητημάτων αυτής που διαμορφώνει την πολιτική σε σχέση με τα πληρώματα των πλοίων. Συμφωνούμε με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές που εκπροσωπεί τους Ευρωπαίους Ναυτικούς Συμφωνούμε λοιπόν με τους κοινωνικούς μας εταίρους προς την άποψή μας ε, από κοινού με το Διεθνές Επιμελητήριο Ναυτιλίας και τη Διεθνή Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές οι οποίοι εκπροσωπούν τους πλειοκτήτες ε, και τους ναυτικούς και τα συμφέροντά τους σε παγκόσμιο επίπεδο έχουμε παρουσιάσει ένα κοινό έγγραφο ανταποκρινόμενοι στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν από τη δημοσίευση της ε, πρότασης ε, της 14η ε, Μαρτίου. Περίπου 90% του ορατού παγκόσμιου εμπορίου μεταφέρεται από εμπορικά πλοία και την χάνει επεξεργασία από, τα λιμένια, από τα λιμάνια παγκοσμίω. Τα λιμάνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι από τα λιμάνια με τη μεγαλύτερη κυκλοφορία γιατί είναι τόποι όπου χιλιάδες ναυτικοί αποβιβάζονται και επιβιβάζονται στα πλοία τους ή παίρνουν την διά τους που είναι απαραίτητη για την ευημερία τους. Υπάρχει μια άρρηκτη σχέση μεταξύ της μετακίνησης των ναυτικών και της διευκόλυνσης του παγκοσμίου εμπορίου. Σε σχέση με την ασφάλεια και την παράτυπη μετανάστευση, το ε, προφίλ κινδύνου των ναυτικών ε, είναι πάρα πολύ ε, χαμηλό. Οι περισσότεροι ναυτικοί εργάζονται στα πλοία χωρίς συγκεκριμένο δρομολόγιο, μη κανονισμένα δρομολόγια και μικρή προειδοποίηση σε σχέση με τα λιμάνια τα οποία θα πιάσουν, που σημαίνει ότι ένα, το ταξίδι ενό ναυτικού πρέπει να οργανωθεί σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και επομένω οι αιτήσει για τι θεωρήσει πρέπει να την χάνουν επεξεργασία σε μικρό χρονικό διάστημα. Για πολλά χρόνια, ναυτικοί τρίτων χωρών έχουν αντιμετωπίσει σοβαρές πρακτικές δυσκολίες προκειμένου να λάβουν θεώρηση για να εισέλθουν να επανεισέλθουν ή να διέλθουν του χώρου Σέγγεν λόγω των διαδικαστικών δυσκολιών και, και των δυσκολι... την διαφορών ερμηνείας των ε, κανόνων. Η πρόταση αναθεώρησης του κώδικα θεωρήσεων είναι μια ευκαιρία για να αναγνωριστεί η ιδιαίτερη, ο ιδιαίτερο χαρακτήρας της εργασία στη θάλασσα και την σημαντική συνεισφορά των ναυτικών στην ευημερία μας. Συνεπώς ε, επικροτούμε την συμπερίληψη του ορισμού ε, για τους ναυτικούς στο άρθρο 2 παράγραφος 12 που θα εξασφαλίζει ότι κανένας ναυτικός δεν θα παραμένει ακάλυπτος. Ε, επίσης χαιρετίζουμε την πρόταση του άρθρου 9 για την παράταση της ε, περίοδου αίτησης για τους ναυτικούς σε 9 μήνες ε, πριν από την ημερομηνία χρήσης της θεώρησής τους, όπως επίσης και αναγνώριση των ιδιαίτερων συνθήκων εργασίας των ναυτικών. Επίσης επικροτούμε την, την προτινόμενη τροποποίηση του άρθρου 23 που θα μειώνει την περίοδο επεξεργασίας των αιτήσεων από 15 σε 10 ημέρες. Αυτό θα είναι υποφελές για τους ναυτικούς γιατί μπορεί να λάβουν εντολές να ταξιδέψουν στο χώρο Σέγγεν και να επιβαστούν σε ένα πλοίο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Το πιο κρίσιμο ζήτημα όσον αφορά τους ναυτικούς είναι η διαθεσιμότητα των θεωρήσεων πολλαπλή εισόδου από πρεσβείες και προξενία των χωρών προέλευσή τους. Οι θεωρήσεις ε, μίας και μόνο εισόδου δημιουργούν δυσκολίες στους ναυτικούς ως προς την επιβίβαση και την αποβίβαση από τα πλοία όταν βρίσκονται ε, στο χώρο Σέγγεν. Η αιτιολογική σκέψη 9 αναγνωρίζει το ότι οι θεωρήσει πολλαπλή εισόδου εξυπηρετούν τα συμφέροντα ε, και των τακτικών ταξιδιωτών αλλά και των προξενείων των κρατών μελών. Ε, σύμφωνα με τους τρέχοντες κανόνες ε, του κώδικα θεωρήσεων του 2009, οι θεωρήσεις πολλαπλής ε, ε, εισόδου θα εκδίδονται στους ναυτικούς. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο άρθρο 24 αποτελεί μια επαναχώρηση στα δικαιώματα των ναυτικών και αυτό μας δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 24, παράγραφος 2α, εισάγει ένα σύστημα ε, διαδοχικότητας για να καθορίσει την επιλεξιμότητα για τις θεωρήσεις πολλαπλής εισόδου. Ε, πρέπει κάποιος να έχει λάβει και να έχει χρησιμοποιήσει τρεις βίζες σε μία διετή περίοδο, ε, κάτι που είναι αδύνατο, με το οποίο είναι αδύνατο να συμμορφωθούν οι πολλοί ναυτικοί. Ένας ναυτικός που είναι 8 μήνες στη θάλασσα και μετά ε, έχει τέσσερις μήνες άδεια πριν από την επόμενη αποστολή του, που πολλοί ναυτικοί το κάνουν αυτό, ε, στην καλύτερη περίπτωση θα έχει την ευκαιρία να λάβει και να χρησιμοποιήσει μόνο δύο θεωρήσεις σε μία περίοδο δύο ετών. Επομένως, ε, όπως είπε και η κυρία Ματσάδο, θα θέλαμε στην παράγραφο 2α να υπάρξει μία τροποποίηση ώστε τα κριτήρια εισαγωγής στο σύστημα αυτό να αλλάξει σε δύο θεωρήσεις ε, κατά τα τελευταία δύο έτη. Όπως προτείνεται στην παράγραφο 24, στο άρθρο 24 παράγραφος 2c, οι θεωρήσεις πολλαπλής εισόδου μπορεί να εκδίδονται σε, σε, ε, στα, στους ναυτικούς ή σε τέτοιου είδους άτομα που έχουν, έχουν πληρώσει τις προϋποθέσεις. Όμως η ειδική αναφορά στους ναυτικούς δεν υπάρχει πλέον, ε, κάτι που θεωρείται επαναχώρηση από, για, τα, για τα δικαιώματα των ναυτικών, γιατί είναι πια δυνητική η διατύπωση και όχι υποχρεωτική. Ε, θα θέλαμε λοιπόν να είναι υποχρεωτική ε, η αναφορά, να είναι shall λοιπόν και όχι may. Ε, λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων εργασίας ε, των ναυτικών που αναγνωρίζονται στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης, είναι απολύτως λογικό να αναγνωρίζεται αυτό και στο αντίστοιχο άρθρο. Οι υποχρεωτικέ θεωρήσει πολλαπλή εισόδου για του ναυτικού θα είχαν ω αποτέλεσμα μεγαλύτερη προβλεψιμότητα ε, και θα μείωναν την ανάγκη ε, αιτήσεων των ναυτικών στα σύνορα της Σέγγεν. Τα κράτη-μέλη εκδίδουν θεωρήσεις στα σύνορα σε πολύ περιορισμένους αριθμούς. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι ναυτικοί μπορεί να μην μπορέσουν να επιβιβαστούν ή να αποβιβαστούν από τα πλοία τους, κάτι το οποίο βέβαια τους αναστατώνει γιατί μπορεί να καθυστερήσει την άφηξη τον επαναπατρισμό τους και να τους παρεμποδίσει από το να ε, πάρουν την άδειά τους. Επίσης, ε, προκαλεί αναστάτωση και στους εργοδότες τους. Ενώ λοιπόν είναι μεγάλη σημασία στο να είναι διαθέσιμες οι θεωρήσεις στους ναυτικούς στην άφηξη στα σύνορα Σέγγεν, ε, το να θεωρηθεί κανόνας ε, αυτό θα, θα μείωνε την, ε, το διοικητικό άχθος ε, για το προσωπικό συνοριακών ελέγχων, συνοριοφυλάκων και θα μείωνε και το άχθος στους πλειοκτήτες και τους άλλους εργαζόμενους στα πλοία. Ε, όσον αφορά τα συνοδευτικά έγγραφα, ε, την, ε, στο άρθρο 14 δεν είναι δεξιοδικό ο κατάλογος και αυτό μας απογοητεύει. Υπάρχουν άνθρωποι που βοηθούν τους ναυτικούς ε, καθημερινά στις αιτήσει του για και ασυνέπειες στα συνοδευτικά έγγραφα λόγω των διαφορών μεταξύ των κρατών μελών στα προξενία τους προκαλούν απώλεια χρόνου και χρήματος. Επίση, μα ανησυχεί πολύ το γεγονό ότι μπορεί να συνδεθεί έκδοση των ε, θεωρήσεων πολλαπλή εισόδου με τη συνεργασία ε, τη χώρα προέλευση του ετούντο με την Ευρωπαϊκή Ένωση σχέση με την επανεισδοχή των παράτυπων μεταναστών. Η προτινόμενη διαδικασία επιτρέπει την αναστολή των δικαιωμάτων σε θεώρηση όλων των υπηκών τη τρίτη χώρα, ε, συγκεκριμένη τρίτη χώρα ή κάποιων κατηγοριών αυτή. Ε, σε αυτή την περίπτωση ε, πρέπει να αναγνωριστεί όχι μόνο η ιδιαιτερότητα ε, του και ο χαρακτήρας της της, α, της άμεσης ανάγκης ταξιδιού ενός ναυτικού, όπως επίσης και το γεγονός ότι το προφίλ κινδύνου τους είναι πάρα πολύ χαμηλό. Θα θέλαμε λοιπόν την αλλαγή στο άρθρο 25α. Επίσης θα θέλαμε να μπορούν οι ναυτικοί να ε, κάνουν αιτήσει στα, στα σύνορα Σέγγεν. στο, η προτείνει στο άρθρο 36.2α ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, διαγραφεί ε, το άρθρο 9 του κώδικα και να υπάρξουν επιπλέον ε, επιχειρησιακές εντολές μέσω ε, εκτελεστικών πράξεων για την ενημέρωση του παραρτήματος. Εμείς θα θέλουμε να συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία ώστε να εξασφαλιστεί ότι ανταποκρίνεται η αλλαγή στις ανάγκες των ναυτικών και του κλάδου. Η δυνατότητα, η ικανότητα των ναυτικών να κάνουν τη δουλειά τους δεν πρέπει να εξαρτάται από την υπηκότητά τους και δεν πρέπει να υπόκειται σε περιορισμούς που ε, περιορίζουν και τα δικαιώματά τους και τη δυνατότητά τους να κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος, κύριε Σπρίγκετ. Που μας παρουσιάσατε την περίπτωση του κλάδου σας. Τώρα θα ακούσουμε την πανεπιστημιακή προσέγγιση. Καλώς ήρθατε κύριε καθηγητά. Ε, Φιλίππο. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Μαρτσέλο τη Φιλίππο, που είναι καθηγητής Διεθνού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Πίζας. Θα μας παρουσιάσει την ε, πανεπιστημιακή σκοπιά και προσέγγιση σε ό,τι αφορά τα ενδεχόμενα κενά, παραθυράκια, δυναμίες, τα υπέρ και τα κατά της τρέχουσας πρότασης για τον κώδικα για τις θεωρίες. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την πρόσκληση, ευχαριστώ τη γραμματεία και θα Ήθελα λίγα δευτερόλεπτα να, του χρόνου μου να αφιερώσω για να εκφράσω τη λανιλεγγύη μου προς τους διερμηνείς που απεργούν εδώ και πολύ καιρό. Γι' αυτό φαντάζομαι ότι είναι σοβαρό το πρόβλημα και ευελπιστώ ότι θα διαθετηθεί η κατάσταση το συντομότερο δυνατό. Ε, καταρχήν, μία σύντομη επισκόπηση Πρώτα απ' όλα οι αδρές γραμμές της παρέμβασής μου και κάποια επιλεγμένα ζητήματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης ή πιο διεξοδικού σχολιασμού σε αυτή τη φάση της διαδικασίας. Επίσης, θα εντοπίσω κάποια προβλήματα που ανακύπτουν και που στο μεταξύ έχουν διαθετηθεί από την πρώτη πρόταση του 2008 με τις νέες προτάσεις του 2014 ή με τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αλλά μερικά προβλήματα <coughs> ανέκυψαν μετά την τελευταία εκδοχή της πρότασης. Κάποιες εισαγωγικέ παρατηρήσεις πρώτα. Συνήθως μιλούμε για την πολιτική θεωρήσεων, αλλά η πολιτική θεωρήσεων δράζεται σε ένα πλέγμα κανόνων δικαίου, που είναι ένα σκλάδος του διοικητικού δικαίου. Και ε, ο κανονισμός είναι πολύ τεχνικός και οι νομοθετικές διατάξεις φαίνονται πολύ ειδικέ και τεχνικές, αλλά θα πρέπει να μας απομακρύνουν από, τους, από τις γενικές αρχές του δικαίου, τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις απαιτήσει του κράτους δικαίου. Το estado de derecho, όπως λέμε στα ισπανικά. Πολλές διατάξεις του κώδικα θεωρήσεων και της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν διαμορφωθεί με τρόπο που ε, χορηγεί στις διοικητικές αρχές, και, δηλαδή κυρίως τα προξενία, τεράστια διακριτική ευχέρεια και περιθώρια για να αξιολογήσουν την κατάσταση. Και αυτό είναι κάπως τρομακτικό από μια πλευρά. Και από την άλλη πλευρά, αν μπούμε στη θέση του ετούντος στη θεώρηση, βλέπουμε ότι είναι τελώς ανήμπορος ε, και αδυνατή να προβλέψει την έκβαση ε, της ε, αίτησή του. Αλλά ακόμη και όταν απορριφθεί η αίτηση θεώρησης, δεν αιτιολογείται διόντως, οπότε δεν κατανοεί για ποιους λόγους απορρίφθηκε ο ετών. Οπότε ο ετών που λαμβάνει την απόφαση της απόρριψης της θεώρησης, του, του αιτήματος θεώρησης, δεν μπορεί καν μερικές φορές να προσφύγει ε, στη δικαιοσύνη για να διορθωθεί η κατάσταση. Γιατί να μην μπορεί λοιπόν να αποταθεί σε ένα δικηγόρο στο δικαστήριο ε, για να ασκήσει τα δικαιώματά του. Αυτό μερικές φορές το ξεχνούμε όταν μιλούμε ε, της προσφυγής, δηλαδή όταν μιλούμε για τον κώδικα θεωρήσεων. Ε, μιλούμε για ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία της ε, ρύθμισης της ε, νόμιμης κινητικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν οι κανόνες της νόμιμης κινητικότητας δεν είναι προσεγμένα, διατυπωμένοι, ένα έμεσο αποτέλεσμα της εφαρμογής τους πολύ σημαντικό είναι ότι οι ο κόσμος καταφεύγει στην παράτυπη μετανάστευση αν δεν μπορούν να αξιοποιήσουν την νόμιμη μετανάστευση. Αν είχαμε καλύτερα διατυπωμένου κανόνες ε, για την νόμιμη μετανάστευση θα είχαμε καλύτερες πρακτικές και θα αποφεύγαμε διακρίσεις στην εξέταση και διεκπαιρέωση των αιτήσεων θεωρήσεων. Οπότε, σε τελική ανάλυση όλα αυτά που θα πω έχουν ένα κοινό παρανομαστή. Την απόπειρα να αναδείξουμε την ανάγκη της αρχής διαφάνειας, ε, μη διάκρισης, ε, χρηστής ε, διαχείρισης και πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Δεν ξέρω πώς από εσά έχετε σκεφτεί τις συνέπειες ε, της ανάγκης να, αποφύγει κανεί, να αποδείξει κανείς την ειλικρινή του πρόθεση να εγκαταλείψει τη χώρα μετά την εκπνοή της θεώρησής του. Το έχετε σκεφτεί αυτό. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το κριτήριο, αυτή η προπόθεση, γιατί είναι πολύ δύσκολο να αποδείξει κανεί την ειλικρινή του πρόθεση. γιατί είναι κάτι που ξεπερνά την υποβολή των δικαιολογητικών εγγράφων. Ο κώδικα θεωρήσεων στη νέα πρόταση δεν αλλάζει την κατάσταση αυτή. Και λέει ότι το προξενείο μπορεί να απορρίψει την αίτηση θεώρησης να αρνηθεί τη χορήγηση, την έκδοση θεώρησης, γιατί ο Ετών δεν έχει ε, αποδείξει επαρκώς την ειλικρινή του πρόθεση να επιστρέψει στη χώρα του, να μην μετατραπεί σε παράνο, παράτυπο μετανάστη. Και αυτή η διάγνωση ουσιαστικά μιας ε, πνευματικής ψυχικής κατάστασης αντιβαίνει στο κράτος δικαίου. Γιατί δίνει ένα όπλο σε κάποιον που θέλει να απορρίψει να το κάνει. Και επίσης ε, καταπατώντας ε, τις στοιχειώδεις αρχές του δικαίου. Και αν επισέλθουμε στις λεπτομέρειες, ε, στο εχειρίδιο περί διαδικασιών, θα διαπιστώσουμε ότι η λογική που χρησιμοποιείται είναι η λογική του υπόπτου, που είναι ακόμη πιο διεξοδική και λεπτομεριακή. Γιατί αναφέρονται κάποια προφίλ προσώπων. Αν διαβάζετε με προσοχή το εγχειρίδιο διαδικασιών θα δείτε τις διαφορές μεταξύ του ε, παντρεμένου, του ε, έχοντος ε, ε, παιδιά. Υπάρχουν διακρίσεις με βάση την οικογενειακή κατάσταση, την εθνικότητα ή την επαγγελματική του κατάσταση. Αν κάποιος είναι καθηγητής νομικής, για παράδειγμα, ή δικηγόρος, ή αν είναι υψηλόβαθμο μέλο μια μη κυβερνητική οργάνωση ή δημόσιο υπάλληλο, θα λάβει την θεώρηση. Αν είναι κανεί εύπορο, θα λάβει τη θεώρηση. Αλλιώ, αν είναι κανεί νέο, αν δεν έχει σταθερή εργασία, αν είναι ανύπαντρο, ή αν προέρχεται από κάποια τμήματα της κοινωνίας από τα χαμηλότερα στρώματα, τότε πολύ πιθανό να απορριφθεί το αίτημά του για χορηγήση θεώρησης. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να καταργήσουμε όλες αυτές τις διακρίσεις ή τουλάχιστον να τροποποιήσουμε τους κανόνες και να προσδιορίσουμε με σαφήνεια ε, πότε μπορεί ε, αυτό το κριτήριο να, ε, το επικληθούν τα προξενία για να αρνηθούν τη χορήγηση θεώρησης. Θέλουμε ένα πολύ πιο αξιόπιστο πρόσωπο, πλαίσιο για τα προξενία για να μπορούν να αποφασίζουν για την αίτηση. Επίσης, η αιτιολόγηση της απόρριψης ή της άνης χορήγησης α, α, θεώρησης. Θεωρείται ότι ε, σε ένα κράτος δικαίου είναι αρκετή αυτή η αιτιολόγηση που προτείνεται γιατί απλώς ο πρόξενος τσεκάρει ένα τετραγωνίδιο και λέει ότι απορρίπτεται το αίτημα θεώρησης για λόγους εθνικής ασφάλειας ή γιατί κάποιος συνιστά απειλή στις διεθνείς σχέσεις ή γιατί ο ετών δεν απέδειξε την ειλικρινή του πρόθεση να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν είναι αιτιολόγηση απόρριψης. Φαίνεται σαν ε, απόρριψη, αλλά είναι μια τυπολατρική και ανεπαρκής αιτιολόγηση. Δεν δίνει στον ετών να καταλάβει γιατί απορρίφθηκε το αίτημά του. Οπότε δεν είναι σύστημα κράτους δικαίου ένα τέτοιο σύστημα. Είναι σαν να γυρίζουμε στο μεσαίωνα που δεν υπήρχε κανένα κράτος δικαίου. Σε αυτά τα θέματα θα πρέπει να βαθύνουμε λοιπόν περισσότερο. Και το καθήκον αναφοράς των λόγων απόρριψης θα πρέπει να επιβάλλεται και να ενισχυθεί αυτό, αυτό το καθήκον αναφοράς διεξοδικών λόγων. Και δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο ή περίπλοκο κάτι τέτοιο. Επίσης το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ήδη έχει υπογραμμίσει ότι οι διοικητικές διαδικασίες που αφορούν αλλοδαπούς και αποφασίζουν για την έκδοση μιας άδειας διαμονής ή την επιστροφή ε, του ενδιαφερομένου αν δεν... είναι σαν να μην υπάρχει υποκειμονικό δικαίωμα για απόκτηση ε, θεώρησης. Ε, ουσιαστικά επιτρέπει διακριτική ευχαίρεια των δημοσίων αρχών και οι αρχές αυτές δεν λογοδοτούν σε κανέναν για την απόφασή τους. Οπότε ουσιαστικά αποδυναμώνεται το δικαίωμα προσφυγής. Χαιρετίζουμε την πρόσφατη απόφαση του ΔΕΚ, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, για την ανάγκη ο, ετών που η απόφαση το έχει απορριφθεί, η αίτηση του έχει απορριφθεί, να έχει δικαίωμα δικαστικής προσφυγής άσκηση έφεση κατά τη απόφαση. Και όποιοι γνωρίζουν, είχαν εμπειρία με τα δικαστήρια, ξέρουν ότι χωρί αιτιολόγηση σε μια απόρριψη ή σε μια αρνητική ε, διοικητική πράξη, υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη δυνατότητα να βρει το δίκαιο του πηγαίνοντα από, στο δικαστήριο. Πάντως η δικαστική προσφυγή θα πρέπει να χορηγείται στον ετώντα τη θεώρηση. Επίσης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες αυτής της κατάστασης. Γιατί αν κανείς μένει στην Αφρική, στην Νότια Αμερική, στην Ασία και λαμβάνει την αρνητική απάντηση του προξένου και γνωρίζει ότι θα πρέπει να πάει στην πρωτεύουσα της χώρας προορισμού της χώρας δηλαδή που ο πρόξενος της είπε όχι στο έτοιμα και θα πρέπει να ε, γύρει τη αγωγή, την προσφυγή στην, στην πρωτεύουσα της χώρας προορισμού. Αυτό δεν είναι δικαιοσύνη. Θα πρέπει να διευκολύνουμε την ε, εύκολη πρόσβαση στη δικαιοσύνη μέσω της χρήσης της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Έχουμε ε, τα εφόδια για κάτι τέτοιο και τα μέσα. Όλα αυτά θα πρέπει να τα εξετάσουμε πολύ πιο διεξοδικά. Επίσης, θα πρέπει να ενισχύσουμε την ε, τοπική προξενική συνεργασία στο χώρο Σέγγεν. Αυτό είναι προ όφελο όχι μόνο των κρατών μελών, αλλά και προ όφελο των ετούντων, θεώρηση. Γιατί να μην χρησιμοποιείται η προξενική συνεργασία για να γίνεται ένα είδο διοικητική αναθεώρηση ε, ε, των αρνητικών αποφάσεων που θα μπορούσε κάλλιστα να γίνεται επιτόπου χωρίς να υποχρεούται ο να βρει δικηγόρο στο, χώ, στο κράτος ε, προορισμού. Και έχουμε πολλά παραδείγματα στο διοικητικό δίκαιο, αλλά και στο ενωσιακό δίκαιο, που δείχνουν τη δυνατότητα ανέβρεσης ρεαλιστικών λύσεων και εφικτών λύσεων για να προσφύγει κανείς κατά μια αρνητικής απόφασης. Και τέλος, ε, κάποια νέα στοιχεία του κανονισμού προβλέπουν ότι η απόκτηση της θεώρησης δεν ε, ε, χορηγεί το δικαίωμα εισόδου. Αυτό το λέει η διεθνής πρακτική. Αν όμως κάποιος έχει λάβει τη θεώρηση σε ένα ταξίδι, θα πρέπει να υπάρχει μια δικαιοσύνη. Σε περίπτωση άσκηση ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα, δεν μπορεί να λέει το κράτος, όχι δεν μπορείτε να περάσετε. Θα πρέπει να διευκρινιστεί η κατάσταση. στον κανονισμό. Και τέλος, κάτι που αναφέρθηκε και προηγουμένως, να μην, φέρ, να μην έρχονται σε ε, δυσμενή θέση οι ετούντες από την ε, συμπεριφορά των δημοσίων αρχών της χώρας προορισμού. Γιατί ε, το να τιμωρείται επειδή η κυβέρνηση μιας χώρας, ε, της χώρας του μάλλον δεν είναι συνεργάσιμη σε θέματα επανειστοχής, θα πρέπει να το καταλογίζεται η απροθυμία της χώρας του να συνεργαστεί και να το πληρώνει με την απόρριψη του αιτήματος θεώρησης. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι δίκαιο το σύστημα, ούτε μια καλή λύση. Επίσης, είναι πολύ κακή η διάταξη της οδηγίας περί επιστροφής, όπου κάποιος μπορεί να μένει σε κράτηση για ένα επιπλέον χρόνο επειδή η κυβέρνηση της χώρας του δεν είναι συνεργάσιμη στην όλη διαδικασία επανειστοχής. Αυτά και ευχαριστώ που με λυπάμαι που μακρηγόρησα. Εμείς ευχαριστούμε. Νομίζω ότι έχουμε μια πλήρη και αντικειμενική εικόνα τώρα με όλες αυτές τις ε, ομιλίες που αλληλοσυμπληρώνονταν και έτσι μας βοηθάνε για να διαμορφώσουμε άποψη για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστούμε λοιπόν όλους. Νομίζω ότι όλοι ασχοληθήκατε με τα θέματα που εντόπισα στην εισαγωγή μου. Όπου ακριβώς ε, τόνισα ότι στόχος της ε, ακρόασής μα είναι να υπενθυμίσουμε ότι οι διαδικασίες τώρα είναι πολύπλοκες, ε, βασίζονται σε μια αρνητική προσέγγιση. Αυτό το τονίσατε εσείς κύριε καθηγητά Ντι Φιλίππο, που το είδατε από μια πανεπιστημιακή άποψη. Θέλουμε λοιπόν να βελτιώσουμε την κατάσταση. Όλες οι ομιλίες τόνισαν ότι πρέπει να διορθώσουμε αυτές τις ανεπάρκειες και το δυσχερές τοπίο και προοπτικές που αντιμετωπίζουν ε, πολλά εκατομμύρια που θέλουν να πάρουν βίζα για να έρθουν στην Ένωση. Και εκτιμώ ε, ορισμένα θέματα που ετέθησαν για τους τουρίστες, για τους ναυτικούς που είναι σημαντικότατος κλάδος για πολλά κράτη-μέλη. Πολλοί λοιπόν χρειάζονται την ε, θεώρηση πολλαπλής εισόδου. Είναι κάτι επί του, οποίου επιμένουμε στη συζήτηση με το Συμβούλιο εδώ και κάποια χρόνια. Έχουμε χρόνο για ανταλλαγή απόψεων. Οι συνάδελφοι, εάν θέλουν να σχολιάσουν, ποιο θέλει το λόγο, ένα, δύο, μάλιστα. Βέβαια, κύριε Μπέκερ. Με συγχωρείτε, δεν βλέπω το όνομά σα. Εσεί, κύριε. Χάλο Άχο από το ECR. Ε, πρώτα εσείς και μετά ο κύριος Μπέκερ. Η ομάδα μας σε μεγάλο βαθμό συμφωνεί με τις απόψεις της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Ενώ παράλληλα μας ενδιαφέρουν ε, και συμφωνούμε με τις επικρίσεις του κυρίου Σπρίγγετ για τις πολλαπλές ε, εισόδους. Η διευκόλυνση κέντρων μετακινήσεων και η ασφάλεια είναι αλληλοσυμπληρώμενα στοιχεία. Η κοινή πολιτική των θεωρήσεων βασίζεται στην εμπιστοσύνη μεταξύ κρατών μελών, όπως και ο χώρος Σέγγεν και το σύστημα Σέγγεν. Πρέπει λοιπόν όλα τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν τους ίδιους κανόνες, να μην υπάρχουν αδύναμοι κρίκοι. Στηρίζουμε τη χρήση της πολιτικής για στι ε, στις ε, διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες που δεν θέλουν να δεχθούν τους πολίτες τους. Αυτό ήδη έχει γίνει από ό,τι άκουσα και έδωσε αποτελέσματα. Τα μέτρα αυτά πιστεύω ότι θα πρέπει να στοχεύουν σωστά τις ελίτ των χωρών αυτών και όχι τους απλούς πολίτες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριο Μπέκερ παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Χαιρετίζω αυτήν την ακρόαση. Πολύ ενδιαφέροντες οι δήμονες. Μας τόνισαν θέματα που και ήδη τα έχουμε αντιμετωπίσει, αλλά και ορισμένα που για πρώτη φορά τα ακούω. Επειδή τώρα θα αρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις ενώ οι ανθρωπιστικές θεωρήσεις θα συζητηθούν χωριστά, είναι σαφές ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με επαγγελματικά ταξίδια, με τουρίστες, ε, αθλητές, καλλιτέχνες. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν σαφείς κανόνες και στόχοι. Και πρέπει να έχουμε και το υπόψη το θέμα bona fide και το θέμα των ναυτικών επίσης. Μας απασχολεί. Δεν ξέρω τώρα ότι ελέγξαμε όλες τις λεπτομέρειες. Και η ψηφιοποίηση βεβαίως. Μείωση του κόστους βεβαίως. Νομίζω ότι συμφωνούμε σε μεγάλο βαθμό. Και κάποια προβλήματα για την ε, χρήση εξωτερικών παρόχων για τις βίζες πρέπει να τα ξαναδούμε. Είχα πολύ θετικές ε, εντυπώσεις από μια επίσκεψη συλλογή στοιχείων στην Κωνσταντινούπολη. Θα τα λάβουμε υπόψη μας λοιπόν και αυτά. Και ο συμπατριώτης μου ανέφερε τα θέματα για τις εκπροσωπήσεις των χωρών, τα προξενία δηλαδή, και πώς μπορούμε να προωθήσουμε το θέμα των βελτίστων αυτών πρακτικών. Θεωρώ επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ισότιμη και δίκαιη συνεργασία με τις τρίτες χώρες και ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε την πολιτική για τις θεωρήσεις ως μέσο πίεσης. Το λέω ανοιχτά. Αυτός είναι καλός τρόπος για να επιτύχουμε άλλα αποτελέσματα. Στο παρελθόν το έχουμε αξιοποιήσει αυτό το μέσο και πρέπει και στο μέλλον να το κάνουμε. Ευχαριστώ για την ενημέρωση που μου έγινε και πιστεύω ότι θα έχουμε καλή συνεργασία. Ευχαριστώ αγαπητέ Άλφε Μπέκερ. Η Έλλη Σλάιν. Ευχαριστώ πολύ. Ένα σύντομο σχόλιο γιατί δυστυχώ ε, ήμουν σε άλλη συνάντηση. Δεν ήμουν εδώ από την αρχή, αλλά με χαράκουσα την παρουσίαση του καθηγητού Ντι Φιλίππο που εκτιμώ πάντα τις ε, παρεμβάσεις του για τα θέματα αυτά. Χουάν Φερνάντο, θέλω να σου παράσχω την πλήρη στήριξή σου στην προσπάθεια να συζητήσουμε το θέμα αυτό εδώ. Πρέπει να είμαστε ειλικρινοί, ειλικρινείς μεταξύ μας. Είμαι η συγγήτρια για τη μεταρρύθμιση του Δουβλίνου από πλευράς της ομάδας μου των σοσιαλιστών. Ένα από τα μεγαλύτερα ελαττώματα του Δουβλίνου είναι ο κανόνας της πρώτης χώρας παράτυπης εισόδου. Αυτό όμως είναι προβληματικό γιατί υπάρχουν τόσο λίγες δυνατότητες ε, ασφαλούς και νόμιμης ε, εισόδου για τους μετανάστες. Γι' αυτό είναι λίγο υποκριτικό να χρησιμοποιούμε αυτό το κριτήριο. Αλλά αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί για να αντιμετωπίσουμε τη διακίνηση, πρέπει να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Ποιε είναι οι νόμιμε δυνατότητε που μπορούμε να παράσχουμε, ούτω ώστε να μπορεί κανεί νομίμω και ασφαλώ να ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά του να κάνει αίτηση ασύλου. Δεν θέλουμε να εξωτερικεύσουμε τα εξωτερικά μας σύνορα με αυτές τις λεγόμενες περιφερειακές πλατφόρμες και η Αφρικανική Ένωση είπε ότι δεν μας ενδιαφέρει, όχι ευχαριστώ. Ούτε η Λιβύη, ούτε η Τινησία. Δεν πάει πουθενά λοιπόν αυτή η ιδέα. Πρέπει να εστιάσουμε στα προγράμματα επανεγκατάστασης, στις ανθρωπιστικές θεωρήσεις, κάτι που είναι οι προτάσεις και τις είπα τις αρμοστίες του ΟΗΕ. Μόνο έτσι θα αντιμετωπίσουμε τους διακινητές και θα δώσουμε μια εναλλακτική λύση. Αν δεν υπάρχουν αυτές οι άλλες εναλλακτικές λύσεις, δεν έχει κανείς δυνατότητα να ζητήσει άσυλο στην Ένωση. Έχεις λοιπόν, Χωάν Φερνάντο, την πλήρη στήριξή μας σε αυτή την προσπάθεια και νομίζω ότι και όλη η τεκμηρίωση που μας δίνεται είναι πολύ χρήσιμη και μας βοηθά. Ευχαριστώ πολύ. Α, και η Μπάρμπαρα Σπινέλη ήθελα να πάρει το λόγο. Καταρχάς, σας ευχαριστώ, Χουαν Φερνάνδο, γιατί δείξατε την αναγκαία επιμονή στον αγώνα που γίνεται αυτόν. Πραγματικά σου είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων γι' αυτό. Και θα σε βοηθήσω και όσο μπορώ Ακούγοντας τις ε, πιο τεχνικές ε, παρουσιάσεις είχα ένα ιδιαίτερα δυσάρεστο συνέστημα ότι τα έχω ξανακούσει όλα αυτά. Θυμάμαι τις διαπραγματεύσεις για την ε, μπλε κάρτα που είναι μια άλλη δυνατότητα νόμιμης εισόδου στην Ένωση για λόγους εργασίας αλλά οι διαπραγματεύσεις απέτυχαν γιατί στο Συμβούλιο δεν υπήρξε ικανοποιητική προσέγγιση. Και, και εσύ πιστεύω, ο Χουαν Φερνάντο είχε την ίδια εμπειρία. Τώρα για αυτόν τον κώδικα για τις θεωρήσεις. Αυτό που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι η συζήτηση για το κράτος δικαίου, όπως το παρουσίασε ο καθηγητής κ. Ντιφιλίππο. Ποιο, θα είναι κατά τη γνώμη μου το πιο σημαντικό στοιχείο στις επικείμενες διαπραγματεύσεις για τον κώδικα για τις βίζες. Τι με ενδιαφέρει περισσότερο. Πρέπει τα πάντα να στηρίζονται στο κράτος δικαίου. Και δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε ορολογία που να μοιάζει με την ιερά εξέταση. Ορισμένοι μιλάνε για προθέσεις και για κυρώσεις. Και ότι ορισμένοι μπορεί να μην κάνουν την αίτηση για θεώρηση με καλή πρόθεση. Μπόνα, φίντε. Δεν είναι θέματα κράτους δικαίου. Αυτά μοιάζουν σαν να είναι εξομολόγηση στον ε, πνευματικό σου για τις αμαρτίες σου. Εάν όμως ως Ένωση απομακρυνθούμε από το κράτος δικαίου, τότε θα προχωρήσουμε σε πολύ περίεργες καταστάσεις. Ξέρουμε τι σημαίνουν αυτά τα περί καλής πίστεως και για εθνικές προελεύσεις. Αυτά ίσχυαν πριν ε, ισχύσει το κράτος δικαίου. Αν θέλουμε λοιπόν να αποφύγουμε ψυχολογικές προηγήσεις πρέπει οπωσδήποτε να το κάνουμε γιατί η ιστορία μας διδάσκει όλα αυτά εάν δεν αποφύγουμε δηλαδή αυτές τις προσεγγίσεις τελικά καταλήγουμε σε διαφθορά Εάν λοιπόν ένας πολίτης τρίτης χώρας δεν μπορεί να εισέλθει νομότυπα λόγω του ότι δεν έχει επαρκή οικονομική επιφάνεια. Ξέρετε τι τεράστια διαφθορά υπάρχει για τις λεγόμενες χρυσές βίζες. Ξέρουμε ότι υπάρχουν φαινόμενα διαφθοράς όχι μόνο στη Μάλτα αλλά και σε άλλες χώρες της Ένωσης, στη Λιθουανία, και την Αυστρία επίσης και στην Πορτογαλία περίπου 11 χώρες 11 χώρες εμπλέκονται σε αυτού του τύπου τις ε, διεφθαρμένες πρακτικές έχουμε αυτές τις ε, δυνατότητες ε, για χρυσές βίζες επειδή κάτι δεν λειτουργεί σωστά στον κώδικα για τις θεωρήσεις επειδή είναι υπερβολικά δύσκολο για κάποιον να πάρει βίζα Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να σας πω ότι συμφωνώ με αυτό που είπατε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό Πραγματικά πιστεύω ότι θα ήταν πολύ σημαντικό να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υπάρχει πλειοψηφία του Κοινοβουλίου εναντί του Συμβουλίου, να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι περνάει από το χέρι μας, για να διευκολύνουμε την εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής. Θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο? Να έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα περαιτέρω διευκρινήσεις Προ την Αυστριακή Προεδρία θα ήθελα να στρέψω το ερώτημα μου. Είπατε ότι θέλετε οι ετούντε να υποβάλουν αιτήσει ε, στο διαδίκτυο, ηλεκτρονικό. Θα θέλα λίγα περισσότερε πληροφορίε σε σχέση με αυτό, κατά πόσο αυτό συμπεριλαμβάνει ολόκληρη τη διαδικασία ή όχι. Και θα ήθελα επίση να καταλάβω λίγο καλύτερα τη θέση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να καταλάβω κατά πόσο έγινε μελέτη αξιολόγηση αντικτύπου λεπτομερή για την εφαρμογή ενό συστήματο ε, ηλεκτρονικού ηλεκτρονικής αίτησης ε, για τις θεωρήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Μπέκερ. Ναι, μια σύντομη συμπλήρωση. Εξέφρασα την ικανοποίησή μου που αντιμετωπίζουμε το θέμα αυτό χωρίς ανθρωπιστικές βίζες των κώδικα θεωρήσεων. Η συνάδελφος ε, όμως έφερε και το θέμα των ανθρωπιστικών θεωρήσεων. Μετά έχουμε μια ακρόαση ακριβώς για τις ανθρωπιστικές ε, θεωρήσεις. Αλλά θα ήθελα να υποφεληθώ από την παρουσία εκπροσώπων της Κομισιόν και του Συμβουλίου να σας παρακαλέσω σύντομα να μας παρουσιάσετε την άποψή σας για το θέμα ανθρωπιστικές θεωρήσεις. Θα μας βοηθήσω πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπέκερ. Καλύτερα να μιλήσουμε ακριβώς με τις ανθρωπιστικές, για τις ανθρωπιστικές θεωρίες στο δεύτερο τμήμα. Το έχουμε ως χωριστό θέμα. Θα ασχοληθούμε πολύ συγκεκριμένα με αυτό το θέμα. Ακούσαμε και τους ευρωβουλευτές και δεν νομίζω να θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο, αν δεν κάνω λάθος. Θα ήθελα όμω και εγώ να ζητήσω κάποιε περαιτέρω διευκρινήσει, ε, αν έχετε την καλοσύνη να μου τις παράσχετε για να μπορέσω να καταλάβω καλύτερα τη ε, δική σας τοποθέτηση που είναι και ο, ο στόχος της σημερινής ακρόασης. Κύριε, μιλήσατε πάρα πολύ για τους ναυτικές ε, εμείς έχουμε λάβει υπόψη ε, το θέμα αυτό ε, στην διαδικασία ε, διαπραγμάτευσης. Βέβαια αυτός ο κλάδος ε, η ναυτιλία, οι πλειοκτήτες, το ε, ανθρώπινο δυναμικό που είναι ναυτική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να, ε, ληφθεί, να ληφθούν υπόψη όταν μιλούμε για τις θεωρήσεις. Αλλά όσον αφορά τις διασώσεις στη θάλασσα, υπάρχει κάποια, κάποιος αντίκτυπος για τους ναυτικούς. Μήπως αυτό δημιουργεί ένα καινούριο πλαίσιο ε, αν, μήπως υπάρχει σχετική νομολογία ή να δημιουργεί ένα προηγούμενο εν πάση περιπτώσει και αυτό που είπε ε, ε, η ECR, ο πρόσωπος της ECR όσον αφορά το ότι μπορεί η πολιτική των θεωρήσεων να συνδεθεί με, το, με την επανεσδοχή. Ε, είναι κάτι που μπορεί να συμβεί. Είναι ένας θεμητός ε, ισχυρισμός. Γιατί υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι συμφωνούν με αυτή τη θέση, άλλοι βέβαια έχουν αντίρρηση στο να υπάρχει αυτή η σύνδεση μεταξύ του κώδικα θεωρήσεων και της πολιτικής επανεσδοχής. Αλλά εγώ θα ήθελα να μου πείτε η εφαρμογή αυτή τη συγκεκριμένη ρήτρα ε, δεν θα πλήξει τον απλό τουρίστα, τον ε, απλό ε, ετούντα θα έχει αντίκτυπο την ε, ελίτ ε, κρατών μελών ε, που θέλει έτσι να, να, να τιμωρήσει τις τρίτες χώρες που δεν συνεργάζονται και θα το κάνει αυτό μέσω της πολιτικής χορήγησης θεωρήσεων. Ακούσατε κάποιες ερωτήσεις, παρακαλώ απαντήστε λάβετε υπόψη βέβαια και το πέρασμα του χρόνου για να έχουμε και χρόνο για το δεύτερο τμήμα της ακρόασης ε, που έχει να κάνει ακριβώς με τις ανθρωπιστικές θεωρήσεις. Το Συμβούλιο παρακαλώ, κύριε Λούξ. Ευχαριστώ κύριε Σίτα. Λοιπόν, από τις τελευταίες προς τις πρώτες. Τι κάνουμε για να πιέσουμε μέσω των ε, θεωρήσεων. Ο στόχος μας δεν είναι να το κάνουμε με πολύ χοντρικό τρόπο. Είναι πολύ στοχευμένα μέτρα. Συγκρίσιμα με αυτά που κάνουμε, για τον κανονισμό 539 για τις απελάσεις. Που ακριβώς προβλέπει στοχευμένα μέτρα. Βεβαίως θέλουμε να ελέγχουμε την κατάσταση, δεν θέλουμε όμως να εμποδίζουμε ούτε τους τουρίστες, ούτε τα επαγγελματικά ταξίδια Θέλουμε να πετύχουμε ακριβώ το στόχο μα. Άλλο θέμα. Ηλεκτρονικέ αιτήσει. Τώρα είμαστε στα Σπάργανα. Τα διάφορα κράτη-μέλη της Ένωσης είναι σε διαφορετικό βαθμό ψηφιοποίηση Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα νομικό μέσο, ώστε να υπάρχει νομική ασφάλεια, ότι είναι δυνατή η ηλεκτρονική αίτηση. Και έχει να κάνει με το πολύ, πολύ περίπλοκο θέμα της ηλεκτρονικής υπογραφής. Είναι εύκολο στη χώρα μου να υποβάλω σε μια αρχή ηλεκτρονική υπογραφή, αλλά για έναν Ρώσο, έναν Πακιστάνο, έναν Κινέζο, είναι πιο δύσκολο να στείλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μία ισχύουσα ηλεκτρονική υπογραφή. Εδώ θα πρέπει στην περαιτέρω διαδικασία να εργαστούμε περαιτέρω. Είναι σημαντικό να υπάρχει δυνατότητα να υποβάλλονται ηλεκτρονικές αιτήσει. Θα διευκολύνουμε έτσι και τον ετούντα αλλά και τα προξενία. Τώρα δεν ξέρω σε τι βαθμό πρέπει να ασχοληθώ με ένα τμήμα της ερώτησης του κυρίου Μπέκερ. Ποια είναι η άποψη της Προεδρίας για τις ανθρωπιστικές θεωρήσεις. Θα επιχειρήσω ως νομομαθής να το αντιμετωπίσω τυπικά. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφερόμαστε στα πλαίσια του κώδικα της θεωρήσης. Θα πρέπει οποιοδήποτε λαμβάνει ε, μία βίζα να, να ξαναφύγει σε 90 μέρες. Όμως, ή ενδεχομένως σε 180 σωσμένες προϋποθέσεις. Οπότε υπάρχει ένα πρόβλημα στην νομική βάση. και χαιρετίζουμε το ότι θα το αντιμετωπίσουμε χωριστά. Γιατί δεν θα πρέπει να υπάρξει σύγχυση των νομικών βάσεων που θα δυσχεράνει την ε, δουλειά για εμάς τους νομομαθείς. Γιατί πάντα ε, οι βίζες συνοδεύονται με 90 μέρες παραμονής. αλλά έχουμε διαφορετικές βίζες. Έχουμε διαφορετικές βίζες, είτε 90 180, αλλά ορισμένες ε, βίζες του εγινε 90 180, ενώ οι εθνικές βίζες μπορεί να είναι και ένα χρόνο. Και όσον αφορά τώρα την άδεια παραμονής, Επιτρέπουν βέβαια μια πιο μακροχρόνια παραμονή εμείς όμως ε, ως ε, νομομαθείς θέλουμε να κάνουμε σαφείς διαχωρισμούς όλων αυτών των δυνατοτήτων. Και γι' αυτό μας ικανοποιεί ότι δεν υπάρχει σύγχυση. Γιατί θα έχουμε πρόβλημα να βρούμε τη σωστή νομική βάση. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα. Κύριε Πρόεδρε, να απαντήσω συντομία σε μερικές ερωτήσεις ευχαριστώντα του βουλευτέ για τα σχόλιά του, αλλά και τι ενώσει, του εκπροσώπους ενώσεων που μίλησαν, γιατί θα συμβάλλουν με τα σχόλιά του ε, στη διαμόρφωση τη πρόταση. Αναφερθήκατε πολύ ε, στο ότι το σύστημα αλληλοδιαδοχής δεν εντάσσεται σε διάφορες κατηγορίες ε, θεωρήσεων πολλαπλών εσόδων. Είπαμε δυνατότητα μέχρι πενταετία για τις ε, θεωρήσεις ε, πολλαπλών εισόδων για ναυτικούς ή άλλες συγκεκριμένες κατηγορίες. Ε, θα πρέπει να έχει δικαιολογημένη πρόθεση για τακτικές, τακτικές μετακινήσεις. Οπότε δεν χρειάζεται να ακολουθούν πιστά το σύστημα Κασκέι τα κράτη-μέλη για τέτοιες ε, εισόδου, για τέτοιες θεωρίες πολλαπλών εισόδων εφόσον θεωρείται καλόπιστο ο ετών ή έχει αποδείξει την πρόθεσή του για τακτικά ταξίδια. Υπάρχει μια ευελιξία στην εφαρμογή των κανόνων. Σε ό,τι αφορά τα σχόλια του καθηγητού Ντι Φιλίππο ε, για το κατά πόσο η πρόταση σέβεται το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Φυσικά και τον τηρεί αυτό το χάρτη. Η Φυσικά απαγορεύονται οι διακρίσεις λόγω φύλου, θρησκείας, εθνότητας και ούτω καθεξής και ως προς τον τύπο υπάρχει υποχρέωση να αναφέρονται οι, οι λόγοι απόρριψης. Θα πρέπει να αναφέρονται ε, η αιτιολόγηση, να γνωρίζει ο τον για ποιο λόγο απορρίφθηκε το αίτημά του. Τώρα είναι σαφή η αιτιολόγηση, αυτό μπορούμε να το βελτιώσουμε στη διατύπωση. Πάντω θα πρέπει να ενημερώνεται ο ετών για του λόγου απόρριψη και υπάρχει δυνατότητα προσφυγή ανάλογα με την νομοθεσία του κάθε κράτους μέρους. Μερικές φορές προβλέπεται και δικαστική προσφυγή. Υπάρχει δυνατότητα ε, προσφυγής και υπάρχει και σεβασμός του κράτους δικαίου για την ψηφιοποίηση, ηλεκτρική, ε, ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων. Ε, ταυτόχρονα με τον κώδικα θεωρήσεων, στις 14 Μαρτίου υποβάλαμε και μια ανακοίνωση και όντως οι ηλεκτρονικές αιτήσει για τις θεωρήσεις είναι το μέλλον και θα διευκολύνουν την κατάσταση και για τα προξενία και για τους ετούντε. Με βάση το σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις, το ΒΙΣ, και μάλιστα το συζητούμε στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο, ε, την αναβάθμιση του συστήματος ΒΙΣ, αυτό χρησιμοποιούν τα προξενία για τη διεκπαιρέωση των αιτήσεων θεώρησης και θέλουμε να το βελτιώσουμε προ όφελο και των ετούντων και των προξενίων. Και μάλιστα ακόμη πιο φιλόδοξα, στα τέλη του έτου, πρόκειται να προτείνουμε μια πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων θεώρησης. Θέλουμε να εφαρμόσουμε πιλωτικά κάποια προγράμματα στα κράτη-μέλη, όχι πλήρως ηλεκτρονικό σύστημα, αλλά να δούμε ποιες πρακτικές ισχύουν στα κράτη-μέλη, τι ε, εργαλεία υπάρχουν και να κάνουμε έναν απολογισμό της κατάστασης προκειμένου στο μέλλον να υποβάλουμε μια πρόταση για περαιτέρω ψηφιοποίηση. Πάντως συμφωνούμε ότι σίγουρα αυτή είναι η σωστή προσέγγιση για το μέλλον. Τώρα η σύνδεση με τη συνεργασία για την επανεισδοχή και θα πρέπει να ισχύει για τον ετώντα. Αυτό ε, γίνεται περιπτωσιολογικά, λαμβάνοντα υπόψη την τρίτη χώρα, την κατάσταση στην τρίτη χώρα και υπάρχει μια ελαστικότητα. Δεν είναι ανάγκη να εφαρμόζεται σε όλου του υπηκού μια χώρα. Μπορεί να εφαρμόζεται σε κάποιε κατηγορίε υπηκών μια χώρα. Και έχουμε ε, μέσα που μας επιτρέπουν το διαχωρισμό και τη δυνατότητα διακοπής ε, της παροχής ε, θεωρήσεων. Επίσης, έχουμε και το θέμα, λαμβάνουμε υπόψη τα δικαιολογητικά έγγραφα. Υπάρχουν ευέλικτοι μηχανισμοί για να λάβουμε υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση του ετώντα. Υπάρχει βέβαια αυτή η δυνατότητα που είναι και εξασφαλίζει και ασφάλεια δικαίου και εξασφαλίζει και τη διαφάνεια. Και, δεν, και είναι και μια ασχατή λύση, δεν είναι η πρώτη μας ε, προσφυγή αυτό το θέμα της επανειστοχής, η διασύνδεση με την επανειστοχή. Ευχαριστώ κύριε Μασάντο. Έχετε κάποια συμπληρωματικά σχόλια, αλλά ο χρόνος τρέχει και μην ξεχνάτε ότι ασκώντας το νόμο δικαίωμα απεργίας η διερμηνείς ανήγγυλαν ότι στις 6.30 ακριβώς θα διακοπεί η υπηρεσία διερμηνίας. Κύριε Μασάντο, ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα σχόλιά της ότι το μέλλον βρίσκεται στην ψηφιοποίηση. Συμφωνούμε απόλυτα με αυτό. Σε ό,τι αφορά τις ε, θεωρήσεις πολλαπλής εισόδου, συμφωνώ και στη μελέτη αντικτύπου αναγνωρίζεται ότι η μέση εγκυρότητα των ε, θεωρήσεων ε, στον Καναδά, είπα και εκείνα, είναι δεκαετούς διάρκειας. Ε, μόνο 5% ε, με βάση από τις διαβουλεύσεις είδαμε ότι θεωρήσει θεωρείς 4-5 ετών. Βλέπετε τεράστια διαφορά με τις ε, ρυθμίσεις άλλων χωρών. Σε ό,τι αφορά το κόστος, η απέτηση της παρουσίας αυτοπροσώπως είναι υπερβολική και αποτρέπει τους ετώντες να καταθέσουν έτοιμα. Και επίσης από τη στιγμή που τα βιομετρικά στοιχεία δίνονται μια φορά και περιλαμβάνονται στο ΒΙΣ, γιατί κάποιο που μπαίνει στο χώρο και λίγε μέρε ή λίγου μήνε μετά θα πρέπει να ε, υποστεί νέο έλεγχο με βιομετρικά στοιχεία. Ε, σε ό,τι αφορά τις εκκλήσεις του ΝΕΤ να ε, έχουμε μια πολιτική που θα ευνοεί τους καλόπιστους ταξιδιώτες και φυσικά θα λαμβάνει υπόψη το κριτήριο της ασφάλειας. Κύριε Δίξ, ευχαριστώ πολύ κύριε Σίγητα. Σε σχέση με τα σχόλια της ε, κυρίας Γκαγιέγκο για την ψηφιοποίηση και την μελέτη μέχρι το τέλος του έτους ή κάποια πιλωτικά προγράμματα από τα κράτη-μέλη, αν θέλει ε, ε, αν θεωρείτε ότι η FS Global μπορεί να συμμετέχει, εμείς για να σας βοηθήσει ευχαρίστως. Κύριε Σπρίγκετ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Ισηγητά. Ε, με, μου κάνατε κι εσείς μία ερώτηση, αλλά θα ήθελα καταρχάς να επανέλθω στο θέμα της προηγούμενης μου παρουσίαση ε, παρουσίασης χάρηκα ιδιαίτερα που άκουσα κάποιους ευρωβουλευτές ε, που είπαν ότι θα λάβουν υπόψη αυτό το ζήτημα και το κατανοούν αλλά θα ήθελα να πω και κάτι που είπε και η κυρία ε, Γκαλιέγκο για τις ε, θεωρήσεις πολλαπλής εισόδου με τους τρέχοντες κανόνες ε, παρά το γεγονός ότι υπάρχει σάλ στο κείμενο, είναι δηλαδή υποχρεωτική η αναφορά στην έκδοση των θεωρήσεων, είναι πολύ σπάνιο στην πράξη ε, να χορηγείται πενταετής θεώρηση και επομένως ε, πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να γίνει μια αλλαγή στο σύστημα αυτό το διαδοχικό για να μπορούν οι ναυτικοί να ε, παίρνουν μια θεώρηση μακράς διαρκείας κατά των πέντε ετών. Ε, αυτό είναι κάτι που θα επιθυμούσαμε. Όσον αφορά ε, τώρα τους ναυτικούς στα εμπορικά πλοία και την διάσωση, το ρόλο τους στη διάσωση, ε, στο πλαίσιο της μετανάστευσης είναι ο παλιότερος κανόνας ε, της ναυτιλίας ε, όταν ένα σκάφος βλέπει ότι υπάρχει άνθρωπος στη θάλασσα πάει να τον βοηθήσει. Αυτό είναι τώρα θεσμοθετημένο στο Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο και μία ακόμη σημαντική διάταξη είναι ότι πρέπει να αποβιβάσουν στον πρώτο λιμένα τον στον οποίο θα φτάσουν το άτομο που έχει διασωθεί. Δεν συμβαίνει πάντοτε και πραγματικά όταν ακούμε στι ειδήσει ότι ένα κράτος μέλος αρνήθηκε τον κατάπλου ενός ε, πλοίου συγκεκριμένη σημαία ε, που είχε διασώσει ανθρώπους ε, στη θάλασσα. Ε, είναι πραγματικά πάρα πολύ ανησυχητικό να το ακούμε αυτό. Πολλές εταιρείε που γνωρίζω εγώ κάνουν λεπτομερείς προετοιμασίες για διέλευση από τη Μεσόγειο θάλασσα γνωρίζοντας ότι θα βρουν άτομα τα οποία πρέπει να διασωθούν. Υπάρχει και κατάρτιση στο πλήρωμά τους ώστε ε, να μπορούν να διασωθούν αυτοί οι άνθρωποι με ασφάλεια και να τους φροντίσουν μέχρι να αποβιβαστούν. Και νομίζω ότι οι εταιρείε αυτές και τα πληρώματα που συμμετέχουν φυσικά πρέπει να επενεθούν για τη δράση τους αυτή. Μερικές φορές τα πληρώματα έχουν ε, λάβει απειλές από τους διασωθέντες, ε, δεν, ότι δεν θέλουν δηλαδή να αποβιβαστούν στις, στο πρώτο λιμάνι. Αυτό Βέβαια μπορεί να είναι μια δύσκολη κατάσταση για ε, τους ναυτικούς, όχι μόνο επειδή έχουν να αντιμετωπίσουν πολλούς ανθρώπους ε, των οποίων η ζωή απειλείται, αλλά ε, και στην αντιμετώπιση των ανθρώπων αυτών. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για την ερώτηση αυτή, κυρία Ισηγητά και πιστεύω ότι είναι ένα σημαντικό ε, σημείο να αναγνωρίσουμε τη σημασία των εμπορικών πλοίων και των ναυτικών ε, σε αυτήν την ε, μενόμενη κρίση. Ευχαριστώ πολύ και ο κύριος Διφιλίππο, καθηγητής Διφιλίππο. Να ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα απαντήσω στα Ιταλικά σε μια ερώτηση της Μπάρμπαρα Σπινέλη. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Μιλήσατε για τη διαφθορά. Είναι ένα από τα προβλήματα όταν δίδονται υπερβολικές εξουσίες ε, στον, δημόσιο, στον δημόσιο τομέα και δεν υπάρχει δυνατότητα να τις ε, ε, διαχειριστούν σωστά Υπάρχουν καταχρήσεις λοιπόν. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι όλα τα προξενία, ε, όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν στα προξενία κάνουν κατάχρηση των εξουσιών τους ε, ε, όσον αφορά πούμε, την επιθυμία εγκατάλειψης μιας χώρας, αλλά είναι μερικές φορές πάρα πολύ δύσκολο να ερμηνευθούν κάποιες καταστάσεις και ο κίνδυνος της διαφθοράς ή της σύγχυσης, για να χρησιμοποιήσω πιο τεχνικό όρο ε, είναι φυσικά υπαρκτό σε μεγάλο βαθμό. Πολλές φορές ε, υπάρχουν ε, νέες γυναίκες ή νέοι άνδρες από συγκεκριμένες χώρες που έχουν, έχουν να αντιμετωπίσουν μια τέτοια κατάσταση και πρέπει να τους διαχειριστούμε με διαφορετικό τρόπο. Πάντα υπάρχει κίνδυνος, δεν υπάρχει τέλεια νομοθεσία, αλλά αν μειώσουμε τους κανόνες ε, και το δημοκρατικό στοιχείο και ε, υπονομεύσουμε τις αξίες μας, ε, τότε αντιβαίνουμε στους στόχους μας. Η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να ξεχνά το γεγονός ότι είναι θεματοφύλακας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας ε, είναι πραγματικά όμως πάρα πολύ δύσκολη και ανησυχητική η κατάσταση. Πρόεδρος, ήθελα να κάνω κάποια καταληκτικά σχόλια, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο, οπότε καλύτερα να πάμε στην, ε, στο δεύτερο κομμάτι της ε, ακροασής μας που αφορά τις ανθρωπιστικές θεωρήσεις. Κύριε Λούξ, κάτι θα ήθελα να πω προς το Συμβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει την πρωτοβουλία και Είδατε εδώ, ακούσαμε μαρτυρίες ε, για τα ε, θεμητά δικαιώματα εκατομμυρίων ανθρώπων ε, να έχουν μία διευκόλυνση στην χορήγηση θεώρησης τους με την, στο πλαίσιο της ομαλής λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της νομικής βάσης που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο της κοινή πολιτικής θεωρήσεων. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε έτοιμοι να συμβιβαστούμε. Το έχουμε δείξει αυτό και γι' αυτό έχουμε αφήσει ε, στην άκρη τις ανθρωπιστικές θεωρήσεις και τους σχετικούς, ε, τις σχετικές μας αξιώσεις που είναι ένα τεράστιο ζήτημα για μας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δικαίως δεν λέω καλά κάναμε συγκεκριμένα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με αυτό το θέμα και να τα καταφέρουμε. Ακούσαμε ας πούμε ε, πολλή επιχειρηματολογία για τη διευκόλυνση για να είναι πιο πρακτική και πιο βιώσιμη όλη η διαδικασία έχουμε περιθώριο ελιγμών, έχουμε χρόνο μπροστά μας, ε, ας το κάνουμε για να μπορέσει να ολοκληρωθεί επιτέλους αυτό το ζήτημα μετά από τέσσερα χρόνια ε, μακρόχρονων διαπραγματεύσεων. Ε, είναι επιτέλους, ε, έχει έρθει επιτέλους ε, η στιγμή να ε, ολοκληρώσει η Αυστριακή Προεδρία, να δεσμευθεί, να αφοσιωθεί ε, στην ολοκλήρωση αυτού του θέματος για την ευημερία όλων αυτών που περιμένουν να ολοκληρωθεί αυτή η νομοθεσία και φυσικά αυτό συμπεριλαμβάνει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να σας πω ποιους έχουμε προσκαλέσει στο δεύτερο ε, πάνελ, γιατί το ζήτημα της ανθρωπιστικής θεώρησης ε, είναι ένα ζήτημα το οποίο ε, το έχουμε αναφέρει πολλές φορές. Να υπενθυμίσω ότι στην αρχή της εντολής αυτής, της κοινοβουλευτικής αυτής θητείας. Η ιδέα ήταν απλώς η απλοποίηση της διαδικασίας. Υπάρχει ένα επιχείρημα για την ουσία της μεταναστευτικής κρίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λέει ότι δεν αφορά τους πρόσφυγες. Η, κρίση με τους πρόσφυγες είναι ουσιαστικά μια πολιτική κρίση η οποία κατά πολλές έννοιες θέτει να αμφιβόλω την πολιτική βούληση ανταπόκρισης ε, με ευρωπαϊκό τρόπο σε ένα κοινό ε, σε μια κοινή πρόκληση που είναι η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων και ειδικότερα των Ευρωπαίων πολιτών ε, εντός των εσωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περί αυτού πρόκειται. Και το έχουμε πει επανειλημμένως ότι έχουν χαθεί πολλές ανθρώπινες ζωές στην προσπάθεια ε, άφηξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όντω πρόκειται για παράτυπη μετανάστευση. Το ομολογούν οι ενδιαφερόμενοι γιατί δεν υπάρχουν νόμιμοι διαβλοί, δεν υπάρχουν νόμιμοι διάδρομοι. Είναι η μόνη λύση που έχουν αυτή η παράτυπη μετανάστευση, αυτή η απόπειρα ε, να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε επίγνωση της ανάγκης να θεσπίσουμε νόμιμους διάβλους, να δημιουργήσουμε ένα νομικό πλαίσιο για την είσοδο στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ασφάλειας και Δικαιοσύνης και στη στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Και ένα από τα βασικά στοιχεία και τα εργαλεία που έχουμε είναι οι ανθρωπιστικές θεωρήσεις. Δεν επινοούμε κάτι, δεν το βγάζουμε το κεφάλι μας. Απλώς ανταποκρινόμαστε σε μία ανάγκη που έχει επανειλημμένως εκφραστεί από πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις, νομομαθείς, ε, συμβούλια, ακόμη και εκκλησίες, εμπειρογνώμονες για θέματα ανθρωπιστικά που απευθύνουν έκκληση προς την καρδιά, την ψυχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θεσπίσει ένα είδος ανθρωπιστικής θεώρησης <laughs> ε, σε ένα όμως ενωσιακό νομικό πλαίσιο και όχι εθνικό πλαίσιο. Να μην επαφείται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών αλλά να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό σύστημα χορήγησης ανθρωπιστικών θεωρήσεων. Και αυτό το θέμα θα εξετάσουμε με τους ε, Καλεσμένος μας εμπειρογνώμονες. Περνάμε λοιπόν στο δεύτερο πάνελ. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Βάουτερ Βαμπάλεγκόη, που θα μας μιλήσει για την ε, μονάδα που εκπροσωπεί την ομάδα Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας ε, της Γενικής Διεύθυνσης του EPRS. Μετά θα ακούσουμε την δόκτωρα Βιολέτα Μορένο Λάξ που θα μας παρουσιάσει τις οικονομικές πτυχές των ε, ανθρωπιστικών θεωρήσεων από το Queen Mary University του Λονδίνου. Μετά την κυρία Μίνα Φερνάντες από το Μιλιέ. Κατόπιν τον κύριο Ντεγέκερ, πρώην Γενικό Πρόξενο της Γαλλίας ε, πρώην επικεφαλής του τμήματος, του κεντρικού γαλλικού τμήματος για την παροχή θεωρήσεων και νυν ε, ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα και τέλος ο κύριος Γιάνν Βαντεβόλτερ από την ε, κοινότητα Σαντεγκίδιο, Τεγκίδιο που έχει ιδιαίτερη εκτίμηση και έγκλης. Θα μας μιλήσει για το ειδικό θέμα αυτής της κοινότητας. Θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Φόουτερ Βαν Μπάλεγκόι που εκπροσωπεί την μονάδα για την ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω πρώτα και μετά θα είναι ο Δόκτωρ Φερνάντες και μετά η Δόκτωρ Μαρίνο Λάξ. Είναι μια πρωτοβουλία ή ε, ένα νομοθέτημα ίδιας πρωτοβουλίας εκφράζει αυτό που θα ήθελε το Κοινοβούλιο και εμείς εδώ κάνουμε μια ευρωπαϊκή αξιολόγηση προστιθέμενης αξίας. Η χρήση αυτής της διαδικασίας είναι να δούμε τι επιπτώσεις και τι προστιθέμενη αξία θα είχαν οι προτάσεις του Κοινοβουλίου. Σε αυτή την περίπτωση είμαστε στην έναρξη της διαδικασίας και το θέσαμε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τις ανθρωπιστικές θεωρήσεις. Εξετάσαμε δύο επιπτώσεις από πλευράς νομικής και θεμελιωδών δικαιωμάτων και οικονομικών και δημοσιονομικών. Αυτά θα τα παρουσιάσουν οι δόκτωρες Φερνάντες και Μορένο Λάξ. Πρώτα απ' όλα, όπως είπατε κι εσείς, όπως έχουν τώρα τα πράγματα, δεν έχουμε ε, σαφή και πλήρη κριτήρια για την χορήγηση ασύλου και δεν υπάρχει και κοινή κατανόηση των ε, διαδικασιών. Πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχουν άλλες διαδικασίες προστατευμένης εισόδου όπως η επανεγκατάσταση. Αλλά συνολικά δεν ε, ανταποκρίνεται στις ανάγκες για άσυλο που υπάρχουν. Η επανεγκατάσταση αφορά μόνο όσους έχουν ήδη αναγνωριστεί ως πρόσφυγες. Δεν αφορά άτομα που δεν έχει καθοριστεί ακόμη το καθεστώς τους. Άρα δεν υπάρχουν νόμιμες διαδικασίες. Και το 90% από όσους λαμβάνουν διεθνή προστασία φτάνουν στην Ένωση μέσω παρατύπων οδών. Αυτή η κατάσταση έχει σοβαρές επιπτώσεις στα άτομα. Ε, υπάρχουν θάνατοι, υπάρχουν επιπτώσεις στην υγεία. Για παράδειγμα, οι 5.000 πνιγμοί το 2016 και που εξακολουθούν. Επίσης έχει υψηλό δημοσιονομικό και οικονομικό κόστος για την Ένωση και τα κράτη-μέλη. Να μην ξεχνάμε ότι η ενωσιακή νομοθεσία δεν είναι μόνο το κόστος που θα προκύψει από την νομοθεσία, αλλά και το κόστος που προκύπτει από την έλλειψη νομοθεσίας. Γιατί χρειάζονται τρομερές χρηματοδοτήσει στον τομέα του ασύλου, του ελέγχου των συνόρων και της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος. Ποια είναι η προστιθεμένη αξία αν έχουμε ένα ε, σαφές σύστημα ανθρωπιστικών θεωρήσεων. Πρώτα απ' όλα θα συμβαδίζει με τις βασικές αξίες. Ε, θεμελιώδη δικαιώματα θα έδινε ασφαλή είσοδο, θα μείωνε την παράτυπη μετανάστευση θα ενίσχυε την νομική ασφάλεια, την προβλεψιμότητα των διαδικασιών, την ε, ενιαία εφαρμογή των νόμων και κανόνων, θα είχαμε καλύτερο συντονισμό της διαδικασίας ασύλου και θα μείωνε, θα το κόστος της υπάρχουσας κατάστασης. Αυτή μας η αξιολόγηση. Εντόπισε τρεις διαφορετικές δυνατότητες για να υπάρξουν ανθρωπιστικές θεωρήσεις. Πρώτον, θα ήταν η προσέγγιση ε, εξαίρεσης από τις θεωρήσεις, που θα σήμαινε ότι για άτομα από ορισμένες χώρες όπου ε, προκύπτουν πρόσφυγες θα εξαιρούσαμε την ανάγκη θεώρησης. Υπήρχε μετά, υπάρχει μετά δυνατότητα της ε, θεώρησης για να ε, εισέλθουν στην επικράτεια του συγκεκριμένου κράτους για να κάνουν αίτηση ασύλου και δεύτερον έχουμε και τις άδειες ταξιδιού για ολόκληρη την Ένωση που θα ήταν μια πιο ενοποιημένη προσέγγιση και θα επέτρεπε να ε, υπάρχει μια διανομή των αιτήσεων μέσω των αντιπροσωπιών της Ένωσης στο εξωτερικό. Αυτή η ε, αξιολόγηση έκανε μια αξιολόγηση για τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων και θεωρεί ότι θα μενόντουσαν και οι παράτυπες ε, είσοδοι, θα γινόντουσαν οι έλεγχοι πριν μπούμε στην Ένωση, χρειάζονται φυσικά ε, νομικές ε, αλλαγές, αλλαγές στην νομοθεσία και θα υπάρξουν και εξοικονομήσεις από αυτό. Εδώ βλέπετε ένα απλουστευμένο πίνακα που θα μας παρουσιάσουν οι επόμενοι ομιλητές. Ε, εφαρμόζουμε τα διάφορα κριτήρια που ανέφερα στις τρεις επιλογές πολιτικής, στις τρεις εναλλακτικές λύσεις. Όλες οι επιλογές και οι τρεις διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις είναι καλύτερες από το status quo. Η κατάργηση, η εξαίρεση από τις βίζες θα ήταν καλύτερη για τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι άλλες δύο εναλλακτικέ θα είχαν σαφή οικονομικά ωφέλη. Πρώτα απ' όλα γιατί θα μειώναμε το κόστος για την εισαγωγή και τις επιστροφές. Γενικά οι επιλογές θα οδηγούσαν σε περισσότερη αποτελεσματικότητα της ε, όλης διαδικασίας χορήγησης ασύλου και καλύτερη κατανομή με βάση την αρχή της ε, αναλογικότητας όλων των κρατών. Τώρα σε 5 λεπτά παρουσίασα ένα κείμενο 90 σελίδων που σας προτείνω να το διαβάσετε το καλοκαίρι και ελπίζω να το ξαναδούμε σε περισσότερη λεπτομέρεια αργότερα και σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Μπαλαγκόη. Θα ακούσουμε τώρα την κυρία Φερνάντες που είπατε θα μιλήσει πρώτα για τις οικονομικές πτυχές των ανθρωπιστικών θεωρήσεων και μετά την καθηγήτρια Μόρεν Ολάξη. Κυρία Φερνάντες, ευχαριστώ. Θα σας παρουσιάσω και εγώ κάποια πορίσματα της έκθεσης που αφορούν τις οικονομικές πτυχές. Επόμενο, επόμενη διαφάνεια. Ε, η παρούσα κατάσταση. Το κόστος της είναι πολλαπλό και μεγάλο. Αυτή ήταν η πρώτη φάση της ε, αξιολόγησης μας ε, και του αντικτύπου στα μεμονωμένα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά. Είδαμε σημαντικές ε, επιπτώσεις. Καταρχήν υψηλό κίνδυνο θανάτου, εκμετάλλευση σωματεμπορία. Ε, πληρώνουν υπέρογκα ποσά στου διακινητέ για να πραγματοποιήσουν το ταξίδι προ την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο αντίκτυπο δεν είναι ίδιο για όλους φυσικά. Πλήττει περισσότερο ε, τα πιο ευάλωτα στρώματα του πληθυσμού, κυρίω γυναίκε και παιδιά, που είναι το μισό αυτών των ε, μεταναστών. Επίσης, για ποιου μιλάμε, οι ε, ετούντε άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 3% του συνολικού πληθυσμού χρηζόντων προστασία με βάση τα στοιχεία της ΥΠΑ του ΟΗΕ. Επίσης, σε ό,τι αφορά τις ε, επιπτώσει στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι χωρίσαμε σε τρει κατηγορίες. Πρώτα, εξωτερικά σύνορα και ασφάλεια. κυρίω παράτυπη μετανάστευση, υπάρχει ε, μεγάλο κόστος για την διαχείριση των συνόρων, την επιτήρηση των συνόρων και τις αποστολές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Δεύτερη κατηγορία ε, είναι οι διαδικασίες ασύλου. Και εδώ το θέμα είναι η έλλειψη διαχείρισης των ε, ροών ε, των αιτήσεων άσυλου και μια οργανωμένη άφηξη των αιτούντων άσυλο και αυτό δημιουργεί αύξηση του κόστους. Και επίσης υπάρχει και κοινωνικό κόστος ό,τι αφορά το οργανωμένο έγκλημα και την παραοικονομία, την ε, άτυπη αγορά εργασία. Σε ό,τι αφορά τις πολιτικές επιλογές, ε, έχουμε μια οικονομική προσέγγιση ε, που καθοδηγεί την επιλογή και τον τρόπο ε, αίτησης ασύλου. Και ε, εξετάζουμε τους διάφορους τρόπους και τις πορείες. Βέβαια υπάρχει και ένα άλλο, άλλος τρόπος στο κόκκινο στη διαφάνεια. Αντί δηλαδή να ζητήσει άσυλο με τους νόμιμους διάβλους, έχουν αναζητήσει, ε, υπάρχει και ένας νέος τρόπος που είναι ανθρωπιστικές θεωρήσεις και με βάση αυτές μπορούν να εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ε, βλέπουμε τι κόστος αντιμετωπίζει ε, ο χρήζων προστασία ε, για να ζητήσει άσυλο. Αυτό που κάνει η ανθρωπιστική θεώρηση είναι να μειώσει το σχετικό κόστος, οπότε ο βασικός αντίκτυπος που βλέπουμε με βάση την οικονομική θεωρία είναι μια αποκατάσταση ουσιαστικά. Δηλαδή είναι σημαντικό αριθμό ε, των μεταναστών που θα ζητούσε με νόμιμου ε, διάβλους ε, το άσυλο στρέφεται πια στις ανθρωπιστικές θεωρήσει. Έχουμε μια μεγάλη μετάβαση, μετατόπιση στον τρόπο, σε διαφορετικό τρόπο τη ασύλου. Επίσης, ένα μικρό, μια μικρή επίπτωση βλέπουμε και στο εισόδημα. Δηλαδή, άτομα της χώρας προέλευσης της γειτονική χώρας με βάση το στατοκβό, ένα τμήμα τους θα ε, εξετάσει αυτή την ε, πολιτική επιλογή, την ανθρωπιστική θεώρηση για να ζητήσει άσυλο. Επίσης, το κόστος ε, της αίτησης ασύλου εξακολουθεί να είναι υψηλό, ανάλογα με το κατακεφαλήν εισόδημα της χώρας προέλευσης. Οπότε, είναι περιορισμένη η εμβέλεια, η χρήση αυτού του μέσου. Οπότε, και οι τρεις ε, αυτές ε, πολιτικές επιλογές ε, είναι προτιμότερες από την παρούσα κατάσταση λόγω του υψηλού κινδύνου και της θρησιμότητας. Η πρώτη πολιτική είναι η εξαίρεση από την υποχρέωση η θεώρηση, είναι η πιο θετική. Έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα και τα 2 και 3 έχουν επιπλέον πλεονεκτήματα για την περίοδο μετά την άφηξη. Τώρα εξετάζουμε το, το κόστος και τα ωφέλη αυτή αυτών των πολιτικών επιλογών. Η πρώτη επιλογή, ε, ελάχιστο κόστος, εξαιρέσεις από τις υποχρεώσεις δηλαδή θεώρησης. Με τις επιλογές 2 και 3 θα έχουμε πιο ε, ε, περισσότερα πλεονεκτήματα στο κόστος. Θα πρέπει όμως να αυξηθεί το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Γραφείου υποστηρίξης Ασύλου για να εφαρμοστεί αυτή η πολιτική. Βασικά ωφέλη. Μείωση της παράτυπης μετανάστευσης. Αυτό είναι το πρωτορχικό όφελος. Ένα επιπλέον όφελος θα είναι καλύτερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και μεγαλύτερη προβλεψιμότητα του συστήματος που είναι χρήσιμη και πριν την άφηξη και μετά την άφηξη του ενδιαφερόμενου. Επίσης, έχουμε κάποια έμεσα ωφέλη ε, σε σχέση με την παρούσα κατάσταση. Ε, σε ό,τι αφορά την επιτήρηση και την διαχείριση των συνόρων, οργανωμένο έγκλημα, ασφάλεια, τρομοκρατία και αναπτυξιακή συνεργασία θεωρούμε ότι το κόστος αυτών των πολιτικών θα μειωθεί χάρη στις ε, νέες επιλογές που προτείνονται. Ε, βέβαια χρειαζόμαστε ε, αποδείξεις που να στοιχειοθετούν αυτά τα πορίσματα και σίγουρα ένα ελεγχόμενο πειραματικό πρόγραμμα των διαφόρων επιλογών θα μας επιτρέψουν μια καλύτερη παρακολούθηση της στρατηγικής και πιο πολλά στοιχεία για τις πολιτικές. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε στις νομικές πτυχές. Ε, η δόκτωρ Βιολέτα Μορένο Λάξ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω με τα βασικά ζητήματα. Τα έχουμε ακούσει ήδη. Το πραγματικό ε, πρόβλημα είναι η πρόσβαση στο άσυλο. Ακούσαμε ότι 90% συνολικού πληθυσμού από αυτούς που μετά χαρακτηρίζονται ε, πρόσφυγες ή δικαιούχοι επικουρικής προστασίας ε, φτάνουν στα κράτη-μέλη παρατύπως μέσω οδών που απειλούν τη ζωή τους. Υπάρχουν βέβαια και άλλα προβλήματα. Υπάρχει ένα πρόβλημα εφαρμογής, ένα αριθμιστικό πρόβλημα Αυτά τα δύο μπορούν να συνοψιστούν ως ύπαρξη ενός νομικού κοινού. Και, ε, και, καινού. Καταρχάς, το πρώτο αφορά ε, την έλλειψη σαφήνειας ε, και πληρότητα των κανόνων για την είσοδο ε, των ετούντων άσυλο και το δεύτερο έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουν τους κανόνες κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, έχουν μια προσέγγιση που την αποφασίζουν τα ίδια κατά τη διακριτική τους ευχέρεια με διαφορετικά κριτήρια είναι διαφορετικές οι προτάσεις εισδοχής και έχουν προκύψει λόγω αυτή τη διαδικασία. Επομένως υπάρχει μια επίγουσα ανάγκη για μια εναρμονισμένη προσέγγιση και αυτό ε, προτείνουμε και εμείς. Ε, για να δούμε τώρα το ρυθμιστικό πρόβλημα που ανέφερα. Υπάρχουν κανόνες, σύνολα κανόνων ε, που αφορούν την είσοδο ε, των ετούντων άσυλο, ε, ο κώδικας των συνόρων Σέγγεν είναι ο πρώτος που έχει να κάνει με τους κανόνες που ισχύουν με τρίτων, για επικός τρίτων χωρών που ζητούν πρόσβαση και είσοδο στα κράτη-μέλη για λόγους διεθνούς προστασίας. υπάρχει μια έλλειψη σαφήνειας και πληρότητα σε σχέση με ε, τον τρόπο της πρόσβασης στην αίτηση ασύλου έχει αντιμετωπιστεί ως τώρα. Ε, μετά έχουμε τη διαδικασία CCV ε, ή το ε, ΣΕΑΣ, δηλαδή δεν υπάρχει κάλυψη των συγκεκριμένων τούτων άσυλο του άρθρου 6 ε, του ε, κώδικα Σέγγεν ούτε στο άρθρο 14 ο κώδικας θεωρήσεων της κοινότητας δεν καλύπτει ε, όσους ε, κάνουν αίτηση θεώρησης και ε, ζητούν άσυλο. Επίσης υπάρχει και το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου που καλύπτει τη διαδικασία με ένα διαδικαστικό τρόπο, δηλαδή υποβάλλεται η αίτηση επισήμως, αλλά το σύστημα δεν ρυθμίζει την πρόσβαση στην ευρωπαϊκή επικράτεια. Οπότε οι αιτούντε άσυλο ουσιαστικά προσωμιώνονται με την κατηγορία των των παρατύπων μεταναστών ε, και πρέπει να αποφύξουν και το ευθύ και το αντιστροφό του. Ε, πρέπει δηλαδή να δείξει κάποιος την δυνατότητα και την πρόθεση επιστροφής στη χώρα προέλευσή τους, ώστε να μπορεί να του δοθεί η δυνατότητα εισόδου. Αλλά αν ισχύει αυτό, τότε αυτός ο παράγοντας δεν τους δίνει τη δυνατότητα της πρόσβασης βάσει του κοινοτικού κεκτημένου. Επομένως και τα δύο καθεστώτα αφορούν ε, ανθρώπους που δεν μπορούν να επιστρέψουν στις θέσεις τους, ε, στις χώρες τους. Αν δηλαδή κάποιος μπορεί να πει ότι μπορεί να επιστρέψει στη χώρα του, αυτό μπορεί να επηρεάσει τη διαδικασία, αλλά παράλληλα δεν θα αναγνωριστούν ως πρόσφυγες. Όσον αφορά τώρα το πρόβλημα ερμηνείας, ε, εκτός από την έλλειψη σαφήνειας του ρυθμιστικού πλαισίου που είδαμε προηγουμένως, η, πρακτική των κρατών μελών βασίζεται στην πεποίθηση ότι δεν υπάρχει υποχρέωση επουδενή χορήγηση θεωρήσεων σε άτομα χρήζοντα διεθνούς προστασίας ε, και ε, αυτές οι διαδικασίες προστατευόμενης εισόδου είναι στη διακριτική ευχαίρεια των κρατών μελών. Και αν δούμε δηλαδή το ε, πρωτογενές και το παράγωγο δίκαιο, ε, βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο έχει ε, συχνά ερμηνευθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Βλέπουμε ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα στο πρωτογενές δίκαιο έχουν ένα ρόλο να διαρματίσουν. Γιατί, γιατί ετούντες άσυλο είναι μια κατηγορία γενική υπηκών τρίτων χωρών ε, που χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση των ε, ε, των αιτήσεων ασύλων, δει τον κανονισμό 539 ε, βλέπει ε, κανείς ότι αυτοί οι υπήκοοι τρίτων χωρών αναφέρονται στο παράρτημα 1 και δεν υπάρχει κανένας λόγος, ε, ούτε νομικός, ούτε λογικός, αυτοί οι άνθρωποι αυτής της κατηγορίας που μετά κάνουν αίτηση για άσυλο στην Ευρωπαϊκή Επικράτη να του χορηγηθεί. Το ίδιο ισχύει για τους ανθρώπους που διέρχονται ή που δείχνουν μία πρόθεση διέλευση των εξωτερικών συνόρων. Είναι το άρθρο 77 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι και αυτό που χρησιμοποιείται ε, στον κώδικα ε, συνόρων Σέγγεν. Δηλαδή οι άνθρωποι που υποβάλλουν αίτηση για άσυλο ε, είναι στην κατηγορία των ανθρώπων που θέλουν να διέλθουν τα σύνορα των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, Αρχίζει να ισχύει εδώ ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτή είναι η ερμηνεία τουλάχιστον ε, στην ε, απόφαση Φράνσον ε, και αναφέρεται και στο άρθρο 51 της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Δεν υπάρχουν λοιπόν καταστάσεις που να καλύπτονται από την ενωσιακή νομοθεσία χωρίς να ισχύει η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ισχύει και το διαβάζω αυτό από την απόφαση Φράνσον γιατί ισχύει η εφαρμογή του, ε, της Χάρτας Εμιλωτών Δικαιωμάτων και η αρχή της μη επαναπροώθησης που αναφέρεται και στο, στα άρθρα 4 και 19.2 της Χάρτας Εμιλωτών Δικαιωμάτων. Οποιοδήποτε μέτρο και η άρνηση βίζας, αν υπάρχει έκθεση λόγω αυτής της άρνησης ενός ανθρώπου σε δίωξη, ε, απαγορεύεται. Και ε, υπάρχει και μία απόφαση Καλταράρου που λέει ότι υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις θετικές που προκύπτουν από το άρθρο 4 ε, της Χάρτας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για να εξασφαλιστεί το γεγονός ότι ε, εξουδετερώνονται τέτοιου είδους κίνδυνοι έκθεσης των ετούντων. Ε, δεν υπάρχει λοιπόν διακριτική ευχέρεια, για, για τα κράτη-μέλη σε κάποιες περιπτώσεις. Με όλα αυτά κατά νου, το, οι δύο διεφαρμογές που έχουν ακολουθηθεί ως τώρα, ε, τα προγράμματα ανθρωπιστικών διαδρόμων, χορηγίας κλπ, που είναι, σημαίνουν μια κατά ερμηνεία, ε, δεν είναι ε, σωστά. Δηλαδή, υπό συγκεκριμένε περιπτώσεις, οι υποχρεώσεις μία επαναπροώθησης μπορεί να δημιουργήσουν θετική θετικά, ε, θετικές υποχρεώσεις που έχουν ως αποτέλεσμα την έκδοση ε, της χορήγησης θεωρήσεων σε όσους χρήζουν ε, διεθνούς προστασίας. Αυτό βέβαια στο πλαίσιο των, της προσέγγισής μας για τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και της πρωτογενούς πρόσβασης των ε, ετούντων άσυλο και των προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Και αυτό το λέω σε σχέση με το πλαίσιο της νομοθεσίας όπως ισχύει αυτή τη στιγμή. Οι λύσεις πολιτικής για τις οποίες μίλησε ο συνάδελφος, ε, δηλαδή αναστολή, η απαλλαγή από τις θεωρήσεις, ε, που θα σημαίνει βέβαια μία τροποποίηση του κώδικα, δηλαδή οι πίκοοι από μία ασφαλή τρίτες χώρες δεν θα χρειάζεται να ε, πάρουν θεώρηση για να ταξιδέψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι να αλλάξουν οι συνθήκες και οι κατάλογοι των θεωρήσεων τροποποιηθούν εκ νέου. Δεύτερη επιλογή θα είναι η χρήση μίας, ε, ενός αναφερειμένου συνόλου κανόνων για τις ε, θεωρήσεις μακράς ε, διαμονής που εκδίδουν τα κράτη-μέλη, οι πρεσβείες των κρατών μελών. Αυτό θα δώσει μια εξατομικευμένη λύση ε, παρά το γεγονός ότι υπάρχει και το Ιταλικό το πρόγραμμα ανθρωπιστικού διαδρόμου στην Ιταλία που θα ακούσουμε λίγο περισσότερα γι' αυτό πιο μετά. Ε, επίσης μια κεντροποίηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή δίνει τη δυνατότητα αίτηση θεώρηση για αίτηση σε άσυλο, να υπάρχουν δηλαδή κάποια κέντρα θεωρήσεων που θα δημιουργηθούν ε, ή μέσω των αντιπροσωπιών της ΕΙΕΒ, με το προσωπικό του ΕΑΖΟ, ε, με ε, την βοήθεια των μη κυβερνητικών οργανώσεων και με τις με την προσβολή αντίθετων αποφάσεων, ε, όπως επίση, πολύ σημαντική θα είναι και η αναδιάρθρωση του συστήματος του Δουβλίνου, να υπάρχει ένα σύστημα μετεγκατάστασης για την υποστήριξη αυτού του, ε, αυτών των λύσεων. Υπάρχουν προβλήματα για ε, τη διαχείριση της συνένεσης που χρειάζεται για αυτή την απαλλαγή από τις θεωρίες. Έχουμε κάνει μια αξιολόγηση των τριών ε, επιλογών και έχουμε αναγνωρίσει τα υπέρ και τα κατά ε, και καταλήξαμε ότι υπάρχει επαρκή νομική βάση στι συνθήκε για κάθε μία από τι τρει εναλλακτικέ επιλογέ. Το άρθρο 77 2α ε, και β σε σχέση με τους ανθρώπους που διέρχονται τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το αρθρο 2 78.2g της Συνθήκης για την ε, Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζητά μέτρα ως με του κοινού συστήματος ασύλου με σκοπό τη διαχείριση των εισρωών των ατόμων που ετούνται ε, διεθνή προστασία δίνει δηλαδή νομοθετική εξουσία στους συνομοθέτες να μπορέσουν να κάνουν τις Αντίστοιχε αλλαγέ Και πάμε και στην επόμενη διαφάνεια να υπάρχει μία σταδιακή προσέγγιση ε, που, θα είναι, που είναι προτιμητέα. Πρώτο στάδιο, το κράτος μέλος ε, που θα δίνει τη θεώρηση μακράς διαμονής ε, πριν από μία κεντρική προσέγγιση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέλος, από απόψε ως δικαιωμάτων, είναι προτιμητέο το πρόγραμμα απαλλαγής από τη θεώρηση. Ο, η, ο εισηγητής δεν έχει συμφωνήσει ρητά με αυτή αυτήν τη λύση, αλλά θεωρούμε ότι είναι ένα σημείο αφετηρία για ε, τη, η σύσταση αυτή. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε τώρα για να υπερβούμε τα μειονεκτήματα της ε, ε μακράς διάρκειας θεώρησης και της σχετικής λύσης, να δούμε δηλαδή ποια είναι τα πλεονεκτήματα του προγράμματος αυτού και να, ε, να υιοθετήσουμε μέτρα τα οποία θα ε, αντισταθμίσουν ε, ενδεχόμενα μειονεκτήματα αυτής της λύσης. Ε, υπάρχει επίσης και το πρόβλημα της αθέτησης υποχρεώσεων, ε, γιατί ε, τα κράτη-μέλη δεν θέλουν ε, να προσελκύσουν περισσότερους μετανάστες λαμβανομένων υπόψη των κανόνων που ισχύουν τώρα στο Δουβλίνο, γιατί το να αφήσουμε όλη αυτή τη διαδικασία 100% στα κράτη-μέλη μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να απορρίπτονται αιτήσει Μπορεί δηλαδή να υπάρξει ένας ε, μηχανισμός εξοεδαφικός ε, για τον καθορισμό του καθεστώτος του πρόσφυγα ε, που θα, είναι, θα περάσει από την πίσω πόρτα. Εμείς δεν θέλουμε κάτι τέτοιο, δεν θέλουμε αυτό να μεταφερθεί σε μια τρίτη χώρα. Θέλουμε ένα σύστημα που να μπορεί κάποιο να ζητήσει μια θεώρηση, να πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά να υποβάλει μια αίτηση για άσυλο βάσει των ισχυών των κανόνων του κοινού συστήματος ασύλου. Αυτό που αναφέρουμε και εμεί στη μελέτη μα και προτείνουμε ω λύσει για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα δύο μειονεκτήματα είναι η εισαγωγή ενό ανεξάρτητου μηχανισμού παρακολούθηση και ενδεχομένω κυρώσεων ε, σε σχέση με τη συμμόρφωση των κρατών ε, μελών ε, βάσει της αρχής αλληλεγγύης και να υπάρξει και μια αντιστοίχηση προτιμήσεων που προβλέπεται στο ΕΑΖΟ και βέβαια αναθεώρηση του Δουβλίνου ε, όπως ε, προβλέπεται και στην πρόταση ε, στην έκθεση ΣΛΑΙΝ... και κεντρική διαχείριση κάποιας, κάποιων ε, εξόδων από τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να μην καλύπτονται κάποια έξοδα από, την, ε, από τα κράτη-μέλη, αλλά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη, να μπορούμε να βασιστούμε στην ε, πληροφορική, στα μηχανογραφημένα συστήματα, συνεργασία με τους μη κυβερνητικέ οργανώσεις και πριν και μετά την άφηξη, να υπάρχει δηλαδή ένας μηχανισμός που θα συνοδεύει καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασία του Ετού και επίση να μην υπάρχουν ε, ε, αντικίνητρα ε, για τη συμμόρφωση των κρατών μελών. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και αναμένω εναγωνίως τα ερωτήματά σας. Εμεί σα ευχαριστούμε. Και τώρα ο κύριο Ντεζεγέρ, που είναι εκπρόσωπος το, του ανεξαρτήτου φορέα MD Visa Consulting. Ευχαριστώ. Εγώ θα μιλήσω καθαρά τεχνικά. Είναι η άποψη των ε, προξενείων που πρέπει να εφαρμόσουν τους κανονισμούς που ψηφίζεται. Οπότε έθεσα την εξής ερώτηση. Οι ανθρωπιστικές θεωρήσεις ανταποκρίνονται στο πρόβλημα. Θα βοηθήσουν να σταματήσει το δράμα της παράνομης μετανάστευσης. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση τι επίπτωση θα είχε για τα προξενία αυτή η βίζα ή τους άλλους διοικητικούς μηχανισμούς που θα ασχολούνται με τις αιτήσει. Πρώτη ερώτηση. Λύνει το πρόβλημα η ανθρωπιστική βίζα. Θεωρώ ότι ο στόχος είναι να δώσουμε θεωρήσεις σε μια ε, καλά καθορισμένη κατηγορία ατόμων. Αλλά είναι πολύ ευρεία. Είναι κάθε άτομο που αιτείται διεθνή προστασία που θεωρεί ότι τη χρειάζεται. Μετά από κάποια χρόνια μεταβατικών περιόδων, αυτή η πρωτοβουλία θα έπρεπε να αφορά τους πάντες. Ο στόχος είναι να επιτρέψουμε σε κάθε άτομο, οπουδήποτε στον κόσμο, να υποβάλει αίτηση για ανθρωπιστική θεώρηση για να ζητήσει προστασία στις χώρες της Ένωσης, στη χώρα της Ένωσης της επιλογής του, αν κατάλαβα καλά τα έγγραφα που μου στείλατε. Δεν έχω στατιστικά για το πόσα άτομα θεωρούν ότι έχουν ανάγκη αυτή την προστασία στον κόσμο. Αλλά υποθέτω ότι οι ενδεχόμενοι υποψήφοι είναι πάρα πολλοί. Η πρόταση προβλέπει επίσης να υπάρξει ευρεία δημοσιότητα για αυτή τη διαδικασία. Αυτή η διαδικασία ωστόσο δεν έχει στόχο να εφαρμοστεί για όσους επιδιώκουν να ε, εισέλθουν παρανόμως στην Ένωση. Αναφέρθηκε ότι 90% των ατόμων που λαμβάνουν άσυλο φτάνουν στην Ένωση, στις χώρες της Ένωσης, παρανόμως. Ωραία. Ένα άλλο στοιχείο που ενδιαφέρει είναι τι ποσοστό μεταξύ όλων εκείνων που εισέρχονται παρανόμως λαμβάνουν τελικά άσυλο. Αυτό είναι ένα στοιχείο που πολύ θα το ήθελα, γιατί δεν το έχω. Γιατί μεταξύ αυτών υπάρχουν οι λεγόμενοι οικονομικοί μετανάστες που δεν υφίστανται διώξεις, αλλά που θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη για να βρουν μια ζωή που την ε, θεωρούν καλύτερη, που τη φαντάζονται καλύτερη. Τα άτομα που δεν θα λάβουν ανθρωπιστική θεώρηση, δεν θα έμπαιναν στον πειρασμό να έρθουν παρόλα αυτά στην Ευρώπη με κάθε τρόπο. Πεδίο εφαρμογή αυτή τη πρωτοβουλία λοιπόν. Είναι ταυτόχρονα και πολύ ευρύ, αλλά ε, όχι κατάλληλο για να αποφύγουμε την τραγωδία της παράνομης μετανάστευσης. Δεύτερη ερώτηση πώς θα αντιμετωπίσουν τα προξενία τα αιτήματα για μια ε, θεώρηση που δεν μπορούν να την αξιολογήσουν και που θα είναι πολλά. Τώρα θα σας μιλήσω ως ε, πρώην πρόξενος. Εργαζόμενος δηλαδή σε αυτό το τομέα. Πρώτη παρατήρηση. Η πρωτοβουλία και αυτή η φιλοδοξία ε, να αφορά όλες τις χώρες και να γίνει ευρύτατα άγνωστη θα έχει ως αίτημα ε, την υποβολή πολλών αιτήσεων αγνώστου αριθμού αιτήσεων αλλά περισσότερων άρα τα προξενία θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν περισσότερες αιτήσει. άρα θα χρειάζονταν περισσότερο προσωπικό μεγαλύτερα περισσότερα γραφεία πιο πολύ ασφάλεια και η χρήση ε, εξωτερικών παρόχων θα ήταν δυνατή. Εδώ βλέπω διαφορετική προσέγγιση μεταξύ του κειμένου που μου έστειλε ο εισηγητής για τον ε, κώδικα για τις θεωρήσεις που αρνείται κάθε χρήση εξωτερικών παρόχων με το σχέδιο εκθέσεως του Κοινοβουλίου που προβλέπει αυτήν την χρήση εξωτερικών ε, παρόχων. Και ποιος θα πληρώσει. Αυτό που κάνει την αίτηση. Δύσκολο μου φαίνεται. Τα κράτη-μέλη. Πότε αυτό μου φαίνεται πολύ πιθανό. Η πρωτοβουλία προβλέπει ότι το κόστος θα αντισταθμιστεί από μια πιο ε, συντεταγμένη άφηξη των ατόμων που χρειάζονται διεθνή προστασία. Αλλά θα ήταν και περισσότερα αυτά τα άτομα. Οπότε φοβάμαι ότι οι αφήξεις ε, των ατόμων που δεν θα έχουν λάβει βίζα ή που δεν θα επιδιώξουν καν να πάρουν αυτή την ανθρωπιστική βίζα θα ήταν ε, όσο άτακτη είναι και τώρα. Και η διαδικασία θα ήταν περίπλοκη. Υποχρεωτική συνέντευξη. Στο προξενείο. Μα αν είναι κάποιο που φοβάται ότι θα διωχθεί αν φανεί στο προξενείο. Πώ θα μπει στο προξενείο. Έχει αστυνομία μπροστά το προξενείο. Θα τον αφήσουν. κατόπιν. Πρέπει να γίνει ε, εξακρίβωση της αυθεντικότητας των αγράφων. Πώς θα γίνει αυτό αν δεν ε, έρθουμε σε επαφή με τις τοπικές αρχές. Και ε, αξιολόγηση του πραγματικού κινδύνου διώξεων. Και επίσης πρέπει να δοθεί απάντηση σε 15 ημερολογιακές μέρες μετά την υποβολή της αίτησης. Μα δεν είναι ρεαλιστικά τα Και αν δεν λάβει θετική απάντηση. Επίση τι θα κάνουμε αν δεν έχει ε, διαβατήριο. Θα του δώσουμε εμεί ένα ταξιδιωτικό έγγραφο. Και αυτό το ταξιδιωτικό έγγραφο θα γίνει δεκτό από τη χώρα διαμονής του. Πώς θα φύγει από αυτή τη χώρα. Θα πάει κάποιο από το προξενείο μαζί του στο αεροδρόμιο. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και αν το άτομο αυτό φτάσει τελικά στη χώρα που του έδωσε την ε, θεώρηση. Τι διαδικασία θα ακολουθηθεί εάν η προστασία που απαιτεί τελικά δεν του αναγνωριστεί. Τι θα κάνουμε. Τώρα, αν το αρνηθούμε αυτή την ανθρωπιστική θεώρηση, η διαδικασία θα ήταν πολύ επιβαρυντική για τα προξενία. Θα πρέπει να είναι ατομική, αιτιολογημένη και γραπτή. Ναι, αλλά θέλει χρόνο κανείς για να τα κάνει αυτά. Άρα και προσωπικό. Και προβλέπεται και προσφυγή. Σε όσους δεν τη λάβουν. Σε όσους την αρνηθούμε. Δεν ξέρουμε. Ούτε πόσοι θα υποβάλουν έτοιμα και ούτε σε πόσους θα την αρνηθούμε. Ίσως στα χίλια άτομα που θα υποβάλουν αυτή την αίτηση, μπορεί μόνο 10 ή 50 να πληρούν τι προποθέσει για αυτή την ανθρωπιστική θεώρηση. Και όλοι οι άλλοι μετά θα κάνουν προσφυγή. Δεν ελέγχουμε καθόλου την κατάσταση. Αντίθετα από ό,τι συχνά θεωρείται, η άρνηση θεώρησης θέλει πολύ, χρόνο, πολύ περισσότερο χρόνο από όσο παίρνει η χορήγηση μιας θεώρησης. Λοιπόν, για να ολοκληρώσω. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που νομίζω ότι έχει πολύ καλές προθέσεις. Δεν έχω καμία νομιμοποίηση εγώ ίδιος για να εκφραστώ υπέρ ή κατά μιας ανθρωπιστικής θεώρησης. Αυτό είναι πολιτικό θέμα. Είναι λοιπόν μια πρωτοβουλία που θέτει πολλά πρακτικά ζητήματα και που θα χρειαζόταν πολύ περισσότερα μέσα και για τα προξενία και για τις αρχές που θα αντιμετωπίσουν μετά τις προσφυγές. Και με βάση την εμπειρία μου, απέχουμε πολύ από το να έχουμε αυτές τις δυνατότητες. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Περνάμε στον τελευταίο μας καλεσμένο, τον εκπρόσωπο της κοινότητας Σαντ Εγκίδιο, τον κύριο Φαν Βόλτερ. Για Γιάντε Βόλτερ, συγγνώμη. Καλώς ήρθατε και πάλι στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Ισηγητά. Δεν είναι όντως η πρώτη φορά που έρχομαι στην Επιτροπή σας. Λυπάμαι, δεν είμαι νομομαθής, οπότε η δική μου παρουσίαση θα είναι μια μαρτυρία ουσιαστικά τι σημαίνει ε, να χρησιμοποιούμε τις, ανθρωπ, τις ανθρωπιστικές θεωρίες για όσους χρήζουν προστασίας, διεθνούς προστασίας, αλλά και για τις χώρες υποδοχής τι σημαίνει κάτι τέτοιο. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Συζητούμε αυτή την πρόταση εδώ και πολύ καιρό. Θα θυμάστε, κύριε Ισηγητά, ότι εκφράστε την ενόχλησή σας για το πόσο χρονοβόρα είναι αυτή η διαδικασία. Ε, θα ήθελα και εγώ να επιχειρήσω αυτή την απογοήτευση και τον εκνευρισμό ε, τόσο συνανθρώπων που περιμένουν μια κίνηση από τη διεθνή κοινότητα και κυρίω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άνθρωποι που προσπαθούν να γλιτώσουν από τον πόλεμο στη Συρία, στη Λιβύη και σε άλλα μέρη του κόσμου και δεν βλέπουν καμία χειρονομία, καμία ένδειξη προ αυτή την κατεύθυνση από τη διεθνή κοινότητα. Και σα ευχαριστώ θερμά για την προσήλωσή σα και τη συνέχιση των προσπαθειών σα προκειμένου να ευοδοθεί αυτή η πρόταση. Τι έχουν βιώσει αυτοί οι άνθρωποι, τι έχουν δει. Έχουν δει μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, όχι μόνο για πιο κλειστή ένωση, αλλά και για όλο και πιο κλειστά σύνορα. Αυτό είδαμε στη Μεσόγειο. Και ε, αυτή η κατάσταση είναι πολύ προβληματική και για τις ίδιες τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικά πρόσφατα, τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες, λόγω των πολιτικών αλλαγών στην Ιταλία, την Αυστρία, τη Γερμανία, αλλά και άλλου στην Ευρώπη, έχουμε διαπιστώσει ότι τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνονται όλο και πιο κλειστά και έχουν σκληρύνει, ειδικά στη Μεσόγειο. Και τα σκάφη διάσωσης μη κυβερνητικών οργανώσεων έχουν προσκρούσει ή άρνηση πρόσβασης στους ευρωπαϊκούς λιμένες, ενώ σε διάσωση ανατίθεται όλο και περισσότερο στην Λιβική ακτοφυλακή. Ένα αποτέλεσμα ήταν τεράστια αύξηση των πνιγμών στην Μεσόγειο, που έχει γίνει ένα υγρό νεκροταφείο. Και με βάση τα στοιχεία της Διεθνούς Οργάνωσης Μετανάστευσης, φέτος πάνω από χίλια άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, έχουν πνιγεί στη Μεσόγειο. Και μάλιστα είχαμε αύξηση το αριθμό των θανάτων τις τελευταίες μέρες. Είναι περίπλοκη η κατάσταση και όντως ομολογούμε ότι είναι πολύ σύνθετη και πολύ διάστατη. Ακούσαμε μια πολύ ωραία πρόταση, όλα καλά και ρόδινα, αλλά ακούσαμε και πολύ ε, επικριτικά σχόλια. Κάτι που δείχνει ίσως μεγαλύτερο ρεαλισμό. Όντως, η κατάσταση είναι περίπλοκη, δεδομένου των εγκληματικών κυκλωμάτων διακίνησης, ε, του τεράστιου αριθμού ε, των πιθανών δικαιούχων για τέτοιες ανθρωπιστικές θεωρήσεις, δεδομένου του μείγματος των οικονομικών μεταναστών και προσφύγων, αλλά και της κόπωσης ε, της ε, κοινή γνώμη της χώρας μας. Όλα αυτά συνιστούν μια πολύ πλοκή κατάσταση. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη έχουν ένα ιστορικό και τρομακτικό καθήκον να δημιουργήσουν μια βιώσιμη πολιτική, χωρί όμω να χάνουν ταυτόχρονα την αλληλεγγύη και τον ανθρωπισμό του, χωρί ειδικά να, να αποποιούνται ε, θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό εδώ μας καλείται ως προσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων που αναζητούν βιώσιμες λύσεις. Αυτό το σκοπό έχει η κοινότητα Σαντατζίντιο που και στη Ρώμη και άλλου στην Ευρώπη αντιμετωπίζει το θέμα της ανθρωπιστικής κρίσης γιατί πολλοί εθελοντές μας δραστηριοποιούνται και υποδέχονται στις ακτές της Λαπεντούζα, της Σικελίας και αλλού ε, μετανάστες και είμαστε υπέρμαχοι της ε, ένταξης, κοινωνικής ένταξης των ε, ε, νεοαφιχθέντων σε πολλές ευρωπαϊκές ε, πόλεις. Γιατί είναι πραγματικά παράλογο. Άνθρωποι που έχουν γλιτώσει από πολέμους χρειάζεται να διακινδυνεύσουν τη ζωή τους, να την παίξουν κορώνα γράμματα και να ξεπουλήσουν τα τελευταία τους υπάρχοντα για να πληρώσουν ύποπτους λαθροδιακινητές για να εισέλθουν στην Ευρώπη και να ζητήσουν άσυλο. Έτσι προέκυψε και η ιδέα των ανθρωπιστικών διαδρόμων. Και όπω όλε οι καλέ ιδέε είναι απλή. Μια μέρα πριν από λίγο, λίγα χρόνια, ο 12 χρονο μου που έβλεπε τα φορτωμένα με μετανάστες πλοία να φτάνουν στι ακτέ, με ρώτησε γιατί δεν πληρώνουμε, δεν αυλώνουμε αεροπλάνα για να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι. Και αυτό το σκοπό έχουν οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι. Εντοπίζουμε στις χώρες προέλευσης ή διέλευσης τους πιο ευάλωτους πρόσφυγες που είναι ε, επιλέξιμοι για διεθνή προστασία, έχουν δηλαδή μεγάλη βεβαιότητα ότι θα λάβουν την διεθνή προστασία από τη στιγμή που θα φτάσουν, θα πατήσουν το πόδι τους στην Ευρώπη, σε χώρε όπω το ο Λίβανο, η Τουρκία, η Αιθιοπία, τους προσφέρουμε ανθρωπιστική θεώρηση και ένα αεροπορικό εισιτήριο για την Ευρώπη και με το μοντέλο αυτό και φυσικά με βασικό γνώμονα την ασφάλεια, την ασφάλεια και για τους ευάλωτους πρόσφυγες, γιατί δεν χρειάζεται πια να παραμείνουν σε πολύ δύσκολε συνθήκε ή να, κινδυνεύσουν, τη ζωή του, τη ζωή των οικείων του ή να γίνουν έρμεα στα χέρια λαθροδιακινητών. Αλλά μα ενδιαφέρει ταυτόχρονα η ασφάλεια και των χωρών υποδοχή. Γιατί οι κρατικέ αρχέ ε, διενεργούν έναν έλεγχο ασφάλειας και γνωρίζουν εκ των προτέρων ποιος εισέρχεται στη χώρα τους. Αυτό λοιπόν το μοντέλο θα καθησυχάσει και το ανήσυχο και αγχωμένο κοινό, την κοινή γνώμη. Η ανθρωπιστική διάδρομη είναι παράδειγμα ασφαλών και νόμιμων διάβλων. Έχουν πραγματοποιηθεί με το μοντέλο της κοινότητας Εντεγίδιο στην Ιταλία, Γαλλία, Βέλγιο και βοήθησαν πάνω από 3.000 πρόσφυγες, κυρίως Σύρους που διαμένουν στο Λίβανο ή Ερυθρέους που διαμένουν στην Αιθιοπία. Και μάλιστα όλος παραδόξως, ε, και αυτό είναι στοιχείο πολιτικού ε, ρεαλισμού. Η κοινότητα Σεντετζίδιο προκάλεσε το ενδιαφέρον και αριστερών και δεξιών παρατάξεων. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, η συμφωνία υπογράφηκε στο Προεδρικό Μέγαρο από τον, πρόεδρο, τον τότε πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ. Αλλά και ο νυν πρόεδρο ε, τη Γαλλία, ο Μανουέλ Μακρόν, είναι έτοιμο να συνεχίσει την προσπάθεια αυτή και μάλιστα να, την ενισχύσει. Ακόμη και μερικά κρατήδια όπω το Σαν Μαρίνο και η Ανδώρα έχουν υιοθετήσει το μοντέλο αυτό για κάποιες οικογένειες και μάλιστα ευελπιστούμε ότι θα επεκτείνουμε αυτό το σχέδιο και σε άλλες χώρες και κοινοτικέ και τρίτες χώρες. Υπάρχει και ένα δεύτερο στοιχείο των ανθρωπιστικών διαδρόμων που καθιστούν αυτό το σχέδιο και καινοτόμο αλλά και ελκυστικό για τις κυβερνήσεις. Η χρηματοδότηση του σχεδίου αυτού είναι ιδιωτική γιατί φαντάζομαι σε ενδιαφέρει το κόστος και ποιος θα το αναλάβει. Η κοινότητα Σαντετζίδη, από τους εταίρους της, που είναι κυρίως καθολικοί επίσκοποι, ε, πρωτοστατικές εκκλησίες στην Ευρώπη, στο Βέλγιο όμως και μουσουλμανικές και εβραϊκές κοινότητες. Αυτές καταβάλουν τα ε, ναύλα των αεροπορικών εισιτηρίων, τα διοικητικά τέλη για τις ε, θεωρήσεις, αλλά και παρέχουν τις στέγη της οικογένειας Και επίσης παρακολουθούν την κοινωνική τους ένταξη. Και μάλιστα αυτή η στήριξη σε ενορίες και κοινότητε ε, στην επικράτεια αυτή έχει κέριο ρόλο για την επιτυχία του προβλήματος ε, για την επιτυχία συγγνώμη, του σχεδίου αυτού. Επίση, έχει αποδειχθεί και αναγνωριστεί και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι τέτοιου είδου ιδιωτικέ χορηγίε διευρύνουν τι ε, ευκαιρίε κοινωνική ένταξη, επιτυχού κοινωνικού ένταξη των ερχομένων, χωρί να φοβίζουν το κοινό. Γι' αυτό προωθούμε τέτοιε μορφέ έμπρακτη αλληλεγγύη που λαμβάνουν υπόψη τη συνεργασία δημόσιο και ιδιωτικού τομέα και δεν επιρρύπτουν όλο το βάρο χρηματοδότηση στο κράτο και ταυτόχρονα μειώνουν τον αριθμό των πιθανών θυμάτων των λαθροδιακινητών ή των σωματεμπόρων. Σε ό,τι αφορά τι τεχνικέ πτυχέ τη ανθρωπιστική θεώρηση, που είναι το βασικό στοιχείο τη συζήτηση, και λυπάμαι γιατί έλαβα πολύ αργά σήμερα το κείμενο, οπότε δεν, δεν πρόλαβα να μελετήσω εδελεχώ στην πρόταση. Πάντω, χρησιμοποιούμε ω νομική βάση αυτή η πιθανότητα που προσφέρει ο κώδικας θεωρήσεων στις κυβερνήσεις να εκδώσουν θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους και μόνο σε μερικές περιπτώσεις χρησιμοποιούμε το άρθρο 25 του, Α, του κώδικα που επιτρέπει στα κράτη-μέλη να εκδώσουν ε, θεωρήσεις με περιορισμένη εδαφική ισχύ για ανθρωπιστικούς λόγους και πάλι. Βέβαια αυτή η διαδικασία δεν είναι συνήθις και έχει ένα μεγάλο βαθμό έκτακτο χαρακτήρα, εξαιρετικού χαρακτήρα. Και μάλιστα η κοινότητά μας είναι ευγνώμων προς τις κυβερνήσεις αυτές που έδειξαν προθυμία και συνεργασία ε, για να δημιουργήσουν τέτοιους ανθρωπιστικούς διαδρόμους και δεδομένων των θετικών αποτελεσμάτων της καλής κοινωνικής ένταξης των προσφύγων και τη χρήση, της χρήσης δικτύων αλληλεγγύης που υπάρχουν στις ευρωπαϊκές κοινωνίες θεωρούμε ότι ένα σχέδιο θα όφιλε και θα έπρεπε να επεκτεθεί σε μεγαλύτερο ρυθμό προσφύγων και σε περισσότερες χώρες μέλη ό,τι αφορά τη διαδικασία για τη λήψη θεώρησης. Αυτό που είδαμε και ακούσαμε για την πρόταση νομίζω ότι είναι πανέμορφο και διαρωτώ με αν είναι και πολιτικά εφικτό, γιατί στη θεωρία είναι πολύ ελκυστικό δεδομένη της ε, ε, απροθυμίας κάποιων χωρών στο Συμβούλιο και της παρακολουτική διαδικασίας κολλησιεργίας που χρησιμοποιούν. Τώρα, σε ό,τι αφορά το νομικό πλαίσιο, καταρχήν ε, θέλουμε η άδεια για την ε, είσοδο για ανθρωπιστικού λόγου, να μην έχει έκτακτο εξαιρετικό μόνο χαρακτήρα, αλλά να γίνει πιο γενική, πιο τακτική και να προβλέπεται σε συγκεκριμένους ε, ε, σε συγκεκριμένα άτομα ή σε επιστοποιημένους οργανισμούς να αναλάβουν τη χορηγία αυτών των ατόμων που είναι επιλέξιμοι για ανθρωπιστική προστασία. Κύριε Ντεβόλτερ, παρακαλώ ολοκληρώστε γιατί έχουμε ε, πρέπει να προβλέψουμε κάποιο χρόνο και για τη συζήτηση. Ναι, δώστε μου ένα λεπτό ακόμη. Και επίσης, ευάλωτοι άνθρωποι με χορηγούς που εξασφαλίζουν την επαρκή υποδοχή τους, την κατάλληλη υποδοχή τους, θα πρέπει να επιτρέπεται σε, στα πλαίσια της προστατευμένης εισόδου. Εν κατακλείδη, αν βοηθά και πιστεύουμε ότι μπορεί να βοηθήσει μία εναρμόνιση σε κάποιο βαθμό και μια ε, διάδοση αυτής της εμπειρίας, γενίκευσή της προς τις ανθρωπιστικές θεωρίες και τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους θα ήταν ευχής έργων. Αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να είμαστε και ρεαλιστές και να μην αποδυναμώσουμε με μια τέτοια πρόταση τη δυνατότητα των κρατών μελών να εισέλθουν σε ένα τέτοιο σχέδιο. Σας ευχαριστώ και λυπάμαι που μακρηγόρησα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φτάνουμε στο τέλος ε, της προγραμματισμένης, ε, του προγραμματισμένου ωραρίου της ε, ακροασής μας. Δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε υπέρβαση ωραρίου. Αν χρειαστεί θα συνεχίσουμε στα αγγλικά. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων τους διερμηνείς, οι οποίοι ανακοίνωσαν ότι στις 6 και μισή να σταματήσουν την διερμηνία. Πρέπει να υπάρχει χρόνος για τους ευρωβουλευτές να θέσουν τα ερωτήματά τους. Κυρία Σπινέλη, αν θέλετε να πάρει το λόγο, οποιοδήποτε άλλος θέλει να πάρει το λόγο, ευχαρίστως ε, να τον ακούσουμε. Πάρα πολύ σύντομα. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Τεφόιτερ για την ε, εμπειρία του και τη μαρτυρία του ε, για τους, ε, από τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους και θα ήθελα να πω και κάτι σε σχέση με το κόστος των επιχειρήσεων για τις οποίες μίλησε ο δόκτωρ Τεγέγκερ. Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο είναι απαραίτητο ή δυνατό να κάνουμε μία αξιολόγηση του κόστους του ανοίγματο των πολιτικών, ε, της πολιτικής θεωρήσεων σε σχέση με το κόστος του μη ανοίγματο των ανθρωπιστικών διαδρόμων και της ύπαρξης ε, νομίμων ε, διαδρόμων. Νομίζω ότι το κόστος της μη ύπαρξης πολιτικής ασύλου είναι πολύ ψηλότερο από το κόστος του να μην μπορούμε να ε, τηρήσουμε το ε, πρωτογενές και παράγωγο δίκαιο, όπως εξήγησε και η κυρία ε, Μορένο. Μορένο Λάξ, γιατί είναι απλώς απλούστερο να έχουμε νόμιμες, ε, νόμιμου, νόμιμες οδούς. Και βλέπω ότι δεν υπάρχει μακροχρόνια προσέγγιση, μόνο βραχυπρόθεσμη προσέγγιση υπάρχει από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δημογραφικά, η δημογραφική τάση δεν είναι καλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τη μετανάστευση, χρειαζόμαστε ανθρωπιστικούς διαδρόμους και νόμιμες ε, διόδους, όπως και την αναθεώρηση του συστήματος του Δουβλίνου, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνονται σεβαστές και κυρίως ε, η αλληλεγγύη. Ο κύριος Μπέκερ. Πολύ σύντομα. Ευχαριστώ πολύ για τις καταπληκτικές και τόσο πλήρης ε, παρουσίασης ενός φάσματος ε, θεμάτων που έχουν να κάνουν με αυτό νομοθετικά, κόστος δύο παρατηρήσεις σας παρακαλώ μην με παρεξηγήσετε αλλά είναι τμήμα της ανάλυσης που πρέπει να κάνω κυρίως ως πολιτικός όχι ως νομομαθής υπάρχει η στρατηγική του Συμβουλίου που είναι υπό συζήτηση που θέλει να παρεμποδίσει τη δράση των διακινητών. Θέλει να δημιουργηθούν κέντρα υποδοχής εκτός της Ένωσης. Εκτός της επικράτειας της Ένωσης. Ακριβώς εκεί από όπου γίνεται τώρα η διακίνηση. Το ότι κάποια κράτη της Αφρικής το απέρριψαν δεν με ανησυχεί. Όλα αυτά είναι διαπραγματευτική τακτική. Αυτό σημαίνει ότι το αίτημα για υποβολή ε, ασύλου θα γίνεται πριν μπει κανείς στην Ένωση. Αυτό με ενδιαφέρει. Γιατί όλα τα άλλα γίνονται όσο πιο δύσκολα. Όσο περισσότερο σας ακούω. Αλλά δεν αποφεύγουμε τις ευθύνες μας. Όχι. Είναι μια διευκρίνηση ότι προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα μοντέλο. Θα δούμε σε τι βαθμό μπορεί να υλοποιηθεί. Το δεύτερο. Αναφέρομαι σε αυτά που είπε ο κύριος Ντεζεγέρ. Ανέφερε σημεία όπου ανοιχτά πρέπει να πω αυτά τα σημεία πρέπει οπωσδήποτε να τα λάβουμε υπόψη στα νομοθετήματα που θα προτείνουμε. Πρέπει να δώσουμε απαντήσεις. Πότε, ποιος, πόσοι, ποιες δυσχέρειες πρέπει να λύσουμε, όλα αυτά που απαριθμίσατε. Και Λυπάμαι που δεν έχετε κάποιο PowerPoint να περιλαμβάνει αυτά που μας παρουσιάσατε. Κατά τα άλλα, δεν νομίζω ότι αλλάζει τίποτα. Στη σωστή άποψη να επιτύχουμε αυτό το στόχο, ούτως ώστε να υπάρξει κάποια τάξη σε αυτό το σύστημα. Γιατί οι ετούντες άσυλο, όσοι χρειάζονται προστασία, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με αυτά που λέει η συμφωνία, ε, η σύμβαση της Γενέβης και όπως είπατε και εσείς ήταν ε, σαφέστατα αυτά που μας είπατε και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Βαλέρο και η Έλλη Σλάιν. Κυρία Βαλέρο. Ευχαριστώ πολύ. Είχα το ίδιο ερώτημα με την Μπάρμπαρα Σπινέλη. Ναι, κοστίζει πολύ. να υπάρξει μια τέτοιου είδου ανθρωπιστική θεώρηση ε, και γι' αυτό πολλέ χώρε ε, δεν την επιθυμούν. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που έχουμε πάντοτε να αντιμετωπίσουμε, ότι είναι πολύ μεγάλο φόρτος εργασία για τα προξενία, για τι πρεσβείε. Αυτό όμω έχει να κάνει με αυτό που είπε ο κύριο Μπέκερ για τα κέντρα αυτά, τα οποία θα βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λογικά εκεί πρέπει να γίνεται η εξέταση της αίτηση ασύλου πριν φτάσει το πρόσωπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα είναι δαπανηρό και αυτό. Πώς θα υπάρξει μία ε, νόμιμη ασφαλής εξέταση της αίτησής, ε, της αίτησής σου ε, σε τέτοιου είδους κέντρα. Πολλές φορές, πολλοί κόσμος δεν κάνει αίτηση γιατί είναι πολύ δαπανηρό. Πρέπει να βρούμε μία λύση νόμιμων διόδων προς την Ευρώπη εντάξει, κοστίζει πολύ να το κάνουμε με εξωτερική ανάμαθεση. Με όποιο τρόπο για να το κάνει κανείς, κοστίζει πολύ. Νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος είναι να ανοίξουν νόμιμες ε, δύο μετανάστευσης για ανθρωπιστικούς λόγους. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πολύ γρήγορα. Και μετά μπορεί στα αγγλικά να συνεχίσουμε για τις απαντήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αφού οι διερμηνείς είναι ακόμη εδώ, θα μιλήσω Ιταλικά. Συμφωνώ και με τους λόγους για τους οποίους απεργούν, να το πω και αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους προκεκλημένους γιατί ε, μας εξήγησαν πολύ καλά το τι μπορεί να κάνουν ε, τα ευρωπαϊκά όργανα αλλά και οι εθνικές αρχές για ένα τόσο περίπλοκο και δύσκολο ζήτημα. Το είπα, ο καλύτερος, ο πιο σωστός τρόπος να αντιμετωπίσουμε την παράνομη μετανάστευση είναι να αποφύγουμε τι ανθρώπινες τραγωδίες στη Μεσόγειο, δηλαδή να δημιουργήσουμε ασφαλείς εναλλακτικέ διόδου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί κανείς να ζητήσει άσυλο γιατί διαφορετικά μόνο πτώματα θα μαζεύουμε στι ακτέ μα. Ε, ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που μας τα είπατε όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για το κοινοβούλιο μας να συνεχίσει τον αγώνα αυτό. Να ευχαριστήσω τον Χουάν Φερνάντο. Πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους, ε, τις νόμιμες οδούς μετανάστευσης και τη σωστή υποδοχή των ανθρώπων αυτών και να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Δυστυχώ που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πριν από δύο εβδομάδες έχασε αυτήν την ιστορική ευκαιρία να προχωρήσει παραπάνω την ε, ε, αναδιάρθρωση του ε, Δουβλίνου, δυστυχώς ούτε αναφέρονται αυτές οι νόμοι μεσοδοί μετανάστευση, γιατί υπάρχει αυτή η αιμονή με την ασφάλεια στο Συμβούλιο. Όταν μιλάει για αυτά τα κέντρα αποβίβασης, πλατφόρμες αποβίβασης, μία νέα απεικιοκρατική προσέγγιση είναι αυτή. πρέπει να ακολουθήσουμε το καλό παράδειγμα που έχει αρχίσει να υπάρχει ε, σε πολλές χώρες. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ε, γι' αυτό ακριβώς ε, συζητούμε για την αλληλεγγύη. Πολλές φορές δεν υπάρχει αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εμείς θα θέλαμε να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας προς τους διερμηνείς για τη δουλειά που κάνουν και για τον αγώνα τους. Τους υποστηρίξουμε. ένας γρήγορος γύρος ε, απαντήσεων. Ε, ποιος θέλει να πάρει το λόγο αν θεωρεί ότι του ετέθη κάποιο ερώτημα με τη σειρά που μιλήσατε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να απαντήσουμε ε, στα θέματα που τίθονται κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων με τη σειρά που ετέθησαν. Ε, θα ήθελα να πω προς τον κύριο Ντεγέγκερ και τον κύριο Ντεβόλιν, διαβάστε τις εκθέσεις μας ε, και να δείτε τις διάφορες ανησυχίες που ε, υπάρχουν και που καλύφθηκαν. Η ανησυχία του κυρίου Ντεβόλιν που προφανώς αναφέρεται στην έκθεση και θα ήθελα να πω επίσης σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Πέκε. Προσπαθούμε και αυτά να τα λάβουμε υπόψη. Ε, θα είναι πάρα πολύ καλό για την ε, ε, συνέχιση των εργασιών στην Επιτροπή σας. Κυρία Φερνάντες. Ναι, θα ήθελα να, σχολήσω για, να, να σχολιάσω το κόστος των ε, πολιτικών ε, που ανέφεραν πολλοί. Αναφέρονται τα ωφέλη, έχουν άμεση σχέση με το πώς ε, εφαρμόζεται η κάθε επιλογή πολιτικής, όπως επίσης και τα αποτέλεσμα εξαρτάται από αυτό. Ε, είδαμε διάφορα τους του ε, ε, που αναφέρθηκαν οι ανθρώπινη πόροι για παράδειγμα η αξιολόγηση της επεξεργασίας των αιτήσεων για χορήγηση θεώρησης και τη δουλειά των προξενείων των κρατών μελών προσπαθούμε όλο αυτό το ρεαλισμό να το συμπεριλάβουμε στην ανάλυση μας Επίσης βλέπουμε τι γίνεται και με την ε, επανεκατάσταση. η αρμοστία έχει ένα εγχειρίδιο σε σχέση με το θέμα αυτό, την επανεκατάσταση και από αυτό μπορούμε να μάθουμε, όπως επίσης και από τις τρέχουσες εμπειρίες με τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους. Ευχαριστώ. Κύριε Λάξ. I wanted to, to reply that this is actually a legal question.